As you know, colleagues, we have a very long afternoon today. Επειδή είναι αρκετά φορτωμένη η ημερήσια διάθεση του σημερινού απογεύματος, θα σας παρακαλέσω να καθίσετε σύντομα για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. For EPP, this... Πρόκειται για την χρυσή στιγμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. γιατί όπου και να στρέψω τα βλέμματα βλέπω συναδέλφους του ΕΛΚ. I am counting how many members. Μετρώ, μετρώ ε, τα μέλη που είναι παρόντα, γιατί χρειαζόμαστε 12 για να έχουμε την απαρτία. Νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στην απαρτία. Έτσι είναι, είμαστε ήδη 12. Ωραία λοιπόν, συνεχίζει η πρόεδρος κυρία Βίκστρομ. Ελπίζω να μπορέσατε να ε, απολαύσετε το μεσημεριανό σας γεύμα και ας αρχίσουμε τώρα με την έκβαση πρώτα της ε, συναντήσεως των συντονιστών που αυτή, αυτά θα ήθελα να σας πω τώρα. Πρώτα, εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη του Απριλίου καθώς και ορισμένα αιτήματα για συμπερίληψη σε άλλες. Για την ατζέντα του Απριλίου έχουμε αναπηρίες, ποιότητα ε, του ατμοσφαιρικού αέρα, διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και ε, αθλητική δημοσιογραφία και η προφορική ερώτηση για τη ΦΑΤΚΑ πηγαίνει για τον Μάιο. Οι, δε, οι δύο αιτήσει κατεπήγοντος εγκρίθηκαν επίσης, δηλαδή πυρηνικός σταθμός Τιάντζ και η έδρα του EMA. Ο Πέτερ Γιάρ έχει ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ. Θα θέλαμε να ασκήσουμε κριτική στην απόφαση των συντονιστών για την διαγραφή από την ημερήσια διάταξη της αναφοράς 636-17. Επαναφέρουμε το αίτημα 636-17 για ε, διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα κλπ. Θέλουμε λοιπόν να καταθέσουμε το αίτημα η αναφορά αυτή να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου. Και παρακαλώ την Πρόεδρο να διεξαγάγει ψηφοφορία στο, εδώ στην Επιτροπή Αναφόρων. Αφού λοιπόν έχετε προσβάλει την απόφαση αυτή σύμφωνα με το 205 του κανονισμού, θα την θέσω υπόψη του συνόλου της Επιτροπής αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ατυχές ότι μόνο μέλη του Λαϊκού Κόμματος βρίσκονται και ένα μέλος της EFDD. Δυστυχώς είναι απολύτως ατυχές. Α, υπάρχει και ένα μέλος των φιλελευθέρων. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν δύο μέλη ακόμη. Και ε, εσείς και η Τουργκάης έχετε ζητήσει το λόγο, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, εγώ ήμουν ε, μέλος ε, της Επιτροπής Αναφορών για 10 χρόνια και ε, εσείς γνωρίζετε, όπως και κάποιοι άλλοι, τον ενθουσιατικό κανονισμό της Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή ξεκίνησε τη συνεδρίαση της σήμερα το πρωί, είχε ένα συγκεκριμένο χρόνο έναρξης, 14 και 30. Όσοι, όσοι βουλευτές δεν είναι παρόντες, πρόβλημά τους. Ο συντονιστής μου ζήτησε κάτι, ζήτησε να μπει κάτι σε ψηφοφορία. Είμαστε εδώ και οφείλουμε να είμαστε εδώ την ώρα που ξεκινάει η ημερήσια διάταξη και η συνεδρίαση της Επιτροπής. Ζητώ λοιπόν, όχι απαιτώ, ε, να λάβετε υπόψη σας το αίτημα του συντονιστού του ΕΛΚ και βάσει του κανονισμού, βάσει του νόμου δηλαδή, ε, να ε, υποβάλλετε το ερώτημα του Πίτερ Γιάρ, του συναδέλφου μου, σε ψηφοφορία. Ασφαλώς και θα το πράξω. Ασφαλώς, μην ανησυχείτε, λέει η πρόεδρος κυρία Βίξτρομ. Νομίζω όμως ότι πρώτα θα σας εξηγήσω όλα τα συμπεράσματα των συντονιστών, δηλαδή θα το αναβάλω για λίγο και ελπίζω σιγά σιγά να προσέλθουν και άλλα μέλη της Επιτροπής ώστε να έχουμε μια ευρύτερη εκπροσώπηση. Θα αναβάλω το αίτημα, την ψηφοφορία για δύο λεπτά. Δύο λεπτά θα είναι. Η ημερήσια διάταξη του Μαΐου, μιλώ για τις αναφορές που θα προσθεθούν στην ατζέντα του Μαΐου για την υδατοκαλλιέργεια, για δε την ατζέντα του διακόπτη κάποιος. Η πρόεδρος. Αντιλαμβάνομαι ότι επιθυμείτε να ζητήσετε την πληροφορία αμέσω. Όχι, Ζήτησα επισήμω να ψηφίσουμε. Είπαμε δυόμιση ώρα και είναι η ώρα έναρξης των εργασιών της Επιτροπής. Ο Πέτερ Γιά ζήτησε και πρέπει να ψηφίσετε. Εσείς το βάλατε. Μιλήσατε για το θέμα, πρέπει να ψηφίσουμε αμέσως κυρία μου. Καλά λέει η Πρόεδρος. Ναι, ναι, θα το κάνουμε. Το αίτημα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι να διατηρηθεί 636-17 στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου. Για να δούμε μήπως είσαστε όμως και υπερβάλλοντα τα μέλη σε αριθμό. Εννέα μέλη σας δικαιούνται να ψηφίσουν. Πίτερ, είστε ο συντονιστής. Εννέα λοιπόν θα ψηφίσουν. Έχει καλός. Συνεχίζει η πρόεδρος. Ο Γιάρεκ είναι ελεύθερο σωματίδιο αυτή την ε, φορά. Okay. Ωραία λοιπόν, να βεβαιωθούμε τώρα ότι όσοι θα ψηφίσουν για το Λαϊκό Κόμμα είναι είτε πλήρη, δηλαδή τακτικά, είτε αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Θα δώσω λίγα δευτερόλεπτα στους policy advisor για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα που θα ψηφίσουν είναι τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Ταυτόχρονα θα παρακαλέσω τους άλλους, policy advisors να ειδοποιήσουν τα δικά τους μέλη. Also, dear Chairman, wir sind dann acht. Members Okay. Ε? Any member. Πρόεδρος. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ψηφίσει, αλλά οι policy advisor να μας ανακοινώσουν ποια είναι τα μέλη αυτά. Είτε τακτικά είτε αναπληρωματικά μέλη. Και αν θέλετε να υπάρχουν τα μέλη, να μας γνωρίσετε από πριν ποια είναι αυτά. E η policy advisor του Λαϊκού Κόμματος και της Ευθυντή σωστά τα κάνανε. Το αίτημα λοιπόν του Λαϊκού Κόμματος είναι να διατηρηθεί η αναφορά 636 του 17 στην ατζέντα του Απριλίου. Ποιος είναι υπέρ? Παρακαλώ σηκώστε καλά τα χέρια. Ένδεκα μέλη λοιπόν λέει θέλει να γίνει σεβαστή η απόφαση των συντονιστών να μπει το Μάιο και μάλιστα στη λίστα Β. Τα δύο μέλη της ομάδας EFDD. Καλώς λοιπόν. Λάβαμε απόφαση. Η απόφαση λήφθη. Θα ήταν καλό τα μέλη που ήρθαν ειδικώ για την ψηφοφορία είτε να παραμείνουν καθισμένοι είτε να αποχωρήσουν διακριτικά. Δεν εννοώ τον κύριο Πρέντα ειδικώ. Η μερίσια του Ιουνίου. Α, Ελεονόρα, παρακαλώ εσεί. Συγγνώμη. Να πω απλώ ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι φυσιολογική και θα ήθελα να σημειωθεί γιατί θα μπορούσε να συζητηθεί για περαιτέρω συζήτηση σε επόμενη συνάντηση των συνεδρίων των συντονιστών. Can, Να απαντήσω στην ε, κυρία Εύη. Και εγώ, και εγώ ε, δεν είμαι διόλου ικανοποιημένη από τον τρόπο που χειριστήκαμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά δεν μπορώ να κάνω και τίποτε άλλο. Με φέρατε σε ε, εξαιρετικά δύσκολη θέση και νομίζω ότι το στοιχείο συναδελφικότητας μεταξύ συναδέλφων από διάφορες πολιτικές ομάδες θα πρέπει να βελτιωθεί. Δεν είναι αξιοπρεπής ε, τρόπος συνεργασίας αυτός μέσα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι απολύτως ανώριμη η στάση αυτή και αγενής. Όσοι μας παρακολουθούν σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το σώμα θα ήθελε να λειτουργεί πολύ διαφορετικά και αυτό ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο ε, συζήτησαν οι συντονιστές σήμερα το πρωί αλλά και για το πώς έγινε η ψηφοφορία τώρα μόλις. Ε, λυπούμε πολύ λοιπόν. Φέρετε τη λύπη μου γι' αυτό. Η κυρία Τουργκάης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Τουργκάης. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι το ζήτημα και το πρόβλημα δεν αφορά ε, αυτούς που έρχονται να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά αυτούς που δεν έρχονται επαναλαμβάνω, στις 2 και μισή για όλους τους συναδέλφους ε, ε, ήταν ε, η ώρα εκκίνησης της συνεδρίασης. Ρωτήστε λοιπόν τους άλλους από τις άλλες πολιτικές ομάδες γιατί δεν ήταν εδώ στις δύο και μισή. Αυτό που λέω εγώ, λέει η Πρόεδρος, είναι ότι συμφωνώ με την κυρία Εύη ότι αυτό το θέμα θα ξαναπροκύψει στις επόμενους συντονιστές και τους μεθεπόμενους κλπ. Μπορούμε να προβλέψουμε λοιπόν μια μακρά χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να χειριστούμε το θέμα αυτό. Εάν θέλετε να το κάνουμε σωστά και απολύτως σύμφωνα με τους ε, διαδικαστικούς ε, κανόνες, θα το έχουμε μπροστά μας για πολύ καιρό ακόμα. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε αυτά που έλεγα. Τι άλλα έκαναν οι συντονιστές το πρωί. Ελευθερία έκφρασης ε, στην Μάλτα και δημοσιογράφη στην Μάλτα. Ε, επίσης ε, παραβίαση ε, του κανονισμού 338 και τα, στη Βουλγαρία τα δικαιώματα των καταναλωτών θα μπουν σε σε διάταξη. Όσον αφορά γνωμοδοτήσεις, εγώ θα είμαι ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, υπεύθυνη για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Επίσης η Άλτε θα ετοιμάσει την ειδική έκθεση για τον ε, συνήγορο του πολίτη. Οι πράσινοι θα κάνουν την έκθεση για την αναθεώρηση του καταστατικού για τον ε, Ombudsman και δεν θα συζητήσουμε το θέμα των μειονοτήτων για την Ευρω... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης όσον αφορά τις συστάσεις, εκτός από την 10 54 ε, ε, και την 1081, 1111 και 1122. Αυτές θα παραμείνουν ε, όλες εκτός από τη 1054. Επίσης, λεπτομερείς συζητήσεις θα λάβουν χώρα όσον αφορά τα θέματα B και όλες οι αποφάσεις αυτές θα γραφτούν, θα βρεθούν σε γραπτή μορφή. Ε, επίσης αποφασίστηκε να επισκεφθούμε την Βαλεντόρα και την Δονάνια στο δεύτερο μισό ε, του ε, χρόνου και επίσης ε, η Επιτροπή για τις Αναπηρίες ε, θα ε, δώσει τη θέση της σε μια ακρόαση. Όσον αφορά την Επιτροπή ΕΜΠΛ, θα ασχοληθεί και θα εμπλακεί με το θέμα της καταπολέμησης επισφαλούς και προσωρινής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό θα υπάρξει αργότερα έκθεση. Επίσης αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για θέματα τα οποία θα αποφασιστούν με γραπτή διαδικασία. Όσον αφορά τον παλεγιάζ, θα επανέλθουν στο θέμα αυτό ε, την αρχή του επόμενου χρόνου οι συντονιστές. Και επίσης όσον αφορά την διακριτική μεταχείριση ε, στην Σουηδία πολιτών ε, είχε γίνει μια διαρευνητική αποστολή εκεί και αποφασίσαμε ότι θα σταλεί επιστολή ε, που θα υπενθυμίζει όλα τα ζητήματα τα οποία γύραμε στη διάρκεια της συνάντησης στη Σουηδία. Επίσης, οι συντονιστές έλαβαν γνώση των θεμάτων προς πληροφόρηση και αυτά είναι όλα που είχα να σας πω για τους συντονιστές. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 13 η 2191 του Πιέρο Μπρούνι ε, σχετικά με τη ρήπανση της λίμνης Μπολσένα. Είναι παρόν ο κύριος Μπρούνι. Yes, there you are. And I am happy to invite you to take the floor for five minutes. Βάδο. Να ξεκινήσω, λέει ο κύριος Πιέρο Μπρούνι. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά ε, την παρουσία φωσφόρου ε, στην ε, λίμνη Μπολσένα σε μεγάλη πυκνότητα. Μάλιστα, 8 έγιναν 16 μικρογραμμάρια αυτές οι συγκεντρώσεις και αφορούν πλέον το σύνολο της λίμνης και αντιπροσωπεύουν περίπου από 75.000 κιλά μέχρι και το διπλό. Πρόκειται ε, για αύξηση 17 κιλών ε, που ε, οφείλονται στη γεωργία καθώς επίσης και στα αστικά απόβλητα. Όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, Το σχήμα που έχουμε δείχνει ότι ε, αυτά, ε, όλα αυτά τα απόβλητα ε, οδηγούνται σε έναν κεντρικό ταμιευτήρα. Όμως, επειδή ο ταμιευτήρας αυτός είναι απροστάτευτος, στην ουσία καταλήγουν ή στην λίμνη έγινε ε, μία προσπάθεια ε, λύσης του προβλήματος μέσω 20 ε, αντιλιών, σταθμών απάντησης. Ωστόσο, οι σταθμοί που μας απασχολούν περισσότερο είναι οι παριθμών 9 που τη βλέπετε στη διαφάνεια, καθώς επίσης και ο σταθμός 20. Ο σταθμός 20 είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται έξω από την πράσινη περιοχή και συλλέγει στην ουσία όλα τα απόβλητα του, ε, ε, ε της ε, λίμνης που καταλήγουν στην λεκάνη αποστράγγισης και εν τέλει στο διπλανό ποτάμι. Επάνω αριστερά βλέπουμε τον κεντρικό σταθμό Τέμπη που στην ουσία, στην πραγματικότητα δεν είναι όμως ε, ε, ε, ε συνδεδεμένος με τον ταμιευτήρα και βλέπουμε επίσης ε, ότι η ποσότητα του υγρού δεν μπορεί να, είναι, να αφορά 30.000 κατοίκους, είναι πολύ χαμηλότερη και επομένως ε, πολλά υγρά απόβλητα στην ουσία χάνονται στην, στην λίμνη πριν φτάσουν στο σταθμό απάντηλησης 20. Ο δεσταθμός 9 που είχα αναφέρει προηγουμένως βγάζει, χύνει αν θέλετε όλα του τα απόβλητα, υγρά απόβλητα, ε, εις την λίμνη Μπολσένα. Στην πραγματικότητα, στο σύνολο των εγκαταστάσεων, το 75% του φωσφόρου που τελικά καταλήγει στη λίμνη ε, προέρχεται από τα αστικά απόβλητα και μονάχα 25% ε, προέρχεται από τη γεωργική δραστηριότητα. Εδώ πρόκειται βέβαια για χονδροειδείς υπολογισμούς, ωστόσο αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Ε, occorre, prima di tutto πρωτίστως πρέπει να αλλάξει, να διορθωθεί ο κεντρικός ταμιευτήρας και μετά να υποστηριχθεί ε, η ε, ε, γεωργία μέσω κινητροδότησης βιολογικών καλλιεργιών. Επίσης, χρειάζεται να ε, συσταθεί ένα ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο. Όσον αφορά τη βιώσιμη γεωργία, αντί να προωθούνται ε, καλλιέργειες βιώσιμες, ε, προωθήθηκε η φουντουκιά, η οποία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Εδώ βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε και πολύ καλά βέβαια, ε, λέει ο μιλητή, γιατί το σχήμα δεν είναι πολύ καθαρό. Ε, βλέπετε ιστορικά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Το 2009 συνεργαστήκαμε έτσι ώστε να συστήσουμε ένα σχέδιο διαχείρισης της λίμνης Μπολσένας. Αυτό το σχέδιο διαχείρισης ανεφέρεται ότι ε, δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε, δεν θα έπρεπε να υπερβούμε τα 10 μικρογραμμάρια ανά λίτρο και ότι χρειαζόταν μία ε, ε, ενιαία διαχείριση της λίμνης. Εγκρίθηκε το σχέδιο αυτό από την ε, επαρχία, αλλά το αγνόησε η περιφέρεια. Το καλοκαίρι του 2011 ε, ε, συλλέξαμε 14.000 υπογραφές διαμαρτυρίας που κατετέθησαν, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Το 2013 στράφημε προς την Επιτροπή Αναφορών. Υπήρξε μία περίοδος διακοπής λόγω των εκλογών, άλλαξε η Προεδρία και το 2015 επομένως είχαμε την πρώτη μας ακρόαση κατόπιν της οποίας ε, η παρούσα πρόεδρος της Επιτροπής έστειλε μια επιστολή στην περιφέρεια του Λάτσιο ε, ζητώντας ε, την διαθέτηση του προβλήματος του ταμιευτήρα καθώς επίσης και την βελτίωση της βιώσιμης γεωργίας. Λίγο μετά έλαβε χώρα διαγωνισμός και μετά επελέγει ε, η σχετική επιχείρηση. Αλλά ε, ωστόσο μόνο το Σεπτέμβριο ξεκίνησε ε, η εταιρεία να εργάζεται επί του ταμιευτήρα. Κύριε Μπρούνι, πέντε λεπτά είπαμε. Μήπως θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε την παρέμβασή σας και έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την παρουσία του θέματος, παρουσίαση του θέματος. Ναι, Εν πάση περιπτώσει, περιμένοντας και περιμένοντας, ε, ε, έχει ακόμα ε, επιδεινωθεί η κατάσταση της λίμνης Μπολσένα. Πρόεδρος, σας διαβεβαιώ ότι όλοι γνωρίζουμε το θέμα, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε διαβάσει. Δεν θέλω να είμαι αναγωγή, αλλά έχουμε πολύ βεβαρημένη ημερήσια διάταξη και δεν μπορεί η κάθε παρουσίαση να είναι τόσο μακροσκελής. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ και θα σας δώσω και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Γκασπαρινέτη. You need to put on the micro. Ανάψτε το μικρόφωνο. My apologies. Μάλιστα, ωραία. Καταρχά θέλουμε να συμβάλλουμε στην εξαιρετική δουλειά που έκανε ο αναφέρον κ. Μπρούνι που επέβαλε νέα αποδεικτικά στοιχεία Περιλαμβάνει δε στοιχεία τα οποία διαφέρουν από τις υποχρεώσεις αναφοράς των κρατών μελών. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις επίσημες εκθέσεις του κράτους μέλους σε σχέση με που αναφέρεται σε προηγούμενα έτη όπου η οικολογική ε, κατάσταση της λίμνης ήταν ακόμα καλή. Πιο πρόσφατες όμως αποδείξεις που μας έδωσε ο, που υπέβαλε ο αναφέρον, η οικολογική κατάσταση της λίμνης είναι ε, τώρα ε, επαρκή. Σε αυτό μπορεί να αποτελεί παραβίαση της οδηγίας πλαισίου όσον αφορά το άρθρο 4 τις οδηγίες για τα είδατα και σαφώς δηλώνει την αρχή της μη επιδίνωσης. Η προσωρινή επιδίνωση της κατάστασης των υδάτων δεν θα πρέπει να παραβιαστεί εάν αυτό είναι αποτέλεσμα περιστάσεων φυσικής, ε, ε, φυσικών αιτίων ή ανωτέρας βίας που είναι εξαιρετική, που δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ιδιαίτερα συγκεκριμένα πλημμύρες ή ξηρασία. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτές οι, η πιθανή επιδείνωση ε, υπόκειται σε πολύ αυστηρούς όρους, ε, ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις. Ενώ τα γραφήματα που επέφερε, υπέβαλε στην προσοχή σας ο κ. Μπρούνη δείχνουν ότι αυτό ήταν προβλέψιμο. Κατά συνέπεια, η Κομισιόν θα ερευνήσει περισσότερο αυτή την υπόθεση ε, και Είμαστε ευγνώμονε για την προσοχή που δώσατε στο συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκασπαρινέτη, πράγμα που επιβεβαιώνει τα όσα δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο αναφέροντας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Ωραία λοιπόν και τώρα το λόγο μπορούν να πάρουν οι συνάδελφοι. Ναι, σας είδα, αλλά δεν βλέπω το όνομά σας. Ταμπουράνο. Ταμπουράνο. Non ha potuto eh, elencare tutto. Ο κύριο Σταμπουράνο. δεν μπόρεσα να ιεραρχήσω τι διάφορε ερωτήσει. Θέλω μόνο να πω και τα όσα εκείνο δεν μπόρεσε να πει. Ο κίνδυνο που προβλέπεται από την ε, γεωθερμικό σταθμό του Καστελ Τζόρτζιο, που θέτει ακόμα, είναι ακόμα μεγαλύτερο για την ποιότητα των υδάτων τη λίμνη. Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι και εγώ προσπαθώ να είμαι σύντομο. Κάθε 24 ώρε ένα όγκο γεωθερμικών ε, υγρών, 9 με 10 Ολυμπιακών ειδικών διαστάσεων πισίνες ε, ε, ε, ρίπτονται και μεταφέρονται σε χιλιόμετρα απόστασης και άρα το σημείο ρήψης και το σημείο ε, ε, της έρευνας δεν είναι πάντοτε δεν συγκοινωνούν. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτή, αυτή τα γεωθερμικά υγρά υπόκειται σε πολύ τεράστια πίεση και μάλλον θα υπάρξει ρήξη και θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και η λίμνη. Άρα λοιπόν ο υδροφόρος ορίζοντας και η λίμνη ακόμα και αν ελαφρώς υπάρξει ρήγμα στο αδιάβροχο φράγμα το οποίο έχει φτιαχτεί. Βλέπουμε ότι ακόμα και όταν χυθεί πετρέλαιο στην θάλασσα μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα ε, με τις τεχνολογίες που έχουμε σήμερα. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν συστάσεις, συγκεκριμένες οδηγίες και υπάρχουν συστάσεις και για να αποφευθεί το φράκινγκ. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα για τις ακόμα πιο επικίνδυνες γεωθερμικές γεωτρήσεις. Γι' αυτό ε, ζητώ η Κομισιόν να μελετήσει αυτού του είδους τα προβλήματα ε, που δεν υπάρχουν μόνο στην Ιταλία αλλά και σε διάφορα κράτη της Ένωσης και να αξιολογήσει εις βάθος την ανάγκη πρότασης ad hoc νομοθεσίας για την ε, έρευνα και την γεωθερμική γεώτρηση εντός, σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερο αίτημα προς τους συναδέλφους εδώ να σας παρακαλώ να, παρα... να κρατήσετε αυτή την αναφορά ανοιχτή και αν είναι δυνατόν να επισκεφθείτε και προσωπικά το μέρος, ε, το χώρο στον οποίο αναφέρεται αυτή εδώ η αναφορά. Σας ευχαριστώ. Mr. Mandel. Thank you, Madam Chair. Uh, also want to thank Mr. Bruni for visiting us and being on. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρούνι που ήρθε και που μας ε, ε, έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία. Ακούσαμε με προσοχή τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που είπε ότι θα ερευνήσει περαιτέρω αυτό το θέμα και έτσι μπορώ να πω εξ ονόματος του ΕΛΚ ότι προτείνουμε να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά για να περιμένουμε περισσότερα αποτελέσματα από πλευράς της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον αναφέροντα τον κύριο Μπρούνη δεν είναι η πρώτη φορά μάλιστα που έρχεται να μας βρει εδώ σε αυτή την Επιτροπή και να μας ε, παρουσιάσει το είναι αναφορά του που θίγει ένα από τα διάφορα προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρεται αυτή εδώ η αναφορά αλλά είναι πολλά τα προβλήματα που αναφέρει ο αναφέρον ναι, ρήπανση των νερών της λίμνης Βουρσένα και όπως είπε και ο συνάδελφος Ταμπουράνο αναφέρει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι ε, σε σχέση με τις δραστηριότητες γεώτρεσης για την ε, γεωθερμική ενέργεια. Ε, τώρα, για τα όσα είπε για τη θάλασσα. Ε, επίσης είναι σημαντικά και εγώ επαναλαμβάνω το αίτημα ότι πρέπει να στείλουμε αυτές τις πληροφορίες και στις Ιταλικές αρχές που θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ε, κίνδυνους κατασκευής τέτοιου είδους εγκαταστάσεων. Και επίσης να υπογραμμίσουμε προς τις Ιταλικές αρχές ότι η ποιοτική κατάσταση των νερών πολλών ε, υδάτινων πόρων της Ιταλίας είναι πολύ άσχημη και θα έπρεπε να υπάρξει Προβληματισμό ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους ομιλητές στον καταλογό μου. Μπορώ να σας δώσω και πάλι το λόγο κύριε Μπρούνη για να αντιδράσετε σε όσα είπε η Κομισιόν και όσα είπαν οι συνάδελφοι. Μπορείτε να μιλήσετε για άλλα δύο λεπτά. Ε, ε, θέλετε να προσθέσω κάτι για την γεωθερμία. Ωραία. Θα προσθέσω λοιπόν δύο, δύο πράγματα θα πω για την γεωθερμία. Πρώτον, η γεωθερμία βασίζεται σε μία απλή αρχή. Δηλαδή, ότι από την ε, ε, ε, περιοχή στα δεξιά της επανέγχυσης βλέπετε ότι το υγρό ε, ε, ε, κυλάει προς την άλλη πλευρά. Τώρα όμως, εάν στο υπέδαφος δεν είναι δυνατόν να γίνει ο κύκλος, τότε αυτό σημαίνει καταστροφικό αποτέλεσμα γιατί από τη μία πλευρά εγκύεται το υγρό, από την άλλη πλευρά συσσωρεύεται και επομένως μιλάμε για χιλιάδες τόνους ανά ώρα. Ε, αυτό, αυτό όταν συμβαίνει επί 25 χρόνια προκύπτει ε, η καταστροφή. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι εδώ δεξιά έχετε την ε, λίμνη ε, Μπολσένα και βλέπετε τα πρανή δίπλα από την λίμνη που σημαίνει ότι τα, υγρά κυλούν στην ουσία προς την λίμνη και σε πορεία παράλληλη με την ακτή. Αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο για την λίμνη Μπολσένα. Ευχαριστώ. Uh, thank you Ευχαριστούμε κύριε Μπρούνι και ευχαριστούμε πάρα πολύ που θίξατε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και δώσατε τις γνώσεις σας στην ε, Επιτροπή ε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ταλαιπωρηθήκατε ξανά για να έρθετε στις Βρυξέλλες και εύχομαι ασφαλή ε, ταξίδια επιστροφή στην Ιταλία. Θα προσπαθήσω τώρα να ολοκληρώσω το θέμα της αναφοράς, να δούμε τι μέλη γενέστε. Όπως ακούσαμε και από εσά, αλλά και από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, έχουν προκύψει νέα στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί και επιβεβαιωθεί και από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να μας δώσετε γνωμοδότηση γραπτά. Θα σας ζητήσω λοιπόν να μας στείλετε γραπτά την απάντησή σας ε, και μπορούμε να στείλουμε και ε, ε, ε, αυτή την αναφορά και με τις νέες πληροφορίες που έχουμε στην Επιτροπή Περιβάλλον, Επιτροπή Ένβη και να την δούμε από κοινού με άλλα, άλλες αναφορές που αφορούν εξορίξεις, γεωτρήσεις, γεωθερμία κλπ. Να τα δούμε παράλληλα. Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά Συμφωνείτε όλοι εξαιρετικά. Let's move to Mrs. Rosier. Κυρία Ρουζιέρα, έχετε Διαδικαστικό, ναι κυρία Πρόεδρε, έχω ένα διαδικαστικό ε, και ζητώ, ε, ζητώ συγγνώμη από τους αναφερομένους. Ε, δεν ήμουν στην αρχή της συνεδρίασης, αλλά παρακολουθούσα εξ αποστάσεως στο web streaming τις συζητήσεις και εξεπλάγην από τις αποφάσεις, από την αμφισβήτηση μάλλον των αποφάσεων στην αρχή της συνεδρίασης, των αποφάσεων των συντονιστών που μάλιστα επικυρώθηκε η αμφισβήτηση συζήτηση αυτή και από μία ψηφοφορία. Κατά την άποψή μου, ε, η αλλαγή κάποιας απόφασης ε, των συντονιστών ε, με ελλειπή αντιπροσώπευση στην αρχή της συνεδρίασης είναι και παράτυπο, είναι και παράνομο και είναι και ανίκιο. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω ότι και να επιβεβαιώσετε κι εσείς ότι υπερέχει η απόφαση η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση των συντονισμών. Σύμφωνα όμως λέει η πρόταση με τον κανονισμό 205 οτιδήποτε ε, αμφισβητείται μπορεί να αμφισβητηθεί οποιαδήποτε δηλαδή απόφαση των ιστορών μπορεί να αμφισβητηθεί ή στην ε, Επιτροπή στο σύνολό της ε, πρέπει τα μέλη να είναι πάντοτε με φυσική παρουσία από την αρχή της συνεδρίασης. Αυτό είπαν και οι policy advisors και οι συντονιστές συμφώνησαν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να είναι παρόντες οι βουλευτές. Ίσως είναι πρώτη φορά που το βλέπετε εσείς από όταν ήρθατε στο κοινοβούλιο, αλλά έχει ξανασυμβεί, υπάρχει ο κανόνας υπαριθμών 205 και επομένως εγώ δεν μπορώ να ακυρώσω την απόφαση. Ωραία το σημείο σημειώνουμε και ε, τότε ε, στο μέλλον θα πρέπει να περιμένετε ότι μπορούν να υπάρξουν ε, παρόμοιες αμφισβητήσεις συχνά. Δεν ξέρω αν αυτό σας αρέσει και αν αυτό αποφασίζετε, αλλά θα σας, θα σας έρθει μία πλημμυρίδα από τέτοιου είδους αντιδράσεις. Πρόεδρος, δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι απόφαση του συνόλου της Επιτροπής και παρακαλώ πολύ να διαβάσετε προσεκτικά τον κανονισμό. Είναι ο κανόνας 2.0 μηδέν Όχι, δεν θέλει κανένας να πάρει το λόγο. Πολύ ωραία, περνάμε επομένω στην επόμενη αναφορά που είναι η 0614 εξ ονόματος ε, του φόρουμ Meetup Κασάνα ε, του, ε, κυρίου, του Λάρι Movimento για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας σε μια περιοχή με ιαματικά λουτρά, κατά της εκμετάλλευσης, σε πάση περιπτώσει. Σας έχουν σταλεί τα στοιχεία και θα στραφώ στον κύριο Γκάσπαρινέτη για να μας πει τα τελευταία νέα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή, αλλά και η επόμενη που θα συζητήσετε αμέσως μετά, είναι πολύ παρόμοιες κατά το περιεχόμενο. Πρόκειται για μια ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ στόχων προστασίας του κλίματος και κάποιων ε, τοπικών ε, έργων. Η γεωθερμική ενέργεια είναι μία από τις βασικές πηγές ενέργειας που καλύπτονται από τον κορισμό 2009 2009-09 που εγκρίθηκε το 2009 από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Με την οδηγία, μάλλον πρώτη οδηγίας μπαίνει ένας στόχος 17% δεσμευτικός στόχος άντλησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ήταν σαφές εξ αρχής ότι η υδροελεκτρική ενέργεια και η γεωθερμία θα ήταν οι βασικές πηγές σε ό,τι αφορά την Ιταλία. Η γεωθερμική δεν είναι καλή ή κακή, εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και γι' αυτό το λόγο έχουμε υποχρεωτικές μελέτες αντικτύπου, περιβαλλοντικού αντικτύπου και όπου δίδεται λόγος να πιστεύσει κανείς ότι υπό τις τοπικές συνθήκες ίσως να μην είναι κατάλληλη η γεωθερμική ενέργεια λόγω των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ζήτημα είναι τότε των τοπικών αρχών να σταματήσουν το έργο. Γνωστό είναι αυτό βέβαια και στην περιοχή Κασάνα και για την ε, ε, ύπαρξη αρσενικού στο πόσιμο νερό και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν μάλιστα πλήρωνες αναφορές για τα θέματα αυτά. Όμως αυτά πρέπει να τα αξιολογήσουν οι αρχικές, αρχικώς αρμόδιες τοπικές αρχές. Ξεφεύγει από την αρμοδιότητά μας. Η δε μελέτη αντικτύπου γίνεται ακριβώς για το λόγο αυτό. Εάν θέλετε να υπάρξει ευρωπαϊκή ρύθμιση όπως ζητεί ο κ. υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητεί για την ώρα την αναθεώρηση της συγκεκριμένη οδηγίας και αν μου επιτρέπετε να παραπέμψω στο δικό σας έγγραφο, γιατί περιλαμβάνεται και μια θαυμάσια σύνοψη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση τον Νοέμβριο 2017, όπου περιλαμβάνεται απόφαση εκ νέου παραπομπής στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της θέσεως του Κοινοβουλίου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανανεώσιμες ενέργειες και ιδίως σας επισημαίνω το άρθρο 26 της προτάσεως που μιλεί για βιωσιμότητα, για κριτήρια βιωσιμότητας, ιδίως για βιολογικά καύσιμα και ούτω καθεξής, αλλά προνόμιο του Κοινοβουλίου είναι να επιφέρει τροποποίησης και εφόσον θεωρείτε ότι κάτι παραπάνω πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, ανοίγεται η ευκαιρία εκεί στην διαδικασία συναπόφασης και όχι σε αναφορά που βεβαίως το περιθώριο εκεί ενεργειών μας είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Σας ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος, να προχωρήσουμε στην λήψη μιας αποφάσεως για όλες αυτές τις αναφορές με παρόμοιο τρόπο. Ας περάσουμε στο επόμενο που είναι η 621 σχετικά με την αναστολή γεωθερμικών γεωτρήσεων. Εδώ η κυρία Γκαλιέρο εκπροσωπεί τον αναφερόμενο και λαμβάνει το λόγο για δύο λεπτά. Ah, ok. Eh, eh, Ευχαριστώ την Κομισιόν που ε, ακούει τα όσα έχω Στην αναφορά λέμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της ε, Ιταλίας, ε, τη Ρώμη, υπάρχει ένα project για ε, γεωτρήσεις σε τέσσερα πηγάδια που θα φτάσουν τις 4.000 μέτρα βάθος για να βρουν θερμότητα για βιομηχανικό και κερδοσκοπικό σκοπό να εκμεταλλευτούν δηλαδή τις διάφορες νομοθεσίες που προκύπτουν απορρέων από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009-28 για την ε, ε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, όμως το, και μάλιστα το ποσοστό της ενέργειας που θα παράγεται είναι περισσότερο από τα μεγάλα αιωλικά πάρκα. Φαίνεται λοιπόν σαφές ότι η γεωθερμοηλεκτρική ενέργεια, εάν δεν ε, έχει κίνητρα, δεν τη δόθουν μάλλον κίνητρα, δεν θα είναι ανταγωνιστική με τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το project αυτό που ονομάζεται πρίμα αφορά το εν λίμνη του που περιλαμβάνει τουριστικούς χώρους, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι πλούσια σε γεωργικές περιοχές, SIC, ZPS, σημαντικές περιοχές ή περιοχές Natura 2000 αλλά και ε, περιοχές ε, ε, ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης, δηλαδή ε, παραγωγής ε, τροφίμων ψηλή ποιότητας. Ο αντίκτυπος αυτών, αυτής της γεωθερμικής ε, ενέργειας θα είναι καταστροφική, γιατί παράγει ε, ψευδάργυρο, ράδιο και διάφορα άλλα στοιχεία που μπορεί να εκλειθούν στον αέρα και μπορεί να ε, ρηπάνουν και ποτάμια αλλά και υδροφόρους ορίζοντες. Ε, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για αυτό το project λέει ότι μπορεί να υπάρχουν και, και θείουχα αέρια τα οποία εκλείονται θικόξη, το οποίο εκλείεται στην ατμόσφαιρα. έχουμε τεράστια συγκέντρωση ε, που μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό είδημα. 530 ppm ε, πρόκειται να είναι η έκκληση. Πρόκειται για πολύ ψηλές συγκεντρώσεις, ε, τις ψηλότερες σε ολόκληρη την Ιταλία. Τώρα, η εταιρεία αυτή βάζει και μια τιμή στις εκπομπές σε ppm 295 γραμμάρια την ώρα. Επιπλέον αυτό το project για αυξάνει τους υγειονομικούς κινδύνους γιατί η οι θα εκτίθεται και στο αρσενικό λόγω όλες αυτής της δραστηριότητας οι δε επιχειρήσεις ε, εξαγωγής και επανέρχησης γεωθερμικών υγρών μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και σεισμούς. Αυτό που θέλουμε να θυμίσουμε είναι ότι όλα αυτά είναι αντίθετα στις ευρωπαϊκές οδηγίες 98, 83, 2001, 60 του 2000, 99 του 13, 35 του 4, 18 του 12, 50 του 8, 62 του 96, 81 του 2001, 29 του 96 ευρατόμα και 75 του 2010, καθώς και την 87 του 2003. Όλες αυτές είναι οδηγίες που σχετίζονται με, το, με τις οριακές τιμές των ρήπων, των, επικίνδυνων ουσιών, την αρχή του «ο πληρώνει», την προστασία της κατάστασης των υδάτων, ε, και πρότυπα ασφάλεια για, τους, για τον πληθυσμό. Ζητάμε λοιπόν επί τη βάση του άρθρου 44 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 227 τη Εθνικής Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης πάυση των ε, γεωθερμικών ε, γεωτρήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε σεισμούς και θέτουν τους Ευρωπαίους πολίτες σε πολύ ψηλούς περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους. Ε, και μάλιστα οδηγούν σε απώλεια αξίας των ε, κτηρίων αλλά και των γεών καθώς και ε, διατηρούμε το δικαίωμά μας να ε, στραφούμε κατά του κράτους επί τη βάση όλων αυτών των άρθρων. Κύριε, Κασπαρινέτη, με συγχωρείτε που σας ενοχλώ κάπου κάπου. Για τελευταία φορά όμως τώρα σας καλώ να λάβετε το λόγο και μετά θα σας δώσω διάλειμμα καθήκον μου, το καθήκον μου και ευχαρίστηση άλλωστε. Κυρία Πρόεδρε, θα απαντήσω στα Ιταλικά γιατί χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι ε, όροι τους οποίους θα ήθελα να ε, αναφέρω στην ίδια γλώσσα. Ακούω να γίνεται λόγος για παύση μορατόριουμ γεωτρήσεων ή ε, γεωθερμικών. Αναφέρεστε στην, στο, γιατί έχει αυξηθεί εκεί το αρσενικό στα βραχώδη στοιχεία ή είναι ευρωπαϊκού επίπεδου. Ε, επίσης ε, υπάρχει μία μετατόπιση ε, Επομένως, γιατί υπάρχει ήδη μία υποσυζήτηση πρόταση οδηγίας ε, η οποία αυξάνει ε, τις υποχρεώσεις ε, των κρατών μελών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο μίξ έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και είναι σαφές ότι μία παύση, ένα μορατόριουμ σε γεωτρήσεις υδροθερμικές, γεωθερμικές συγγνώμη, οπωσδήποτε θα αντιτίθεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου και της ε, Κομισιόν. Ε, βέβαια δεν ξέρω, ε, εγώ είμαι τεχνικός της Κομισιόν, δεν μπορώ να πω κάτι για το Κοινοβούλιο. Όμως, εάν το μορατόριο μου στο οποίο ο αναφερόμενος ε, αναφέρεται ε, αφορά μονάχα το συγκεκριμένο τοπικό περιβάλλον, ε, τότε θα πρέπει να δούμε εάν και κατά πόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες της συγκεκριμένη περιοχής μπορούν πράγματι να δημιουργήσουν, να προκαλέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, τότε θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επιληφθούν του θέματος. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε μονάχα σε τοπικό επίπεδο και σε τοπική κλίμακα να προκύψουν προκύψει αυτό το μορατόριου όσον αφορά τις γεωθερμικές γεωτρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, ερωτήσατε λοιπόν την αναφερομένη κυρία Μιράντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με διαφορί πολύ ε, αυτό που είπε η αναφερόμενη σχετικά με τα Μπεκερέλ ε, γιατί εδώ υπάρχει η οδηγία η οποία ε, πρέπει η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία μέχρι την 8η Φεβρουαρίου εάν δεν κάνω λάθος η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη στα στοιχεία γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι ο καθαρισμός του ραδίου θα πρέπει una jornada, una audición sobre el του ε, ε, Ράδο είναι συγκεκριμένη ε, και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα οπωσδήποτε και στους ανθρώπους, μπορεί να μολύνει σχολεία, σπίτια κτλ. Ζητώ λοιπόν από την αναφέρουσα να μου πει ε, ε, υπάρχουν ε, γειτονικά σπίτια, γειτονικές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεαστούν γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υποστηρίξει η ομάδα των Πρασίνων μια τέτοια διαδικασία. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο προς ώρας. Α, και εσείς. Ο κύριος Ταμπουράνο. Ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο το θέμα όσον αφορά την διαδικασία συναπόφασης. Εμείς ε, προτείναμε και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Στρασβούρου τη 17η Ιανουαρίου του 2018 και στα πλαίσια της νέας οδηγίας ε, για τι ε, ανανεώσιμε πηγέ στην τροπολογία 36 που αναφέρει ότι σύμφωνα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά μιας χώρα, είναι πιθανόν οι γεωθερμικέ δραστηριότητε να προκαλέσουν έκκληση αερίων, του θερμοκηπίου κλπ. Και βεβαίως έχουμε κάνει και κάποια άλλα στοιχεία ε, τα οποία ακούσαμε και προηγουμένως και τα οποία βρίσκονται και ε, στα σχετικά έγγραφα. Επομένως, ε, οι επενδύσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλεγούν περιπτώσεις οι οποίες δεν θα δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναφέρθηκε ε, ε, γενικώ ε, στις γεωτρήσεις, αλλά για συγκεκριμένες περιπτώσεις που κολλάνε με το Λάτσιο και με άλλες συγκεκριμένες περιοχές στην Ιταλία και που είμαι σίγουρο ότι θα, ότι θα αποτελέσουν ε, αντικείμενο μελλοντικών αναφορών. Ε, μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 λέμε και συνεχίζει η τροπολογία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να κάνει έναν πλήρη κατάλογο όλων των στοιχείων που εκλείονται από τη γεωθερμική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένου και του διοξιδίου του άνθρακος. Αυτό είναι μια αιτιολογική σκέψη. Εδώ βρισκόμαστε σε φάση τριμερών διαλόγων και επομένως δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα καταλήξει αυτή η αιτιολογική σκέψη. Ωστόσο, εσείς ε, από την Κομισιόν ε, έχετε την ε, δυνατότητα και την πρωτοβουλία να παράγετε νομοθεσία. Εδώ λέμε ότι έχουμε μια αναφορά που προέρχεται από την Ιταλία, αλλά στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να προκύψουν και άλλε αναφορέ για τη γεωθερμική ε, δραστηριότητα. Εμείς δεν ζητήσαμε μορατόριου για τη γεωθερμία γενικά, αλλά να μελετήσουμε σε ποιες και υπό ποιες περιπτώσεις η γεωθερμία μπορεί ε, όχι να μην είναι ανανεώσιμη, αλλά να μην είναι βιώσιμη για το κλίμα, για την ε, ζωή των ανθρώπων και των ζώων. Αυτό είναι το, το δικό μας πλαίσιο, η δικιά μας τοποθέτηση. Στον τριμερή διάλογο θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να παραμείνει αυτή η ατολική σκέψη, αλλά η Κομισιόν, ε, άσχετα από το εάν τελικά θα υπάρχει στο κείμενο αυτό το, ε, αυτή η ατολική σκέψη, οφείλει, λέω, η Κομισιόν να μελετήσει το θέμα έτσι ώστε να δει ποια είναι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της αναπερίπτωση και να προχωρήσει στις απαραίτητες και σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στην επόμενη αναφορά. Είναι και όλες πάνω στο ίδιο θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν και οι αναφερόμενοι να παρακολουθήσουν τι έχουν να μου πούν οι μεν και οι δε, αλλά και για μας να δούμε να φωτιστεί το θέμα από διάφορες πλευρές. Θα προσπαθήσω επίσης να συζητήσω μαζί τα θέματα 16 και 17, ώστε να μπορέσει να απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα δυο μαζί. Τώρα έχω την 829 και την 1185 και την 845. Αυτές όλες, τις τρεις δηλαδή, θα τις συζητήσουμε μαζί. Σας διάβασα τα ονόματα. Η αναφερομένη λέγεται Σίλβια Περφέτη και νομίζω μάλιστα έχει και μια παρουσίαση PowerPoint. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να σας δείξω ποιοι είναι οι βασικές πτυχές της γεωθερμίας στην νότια Τοσκάνη της Ιταλίας. Αυτή η κατάσταση αποτελεί το τέλος ενός μύθου, γιατί η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι πράσινη. Οι κλινικές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν υπάρχει ένα όριο κάτω από το οποίο να μην μπορούμε να δούμε την επιρροή της ρήπανσης στην υγεία των ε, κατοίκων και περίκων. Η υπηρεσία περιβάλλοντος του Σκάνες δείχνει ότι οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις ε, εκπέμπουν ε, σε δάργυρο και θικό οξύ ε, και ότι οι, οι τιμές του ψευδάργυρου είναι 17 φορές ψηλότερες στη, γύρω από τις εγκαταστάσεις αυτές. Το 2008 είχαμε αυτό το χάρτη που δείχνει την ε, ρήπανση σε ψευδάργυρο στον Δήμο Πιαν Καστανάιο. Ε, Έχουν δε και αμμονία το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει τις εκπομπές αμμονίας στην ε, ζώνη ε, όπου λειτουργούν αυτές οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις. Εδώ έχουμε τη χωροταξία του 2008 και έχουμε τις ετήσιες εκπομπές αμμονίας στον Δήμο Πιάν Καστανάριο. Η αμμονία μεταφράζεται σε αύξηση των μικροσωματιδίων PM10 και PM2,5 ε, δευτερογενούς προέλευσης. Ε, αυτά συμβάλλουν για το 51, κατά 51% στην εκπομπή αμμονίας ε, στην περιοχή της Τοσκάνης. Σε τούτο το άρθρο που προκύπτει από διεθνείς έρευνες αναλύονται τα μη συμπυκνώσιμα αέρια που εκπέμπονται από τις γεωθερμικές, γεωθερμικές εγκαταστάσεις Μοντα Μιάτα που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, ε, μεθάνιο και άλλα. Στο τέλος του άρθρου λέει ότι αυτού του είδους τα εγκαταστάσεις λόγω των αερίων που εκπέμπουν, που είναι βλαβερά για το, ε, για το κλίμα, ναι, δεν μπορούν να θεωρηθούν carbon free. Το 2010 υπευλήθη από την Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας της Ζωσκάνης η πρόταση επιδημιολογικές μελέτες για να κατανοήσουμε την επιρροή της εκπομπής των αερίων αυτών στην υγεία των ε, γύρω πληθυσμών. Συγκρίθηκαν λοιπόν, συγκρίθηκε η κατάσταση της υγείας των κατοίκων στο βόρεια και στη νότια ζώνη σε σχέση με αυτή ε, κατοίκων 50 χιλιόμετρα πιο μακριά. Ήταν λογική η σύγκριση και με την περίοδο 2000 με 2006 τα αποτελέσματα της γενικής συναισιμότητας για την περίοδο 2000 με 2006 για τους πληθυσμούς που κατηγούν στην γεωθερμική περιοχή ήταν υψηλότερη στους ε, άνδρες κατά 13,1% σε σχέση με τους δήμους που βρίσκονται 50 χιλιόμετρα πιο μακριά. Με εχμές στον δήμο του Πιάν ε, Καστανάιου που έφτασαν στο 27%. Τα αποτελέσματα θρησιμότητας λόγω καρκίνου ε, ήταν ανώτεροι στους άνδρες κατά 19% σε σύγκριση με τους Δήμους που βρίσκονται 50 χιλιόμετρα πιο μακριά, με χμή στον Δήμο Πιάν Καστανάγια, Παντία Σαν Σαλβατόρο και Αρσιντόσο, που έχει φτάσει στο 30%. Στα συμπεράσματα η μελέτη λέει πως υπάρχουν επιστημονικά όρια, αλλά ότι οι περιοχές αυτές αναφέρουν περισσότερα, ε, ε, στο νότο ε, αναφέρουν περισσότερα προβλήματα υγείας από ότι αυτές που βρίσκονται βόρεια. Και αυτό οδηγεί στο να σκεφτούμε γενετικούς, γενετικά αίτια ή σε λάθος στυλ ε, ζωής. Η ίδια όμως υπηρεσία της Τοσκάνης μας παρουσίασε μελέτη που έκανε η ίδια διενήργησε η ίδια, όπου επιβεβαιώνω ότι δεν υπήρχε διαφορετική στυλ ζωή οι άνθρωποι που ζούσαν γύρω από τις εγκαταστάσεις σε σχέση με αυτούς που ζούσαν στα 50 χιλιόμετρα μακριά. Τα αποτελέσματα της επόμενης μελέτης θα τα δούμε όμως μετά από αρκετά χρόνια. Ε, Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αντίφαση στην πολιτική αυτή τη Ένωση ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο τη συνθήκη για την ε, Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωση, είναι το άρθρο 11 και το άρθρο 191 ε, και λέει ότι λέει για προστασία του πολίτη και ακόμα και ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το άρθρο 37 που προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντο καταπατώνται. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. For... Η πρόεδρο, κυρία Βίξτρομ, σα ευχαριστώ. Χρησιμοποίησατε τον χρόνο που σα διαθέσαμε με εξαιρετικό τρόπο. Να προχωρήσουμε στην επόμενη, υπαριθμόν 17, 0845 του κυρίου Ντάριο Ματσαλούπη. Ευχαρίστω θα σας δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε. Στην αναφορά εμείς ε, καταγγέλουμε την έλλειπη εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, την βιοπικιλότητα, ε, την προστασία του εδάφους. Ε, έχουμε επίσης και καταπάτηση της οδηγίας των πτηνών, καθώς επίσης και την 2008 κάθετος 50 και την 2012-18. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009-28 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν λαμβάνει υπόψη στοιχεία βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα ζητούμε να, ε, προ... να υπάρξει και ε, μία άκαμπτη παράμετρος η οποία θα αφορά τη γεωθερμική δραστηριότητα έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, ρήπανση των μόλυνση των υπογείων υδάτων. Ε, στην αναφορά αναφέρουμε μία σειρά από συγκεκριμένες περιπτώσεις φράκινγκ ε, ε, καθώς επίσης και για περιπτώσεις όπου στην Βασιλεία ας πούμε στην Ελβετία δημιουργήθηκαν ρογμές σε γειτονικά σπίτια λόγω ακριβώς των γεωτρήσεων και εν τέλει το το πρόγραμμα αυτό εγκατελείφθη. Ε, είναι δυνατόν λόγω ακριβώς των μεγάλων των γεωτρήσεων και σε μεγάλο βάθος μπορεί να αυξηθεί η σεισμική δραστηριότητα. Στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Ισλανδία, στην Γερμανία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ήδη ενώσεις πολιτών που προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτού του είδους τις γεωτρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις ε, είναι οι οι συγκεκριμένες παράμετροι για τις γεωτρήσεις, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να συσταθεί μια ανεξάρτητη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μελετά το θέμα αυτό, όπως συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, ζητούμε οριστικό μορατόριο όλων των ε, ε, κέντρων γεώτρησης flash και επίσης ζητούμε ε, για τις περιπτώσεις PM10 και PM2,5 λαμβάνοντας υπόψη τον, ε, το ποσοστό του υδραργύρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ε, της αμμονίας παράγεται ακριβώς στην περιοχή της Τοσκάνης και ότι αυτού του είδους τα στοιχεία μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα μη συγκμικρούμενα στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα άσχημα για την υγεία και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ε, υπάρξει ε, με μεγάλη συγκέντρωση αρσενικού στον υδροφόρο ορίζοντα, πράγμα που βεβαίως έρχεται ε, σε αντίθεση με την ε, οδηγία η οποία αφορά την καλή ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, τον ΕΚ 2008, το 513, του 2014-17 και ε, μία σειρά άλλων οδηγιών από τις οποίες ε, προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες γεωθερμικές εγκαταστάσεις ε, προκαλούν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά και πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα από ό,τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, επίσης, ε, να μην λησμονούμε ότι στο άρθρο 227 της Συνθήκης Λειτουργίας αναφέρεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται μία πάυση των γεωθερμικών γεωτρήσεων ε, και αναφέρεται επίσης ότι τα, οι ζημιές οι οποίες μπορούν να προκληθούν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης, ζητούμε να υπάρχει μία ελάχιστη απόσταση των γεωτρήσεων του τουλάχιστον 35 χιλιόμετρων από κατοικημένες περιοχές. Επίσης, ε, να ε, ξεχωρίσουν ε, αυτές οι ανανεώσιμες πηγές οι οποίες είναι βιώσιμες, όπως είναι φωτοβολταϊκά και αιωλικά και οι μη βιώσιμες, όπως είναι η γεωθερμία. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν καλύτεροι ε, σωρευτές και γεννήτριες όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη γεωθερμία. Ε, πρέπει όμως να πούμε ότι τα χρήματα κιόλας είναι πάρα πολλά διότι την γεωθερμία την έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και η Ιταλία αλλά και όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι στην, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται μη καθαρές μορφές ενέργειας. Ε, υπάρχει εδώ λοιπόν ε, μία ε, ένα κενό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και το κενό αυτό ακριβώς προκαλεί σενάρια τα οποία είναι ιδιαιτέρως δύσκολα και επικίνδυνα. Υπό το φως όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 2.27 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούμε και βάσει του άρθρου 2.28 μια τελείως διαφορετική νομοθετική προσέγγιση, ρυθμιστική προσέγγιση όσον αφορά την γεωθερμία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Χος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ήλθατε να μιλήσετε και για τα δύο αυτά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης, 16 και 17. Ε, thank you, Chair. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. η γεωθερμική ενέργεια γενικά. Είναι πολύ λιγότερο ρηπογόνα από τα ορυκτά καύσιμα, από την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, τα γεωθερμικά εργοστάσια αποδίδουν 5 περίπου τις 100 διοξιδίων του ανθρώπου και λιγότερο από 1% οξυδίων του αζότου. Σε σύγκριση με ισοδύναμα εργοστάσια που και άνθρακα. Και για άλλα αέρια είναι σχεδόν μηδενικές οι εκπομπές τους. Όμως, όπως λέχθηκε από τους αναφερομένους, Εξαρτάται αυτό από τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα ή αποδοτικότητα των ε, εγκαταστάσεων και των σχετικών φίλτρων από υπόγεια στρώματα. Οι πραγματικές εκπομπές σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως είναι υψηλότερες από τα ποσοστά που ανέφερα. Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές είναι βέβαια ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος, όπως του Σχεδίου Στρατηγικής Τεχνολογίας, που περιλαμβάνει και τη γεωθερμία Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές από γεωθερμικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, αυτές ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία, μεταξύ άλλων και από την οδηγία περιβαλλοντικού αντικτύπου, αλλά και από άλλες οδηγίες, τις οποίες ανέφεραν και αναφερόμενοι προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Αυτάς Νομοθεσίας από τις Ιταλικές Αρχές και θα αναλάβουμε την κατάλληλη δράση εάν διαπιστώσουμε ότι οι Ιταλικές Αρχές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες, στα απαιτούμενα πρότυπα. Σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, οι χώρε μέλη είναι υποχρεωμένε να τις αναφέρουν στο διεθνέ Πάνελ Κλιματικής Αλλαγής, δηλαδή σύμφωνα με τις κατευθυντές γραμμέ του διεθνού Πάνελ, τονίζουμε ωστόσο ότι ορισμένες φορές δεν είναι εύκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε ανθρωπογενείς εκπομπές και σε εκπομπέ που προκαλούνται με φυσικό τρόπο από τη φύση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μελέτη επί του παρόντος για τις εκπομπές γεωθερμικών εργοστασίων που θα μας προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή όμως και όπως είπα προηγουμένως τα γενικά χαρακτηριστικά της γεωθερμικής ενέργειας ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας είναι ότι έχει πολύ χαμηλότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και πολύ χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα ισοδύναμα εργοστάσια ορυκτών καυσίμων, δεν θεωρεί σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ώρα να ρυθμίσει με κριτήρια βιωσιμότητας μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας. Είμαστε ωστόσο διατεθειμένοι και διατεθειμένες να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα και προβαίνουμε σε ανάλυση και έχουμε αρχίσει να κάνουμε τα σχετικά βήματα για να μπορέσουμε στην βάση αυτών να αναλύσουμε τα θέματα που θέτουν οι αναφερόμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τον λόγο μπορούν να λάβουν οι συνάδελφοι και πρώτος ο κύριος Ταμπουράνο. Συνάδελφε, καταρχά είναι αλήθεια ότι πρέπει να γίνονται μελέτες ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου για τα γεωθερμικά εργοστάσια, όπως ε, και για τις ε, υπόλοιπε μεγάλε υποδομέ, Αλλά δεν υπάρχουν ειδικέ μελέτες για αυτού του τύπου τις γεωθερμικές εγκαταστάσεις. Και άρα λοιπόν θα έπρεπε να μιλάμε για γεωθερμία και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια είδη γεωθερμίες για τις οποίες οι εκπομπές ανά κιλοβατόρα διοξιδίου του άνθρακα είναι χαμηλότεροι από ότι όταν και έχονται στερεά καύσιμα. Ναι, ορυκτά καύσιμα, με συγχωρείτε. Όμω, ορισμένε από αυτέ τι εγκαταστάσει που λειτουργούν και θα λειτουργήσουν και στο μέλλον με ανοιχτό ε, ε, κύκλωμα τύπου flash φαίνεται ότι εκπέμπουν ε, περισσότερα αέρια και όχι μόνο διοξείδιο του άνθρακα από ότι οι θερμοελεκτρικοί ε, σταθμοί που τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα. <clears throat> και αυτό έχει αποδειχθεί με μελέτες. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις ε, εκπομπέ που είναι ε, βλαβερές για το περιβάλλον των διαφόρων τύπων γεωθερμικής τεχνικής, αλλά είναι ένα, μια μεγάλο, ένα μεγάλο φάσμα ε, γεωθερμικές εγκαταστάσεις και εξαρτάται και από το, περιοχή στην οποία λειτουργούν τα εργοστάσια αυτά. Τώρα για την Ιταλία, εγώ θέλω να τονίσω ότι τα γεωθερμικά, τα γεωθερμικά εργοστάσια, αν και εκπέμπουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα, παίρνουν ε, τα βοήθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη ε, των στόχων για το κλίμα. Έχει γίνει βραχικύκλωμα λοιπόν και χρειάζονται περαιτέρω μελέτες. Χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση αυτά τα αέρια μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και εδώ υπάρχει θέμα χρονισμού, ρυθμού με τον οποίο μπαίνουν στην ατμόσφαιρα αυτά τα, φυσικά, αυτά τα αέρια, γιατί δεν είναι φυσικές εκπομπές. Λέμε για εκπομπές σε διοξιδίου του άνθρακα, σε γεωλογικού και μορφή. Οι ανθρώπινες όμως εκπομπές που θα γίνονταν κανονικά σε εκατομμύρια χρόνια, εδώ γίνονται μέσα σε λίγα χρόνια. Δεν είναι λοιπόν μόνο η ποσότητα, αλλά είναι και ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται το διοξίδιο του άνθρακα και η συγκέντρωσή του στην και αυτό προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές. Τέλος, αναφέρομαι και στο ψευδάργυρο. Ιδράργυρο, με συγχωρείτε. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μελέτες γίνανε από το 2007 στην Τοσκάνη και έχουν γίνει μετρήσεις και λένε πόσο εκπέμπεται σε ένα χρόνο 22,5 τόνοι υδράργυρου σε περίπτωση που σπάσει ένα θερμόμετρο, φανταστείτε, έχει 2 γραμμάρια. Εδώ μιλάμε για 750.000 θερμόμετρα που σπάνε και ρίχνουν τον υδράργυρο στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο χωρίς κανένα είδου έλεγχο. Δεν μπορεί να το αγνοεί αυτό το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και οι αρμόδιες αρχές. Μέχρι πέρσι τα κράτη-μέλη δεν ήταν υποχρεωμένα να αναφέρουν τον υδράργυρο που εκπέμπουν ε, αυτές οι εγκαταστάσεις με βάση τις οδηγίες της Ένωσης. Μόνο το 2017 εισήχθη υποχρέωση να ενημερώνουν για, αυτό, για αυτούς τους όγκους. Η Ιταλία δεν έχει ενημερώσει. Κάναμε προφορική ερώτηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα η Ιταλία γιατί μπορεί η Ιταλία να μην σέβεται τους ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Mandel. Thanks to everybody for... Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντλ, ευχαριστώ ε, για την εξήγηση όλων αυτών των λεπτομεριών. Η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις αναφορές είναι βεβαίως να διατηρηθούν ανοιχτές διότι βεβαίως δεν υπάρχει ακόμα επαρκής πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ορισμένες μάλιστα δεν υπάρχει καμία πληροφορία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως σε ό,τι αφορά την 829 εμείς προτείνουμε να διαβιβαστεί στις Επιτροπές Ήτρε και ΕΝΒΙ για να ε, δώσουν ε, περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ, να παρέμβω και εγώ για να επαναλάβω ότι αυτό το, αυτή η αναφορά προφανώς πρέπει να μείνει ανοιχτή. Όλες αυτές οι αναφορές πρέπει να μείνουν ανοιχτές. Συμφωνώ με τα όσα πρότεινε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Είναι σαφές και προφανές ότι αυτές οι αναφορές ε, ρίχνουν φως σε μεγάλες ελλείψεις ε, της ε, νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υποδορέσει να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για να ρυθμίσει αυτόν το τομέα που μέχρι σήμερα λοιπόν λοιπόν ε, δεν έχει ε, ε, δεν διέπεται από τους σωστούς κανόνες για την προστασία της υγείας και του κλίματος. Ακούσαμε μαρτυρίες πολύ συγκεκριμένες και ακριβείς σε σχέση με το ποιο είναι το πρόβλημα. Να αναφέρω μόνο τελευταία που δεν τη συζητήσαμε αλλά που μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική είναι η, η οι σεισμοί που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις εγκαταστάσεις σε μια χώρα όπως η Ιταλία πάνω απ' όλα, που η Ιταλία κι αν έχει υποφέρει πολλές φορές ε, από δραματικούς σεισμούς, ε, ακόμα ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ώστε αυτές οι αναφορές να μένουν ανοιχτές και δραστηρίες για να δραστηριοποιηθούμε σε εθνικό και σε κοινωτικό επίπεδο, ώστε να καλύψουμε αυτό το ρυθμιστικό κενό. Επαναλαμβάνω λοιπόν και εδώ ότι πρέπει πλήρως να ενημερώσουμε ενημερωθούν οι διεθνικές αρχέ και οι περιφερειακέ αρχέ σε σχέση με την επικίνδυνοτητα αυτού του είδου των εγκαταστάσεων. Ευχαριστώ. Thank you very much. You are the, the last speaker on... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ήταν τελευταία ομιλήτρια στον καταλογό μου και θα θέλω τώρα να πιστήσω την προσοχή σας στο πώς όλα αυτές τις αναφορές θα τις χειριστούμε. Ε, ναι, θα είναι για κάποιο λόγο που τις βάλαμε από κοινού σήμερα για να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε όλα αυτά μαζί. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε το εξή. Βεβαίω να μείνουν ανοιχτέ όλε οι αναφορέ. Θα στείλουμε επιστολέ στι διάφορε περιφερειακέ αρχέ για να τονίσουμε πώ μα ανησυχεί πολύ η υπόθεση αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απλώς να τους επιστήσουμε την προσοχή στο ότι τα εξετάζουμε όλα αυτά και μετά τις στέλνουμε και στην Ήτρε για γνωμοδότηση. Και στην ΕΜΠΗ ενημερωτικά, όπως είπε ο κ. Μάντελ ε, τελευταία, ε, και τώρα να επαναλάβω ότι τα προβλήματα φαίνεται να είναι ξεκάθαρα, αλλά χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για το πώς θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ, προσέξτε την 614, 621 1185 και 845. Όλες αυτές αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη θερμο... γεωθερμική ενέργεια. Θα αντιστείλουμε λοιπόν ως πακέτο στις δύο επιτροπές και η διαφορά με τις επιστολές είναι ότι θα πάνε και στις διάφορες περιφερειακές αρχές. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και βλέπω πως συμφωνείτε μαζί μου. Οπότε αυτό θα και θα κάνουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους αναφέροντες που ήρθαν μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, που έχετε επενδύσει τον ελεύθερο σας χρόνο και έχετε αφοσιωθεί σε αυτό και μας ε, έχετε ενημερώσει βεβαίω. Και να σας ευχαριστήσω και την ε, Κομισιόν για την σαφή και καλή συνεργασία σε αυτές τις υποθέσεις. Και τώρα θα στραφούμε στο επόμενο θέμα που είναι μια παρουσίαση της μελέτης περί διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώπη, κύρια προβλήματα και καλύτερες πρακτικές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κρίστιαν Νόιμπάουερ που είναι ο διαχειριστής του project, υπεύθυνο του έργου. Καλώς ορίσατε και σας δίνω αμέσως στο λόγο. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή Αναφορών που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα της μελέτης μας. Λέγομαι Νόιμπαουερ, Αυστριακός και έχουμε κάνει μια αξιολόγηση αναφορών που έχουν σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων. Για 20 λεπτά θα με επιτρέψετε να σας εξηγήσω τα συμπεράσματα της μελέτης μας. ορισμένα βασικά τώρα, ε, θα τα περάσω γρήγορα, θα σας εξηγήσω λίγο σχετικά με τα συμπεράσματα πώς έχουμε ταξινομήσει τις αναφορές, ποια θέματα καλύπτουμε. Θα σας πω λίγες πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία στην οποία παραπέμπουν οι αναφερόμενοι. Πολύ σύντομα επίσης σχετικά με το ποιες αναφορές έχουν αναλυθεί και επίσης ποιες, θεω, εξετάσαμε για την ανάλυση. Πολύ σημαντικό επίσης να σας πω λίγα και για τις βέλτιστες πρακτικές. και για ρυθμίσεις που ήδη έχουν ε, υιοθετηθεί σε ορισμένες χώρες μέλη και ορισμένες εν τέλει συστάσεις για μια βελτιωμένη προσέγγιση. ανατέθηκε από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η μελέτη και διεξήχθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αυστριακής Δημοκρατίας στη βάση δεδομένων που ήταν διαθέσιμα από τους αναφερομένους και κάτι που είναι σημαντικό να αναφέρω είναι ότι όλη αυτή η εργασία έγινε βασισμένη στην προηγούμενη αξιολόγηση που είχε διεξαχθεί το 2011. Το 2011 είχαμε αναλύσει 101 αναφορές. Πέρσι το 2017 εξετάσαμε 10. Όλες πάντα σε σχέση με διαχείριση αποβλήτων. Για να σας δώσω τώρα μια σύντομη σύνοψη, ίσως δεν μπορείτε να διαβάσετε καλά τα γράμματα στην ε, διαφάνεια γιατί είναι μικρά, Βλέπετε τέσσερις κατηγορίες, τέσσερις θεματικές κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενο των αναφορών. Στην πρώτη στήλη είναι οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Για το 2017 το γαλάζιο χρώμα, είναι 2017 ξαναλέω, η κόκκινη ε, στήλη είναι από το 2011. Ε, Έχουμε 52 συνολικά αναφορές που αναφέρονται σε διαδικασίες αδειοδότησης των ε, σχετικών εγκαταστάσεων. Η δεύτερη στήλη είναι η λειτουργία υφιστάμενης εγκατάστασης. Τα διάφορα παράπονα, οι διάφορες καταγγελίες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εγκατάστασης. Συνολικά 54 αναφορές αναφέρθηκαν σε τέτοια θέματα από το συνολικό αριθμό των αναφορών που όπως εξήγησα προηγουμένως είναι συνολικά 111. Εκτός αυτού έχουμε τη θεματική περιοχή της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Εδώ έχουμε 28 συνολικά αναφορές, 25 κόκκινες συντριν στο γαλάζιο και ε, η τελευταία αναφέρεται σε νέα θεματική περιοχή που άρχισε να μελετάται μόνο το 2017 και έχει σχέση με την ακατάλληλη διαχείριση ραδιοενεργών αποβλήτων. Τέσσερις λοιπόν θεματικές περιοχές, ας το πω έτσι, που ε, έχουν απασχολήσει τους αναφερομένους. Κάτι που είναι νέο, είναι πάλι για το 2017, βλέπουμε ότι η λειτουργία εφισταμένων εγκαταστάσεων αποτελεί το κύριο θέμα που απασχολεί τους αναφερομένους. Να έρθουμε ε, στον επόμενο πίνακα τύποι εγκαταστάσεων. Οι χωματερές για το 2017 είναι η μεγάλη στήλη που είναι και η πιο η κυριαρχούσα ας πούμε. Ε, συνολικά έχουμε για το 2011 58 αναφορές για χωματερές και 4 για το 2017 στο γαλάζιο τμήμα της στήλης. Άλλο σημαντικό, άλλο σημαντικός χώρος που κινούνται οι αναφορές είναι οι άλλες εγκαταστάσεις όπως αποδίκευσης ή διαχείριση των αποβλήτων. Εκεί έχουμε τρεις ε, αναφορές για το 2017. Πρόκειται για την από αριστερά τέταρτη στήλη. και τέσσερις από βιομηχανική παραγωγή. Και το πολύ νέο ε, πεδίο είναι εξωδεξιά, γαλάζιο, εκεί που λέει άλλες. Και αναφέρονται βέβαια στην διαχείριση ραδιο, ε, ραδιενεργών καταλήπων. Τώρα σε ό,τι αφορά τον τύπο αποβλήτων, βλέπουμε κυρίως στερεά απορρίμματα ε, από δήμους και κοινότητες. Μιουνίσι πάλι δηλαδή, πάλι για το 2017, βλέπουμε τέσσερις και ε, όπως είπα και προηγουμένως το νέο αυτό θέμα ε, ραδιενεργά κατάλοιπα, έξω δεξιά. Βέβαια επικίνδυνες ουσίες και στερεές επικίνδυνες, επικίνδυνα κατάλοιπα ή απόλυτα είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική προοπτική από τις διάφορες χώρες μέλη της Ένωσης, βλέπουμε περισσότερες αναφορές στο νότιο-ανατολικό μέρος της Ένωσης. Εκεί ε, οι αναφερόμενοι συζητούν θέματα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ε, για παράδειγμα στη Γαλλία. Έχουμε αναφορές που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παρόμοια θέματα. Αυτό που κάναμε επιπροσθέτως είναι να ρίξουμε μια ματιά στην ομοθεσία στην οποία παραπέμπουν οι αναφερόμενοι. Και κάνουμε και μια νομική αξιολόγηση, δηλαδή εξετάζουμε ποια άρθρα είναι αυτά που είναι σημαντικά, ποιων κανονισμών και ποια απασχολούν περισσότερο τις αναφορές. Βέβαια πρόκειται ιδίω για το άρθρο 4 της Οδηγίας Πλαισίου και το άρθρο 11, το άρθρο 11 που αναφέρεται στους στόχους της ανακύκλωσης. Αυτά, σε αυτά παραπέμπουν πολύ συχνά οι αναφορές. Δεύτερο, η οδηγία για τους χιτά ή τις χωματερές. Επίσης ε, γίνονται πάρα πολλές παραπομπές σε αυτήν στις αναφορές και βλέπετε και τους σχετικούς αριθμούς σε παρένθεση. Ένα νέο θέμα είναι, όπως εξήγησα, τα ραδιενεργά υλικά, τα ραδιενεργά απορρίμματα. Εκεί έχουμε νομοθεσία που προκύπτει από τη συνθήκη Ευρατόμ Εκεί αξιολογήσαμε τέσσερις κανονισμούς. Πιο σημαντικός, αυτός που είναι αρμόδιος για την διαχείριση των ε, ραδιενεργών καταλήπων και του ραδιενεργού καυσίμου που έχει ήδη καταναλωθεί. Ένα θέμα είναι για την ενδιάμεση αποθήκευση του ραδιενεργού υλικού. Το άλλο είναι οι παράνομες ε, αποθέσεις ραδιοενεργού υλικού και για αυτά τα δύο θέματα βέβαια υπάρχει η σχετική νομοθεσία και σε αυτήν γίνονται πολύ συχνά παραπομπές. Πάλι έρχομαι στις βασικές, ε, στους βασικούς τομείς καταγγελιών. Πρώτα είναι η διαδικασία διοδότησης, ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ακατάλληλη λειτουργία υφισταμένων εγκαταστάσεων. Τρίτος τομέας είναι οι παραλήψεις στα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων γενικά και τέταρτο είναι η ελλειπής διαχείριση ραδιενεργού υλικού ή ραδιενεργών αποβλήτων. Σε αυτούς τους τέσσερις θεματικούς τομείς προσπαθούμε να ε, τονίσουμε τις βασικές ελλείψεις και να κάνουμε και κάποιες συστάσεις για τη σωστή προσέγγιση. Ξαναλέω, δείχνω σε αυτό το γράφημα, βέβαια είναι πάλι πολύ μικρά τα γράμματα, θα δείτε όμως στον ε, πίνακα αυτών ποιες αναφορές αναλύθηκαν για το 2017. Έχουμε δύο από την Ιταλία, αναφέρονται στην περιφέρεια της Καλαβρίας, δύο από την Ελλάδα, κυρίως για χιτά, δύο από την Ισπανία, αφενός για το σχέδιο διαχείρισης καταλήπων και αφετέρου ε, άλλο για, την, για ορισμένες ε, ε καταγγελόμενες ε, παραβιάσεις και τις υπόλοιπες όπως δείτε, ενδεχομένω από την διαφάνεια. Προσπαθούμε να επισημάνουμε και σε ποιους τομείς αναφέρονται οι σχετικές αναφορές, να κάνουμε τη σχετική ανάλυση και να φωτίσουμε τις βασικές ελλείψεις και να κάνουμε και κάποιες συστάσεις σχετικά. Το πρώτο θέμα είναι οι διαδικασίες αδειοδότησης. Ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις που, στις οποίες παραπέμπουν οι αναφορές. Για παράδειγμα, σχετική εγκατάσταση δεν λειτουργεί σύμφωνα με την άδεια που έχει λάβει. Δεν υπάρχει επαρκής εμπλοκή μερών, των ενδιαφερομένων μερών, των stakeholder. Είναι ανεπαρκής η μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον ή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες που να ε, κοινοποιούνται στις αρχές. Οι συστάσεις που κάνουμε προκειμένου είναι γενικού χαρακτήρα. Πρώτη είναι βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των αρχών, των ε, διαχειριστών και όλων των διαφερμένων μερών. Η εισαγωγή συστημάτων ελέγχου και επαλήθευσης για τις ε, μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου, να υπάρχουν επαρκείς διοικητικές ικανότητες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και τέλος να αναπτυχθούν πρότυπα και ακόμα περισσότερο, δηλαδή να προωθηθούν τα πρότυπα για τις ε, συγκεκριμένες ε, βλάβες του περιβάλλοντος. Βέλτιστες πρακτικές τώρα και κανόνες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θελήσαμε εδώ να βάλουμε στην μελέτη κάποια παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών όπου αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που επισημάναμε προηγουμένως και όπου κάποιοι μηχανισμοί έχουν ήδη καθιερωθεί για να βελτιωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την ε, μελέτη αντικτύπου, υπάρχουν βεβαίως ομάδες εμπειρογνωμόνων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, ε, υπάρχουν και διαθέσιμες εκθέσεις για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της οδηγίας μελέτης αντικτύπου στο περιβάλλον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά ως βέλτιστες πρακτικές και ως κατευθυντήρες γραμμές για να επιτρέψουν να εντοπιστούν ε, ποιες είναι οι καλύτερες ε, πρακτικές για το μέλλον. Επίσης βεβαίως δημόσια διαβούλευση. Εκεί υπάρχουν οι σχετικές συμβάσει, η γνωστή σύμβαση του Άρχους Εκεί μπορούν να βρεθούν πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση οι ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει βέβαια και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης το οποίο θεσπίζει πρότυπα και είναι πολύ σημαντικά για τις διαδικασίες αυτές διότι τα πρότυπα δίνουν κάποια κατεύθυνση, ένα προσανατολισμό. Για παράδειγμα πόσο μακριά επιτρέπεται να είναι μια εγκατάσταση ε, καθαρισμού των ε, αποβλήτων ή των ε, νερών της αποχέτευσης από κατοικημένες περιοχές και ούτω καθεξής. Το δεύτερο ε, θέμα είναι οι επιπτώσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Εδώ οι βασικές ελλείψεις που μπόρεσαν να εντοπιστούν είναι πρώτα κίνδυνοι ε, σε βάρος της υγείας και του περιβάλλοντος λόγω της ανεπαρκούς λειτουργίας της εγκατάστασης, δηλαδή υψηλά επίπεδα εκπομπών που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην υγεία, ανεπαρκής έλεγχη και διαδικασίες παρακολούθησης στην φάση λειτουργίας, έλλειψη για παράδειγμα παρακολούθησης ή ε, συστημάτων παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης, ανεπαρκής τεχνική προσαρμογή της υφιστάμενης εγκατάστασης, γνωρίζουμε ας πούμε ότι σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι εγκαταστάσεις πρέπει να υιοθετούν τα βέλτιστα πρότυπα. Ορισμένοι ισχυρίζονται σε κάποιες αναφορές ότι δεν γίνεται αυτό με σωστό τρόπο. Και τέλος, παράνομη λειτουργία εγκαταστάσεων ε, επεξεργασίας καταλήπων ή αποβλήτων. Οι συστάσεις που κάνουμε προκειμένου είναι πάλι γενικού χαρακτήρα και τονίζονται επίσης στη μελέτη μας, δηλαδή να προβλεφθούν διοικητικές ικανότητες ε, των εθνικών, ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση και την παρακολούθηση να γίνονται επιγραμμικές μετρήσεις online δηλαδή για βασικές εκπομπές και παραμέτρους των διαδικασιών να γίνονται επίσης διαθέσιμες online στο διαδίκτυο δηλαδή οι μετρήσεις και να είναι ε, δημόσιο κτήμα για να μπορεί έτσι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού και να εμπλακεί περισσότερο το κοινό ε, στην ε, διαδικασία λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Ξαναλέω να εμπλακεί περισσότερο το κοινό στην λειτουργία της εγκατάστασης. Και τέλος, να γίνονται επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ε, αποβλήτων. Και αυτό έχει σχέση και με, την, με το πρώτο θέμα. Είναι σημαντικό δηλαδή οι αρμόδιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να επιθεωρούν τακτικά τις διάφορες εγκαταστάσεις. Βέλτιστες πρακτικές που προτείνουμε εδώ για τον δεύτερο θεματικό τομέα, ε, για τις υφιστάμενες πάντα εγκαταστάσεις, βεβαίως έχουμε πάλι ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, το ΙΜΠΕΛ που βλέπετε που λειτουργεί καλά, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο δηλαδή, που είναι δίκτυο αρχών που μάλιστα αναλαμβάνουν και κοινέ δραστηριότητες και κοινέ επιθεωρήσεις, για παράδειγμα σε παραμεθόριες περιοχές και είναι πολύ σημαντική βασική αρχή αυτή για τη σωστή λειτουργία. Το δίκτυο ΙΜΠΕΛ το οποίο ε, ασχολείται με τις επιθεωρήσεις των ΧΙΤΑ, υπάρχει εκεί σχετική τεκμηρίωση για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι επιθεωρήσεις. Δεύτερο, βέβαια, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, BAT, Best Available Techniques, αυτή βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης τώρα, τώρα και θα της δοθεί τελική μορφή νομίζω στις 12 Απριλίου όπου η Επιτροπή του άρθρου 75 θα συνέλθει για να ψηφίσει αυτό το έγγραφο των βέλτιστων πρακτικών για τον τομέα της ε, επεξεργασίας αποβλήτων. Εκεί, στο έγγραφο αυτό, περιλαμβάνονται οι σχετικές βέλτιστες πρακτικές και επίσης ε, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης που πάλι θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ένα τελικό σχέδιο ήδη από το κοινό κέντρο ερευνών της Ευήλης όπου μπορούν να βρεθούν, μπορεί να διαβάσουν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι, βέλτιστες πρακτικές για εταιρείε για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Το τρίτο ε, θέμα είναι τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Εδώ μπορούμε να δούμε τις σχετικές ελλείψεις σε ό,τι αφορά ανάκτηση, ή μάλλον ανάκτησης και διάθεσης, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς τέτοιες. Δεύτερον, όπου οι πολίτες αντιτίθενται με ισχυρό τρόπο απέναντι στην εγκατάσταση τέτοιων έργων στην περιοχή τους. Είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά not in my backyard, είναι όχι στη δική μου αυλή δηλαδή, και πολύ συχνά αντιδρούν οι τοπικοί πληθυσμοί. Τέλος, παράνομες μεταφορές και παράνομη απόθεση αποβλήτων ή απορριμμάτων, πάλι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς καταγγέλλοντες στις αναφορές τους. Ίσως με επιτρέπετε να προχωρήσω λίγο γρηγορότερα γιατί μου μένει μονάχα ένα λεπτό. Θα αφήσω τις συστάσεις αυτές ε, κατά μέρο, διότι κινούνται λίγο πολύ στην ίδια κατεύθυνση. Θα δείτε και τις βέλτιες πρακτικές για τούτο εδώ το θέμα που ανέφερα ε, προηγουμένως, το υπαριθμόν 3. Πάλι θα μπορέσετε να βρείτε στα ίδια έγγραφα guidance για επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματα κοινών ε, εγχειρημάτων που αναλαμβάνουν εθνικές αρχές και τοπικές αρχές και μπορείτε εκεί να βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά. Και θα ήθελα να πω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πλατφόρμες ε, ε, από τις οποίες μπορείτε να βρείτε στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες και συχνά στα site της αστυνομίας επίσης υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές σε μελέτη κάνουμε τέτοιες αναφορές. Τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι κάναμε αυτήν την ε, σχετική ανάλυση βάσει των τεσσάρων ε, αναφορών του 2017 ε, και μάλιστα αυτές βασίζονται σε ευρήματα του ήδη του 2011. Ελήφθησαν υπόψη λοιπόν όλα τα στοιχεία αυτά σε αυτήν την μελέτη την οποία σας παρουσιάσαμε σήμερα. Absolutely timely. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έγκαιρη η πληροφόρηση. Έρχεται δηλαδή την κατάλληλη στιγμή, γιατί εδώ έχουμε πολλά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων αυτή η διαχείριση αποβλήτων έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες. Θα ήθελα ιδιαίτερως να σας ευχαριστήσω κύριε Μπάουερ, γιατί δεν μακρηγορήσατε, είσαστε πολύ συγκεκριμένος και όπως ε, ε, είπατε η προηγούμενη ε, έρευνα του 2011 έχει πλέον επικαιροποιηθεί. Είναι αυτή που σας δείχνω και πραγματικά σας συστήνω την ανάγνωση αυτής της έκθεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Εδώ βασιζόμαστε, βλέπουμε εδώ πολλούς ε, Έλληνες βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες. Δε, δώστε τα και στους τοπικούς άρχοντες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ωραία. Πριν αρχίσουμε τις αναφορές, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, ε, Κομισιόν, τον κύριο Ντίας Δελκαστήγιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι από την Μονάδα Αποβλήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την τόσο συμπεριληπτική μελέτη. Ε, είναι δύσκολα πράγματα αυτή η διαχείριση των αποβλήτων και των ράδιο ενεργών ε, ε, αποβλήτων ήδη αντιμετωπίζεται από κατάλληλα κείμενα. Είδα τη διαφάνεια υπαριθμών 7, αυτό τον χάρτη ε, που λέει ήδη από το 11 ε, που συγκεντρώνονταν οι περισσότερες αναφορές. Ε, δεν εξεπλάγει γιατί είδα ότι η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι οι πρωταθλητές. Εκεί συγκεντρώνονται οι περισσότερες αναφορές και στις τρεις περιπτώσεις χωρών η Κομισιόν ανέλαβε νομική δράση και ανέφερε μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαδικασίες επί παραβάση. Αυτά, αυτές οι διαδικασίες αφορούν και τις τρεις χώρες ε, για ελληπείς διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων που ε, οδήγησαν τελικά σε παραβιάσεις. Η Ιταλία και η Ελλάδα πληρώνουν πάρα πολύ ε, βαριά πρόστιμα για την ύπαρξη χιτά. Η δε Ελλάδα έχασε την υπόθεση σχετικά με την μη ικανοποιητική διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Το λέω αυτό για να μην κατηγορήσει κανείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αδράνεια όσον αφορά τα θέματα αυτά. Επίσης να πω ότι έλαβα γνώση των διαφόρων ε, ελλείψεων που έχετε σημειώσει και των συστάσεων που κάνετε ε, και βεβαίως θα ε, μεταφερθούν αρμοδίως στους συναδέλφους της Επιτροπής. Το 2015 με το σχέδιο δράσης ε, της ε, κυκλικής ε, οικονομίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε τη διαχείριση των αποβλήτων σε διάφορα επίπεδα και κυρίως σε ε, πιο ε, φτωχά κράτη-μέλη και οι πιο πρόσφατα ε, κράτη-μέλη. όσον αφορά, ας πούμε, χώρους υγειονομικής ταφής που δεν καλύπτουν τους κανόνες ή ε, που δεν καλύπτουν επίσης κανόνες. Στην ουσία, θα πρέπει να ξεχάσουμε τις χωματερές ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια υψηλής ποιότητος ανακυκλωτική κοινωνία βάσει ε, των υψηλών στόχων που πρέπει να θετεθούν για κάθε κατηγορία αποβλήτων. Ωστόσο, θα πρέπει να καλυφθούν δύο κενά. Το ένα είναι ε, το κενό της νομικής εφαρμογής όσον αφορά ε, τα αρχεία διαχείρισης ε, αποβλήτων από τη μία και από την άλλη πλευρά τις ελλείψεις όσον αφορά τις επενδύσεις. Υπάρχει ε, σχετική, σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια. Η Κομισιόν μπορεί να βρει κάποιες πιο σκληρές λύσεις, ε, να πάει δηλαδή τα κρατημέλη στο δικαστήριο. Ε, ωστόσο, πριν από αυτό, προτιμάει η Κομισιόν να ξεκινήσει με την παροχή αρρωγής στα κράτη-μέλη, παροχή δηλαδή ε, τεχνικής αρρωγής κλπ. Δεύτερον, Παρέχουμε επίσης σεμινάρια συμμόρφωσης για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν να ε, ε, ε, εξυπηρετήσουν τους στόχους ε, έχουμε επίσης peer-to-peer -peer σεμινάρια, σεμιναρια ομοτήμων από τη μία χώρα στην άλλη. Ε, παρεπιπτόντως δε, να σας πω ότι είχαμε ε, και Ιρλανδούς αξιωματούχους που πήγαν στην Ρουμανία έτσι ώστε να τους ε, δείξουν πώς έλυσαν το σχετικό πρόβλημα ή σε την Ιρλανδία. Επίσης έχουμε μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης. Άρα εμείς κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπουν στο σωστό δρόμο. Μόνο και εφόσον όλες αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν τότε η Κομισιόν αναλαμβάνει ε, νομική ε, δράση και ξεκινάει διαδικασία επιβαραβάση. Ε, σε περιπτώσεις συστημικών αδυναμιών ε, και όταν δεν μπορούμε βέβαια να μελετήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κάθε μία ε, περίπτωση, διαλέγουμε αυτόν τον πιο αυστηρό τρόπο. Επομένως, επομένως σας λέγω ότι υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι, οι χώρες μέλη είναι αυτές οι οποίες είναι υπεύθυνε για να ενσωματώσουν στην νομοθεσία τους την σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ και που, μας, ε, ε, που έχετε δεσμευτεί και που ε, σπαταλάτε χρόνο και προσπάθεια για να είστε εδώ. Ας ελπίσουμε ότι ε, θα γίνουν τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα και όλοι θα υλοποιήσουν σωστά τα κείμενα και τις οδηγίες. Δυστυχώς για την ώρα, όπως θα δούμε και αργότερα με τη συζήτηση, αυτό δεν γίνεται. Η κυρία Μιράντα όμως, ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ε, εδώ δεν γίνεται αρκετή αναφορά στην περίπτωση της ε, Γαλλικίας. Υπάρχει ένα κενό κατά την άποψή μας, ε, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων στην Γαλλικία. Και μια και είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι το 2014 η πλατφόρμα της Γαλλικίας που αποτελείται από 35 οργανισμούς είχε υποβάλει μία αναφορά που ήταν πάρα πολύ, ε, α, πάρα πολύ απλή που έλεγε ότι θα πρέπει ε, να φτάσουμε στο zero waste όπως και άλλωστε το λέει και η ίδια η Κομισιόν και η μείωση απλώς ή η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων δεν μπορεί να αποτελέσει ε, λύση. Η καλυτερη διαχειριση των αποβλητων δεν μπορει να αποτελεσει λυση η αποτεφρωση ε, στην περίπτωση της Γαλλικίας ας πούμε αυτό που έγινε στην αρχή της εφαρμογής του προγραμματικού προγράμματος του 2010 ε, η αποτέφρωση ε, δεν ε, οδήγησε ούτε σε κομποστοποίηση ούτε ε, σε δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Επομένως δεν ήταν καλή, καλό σχέδιο διαχείρισης και μάλιστα αυτά τα σκουπίδια μεταφέροντο πάνω από 50 χιλιόμετρα μακριά και φυσικά στην ουσία μέσω της καύσης παρήγεται το διοξίδιο του άνθρακος και άλλου είδους ρηπαντές. Βεβαίως δεν είστε υπεύθυνος ε, για το σχέδιο αυτό, απλώς ε, εγώ δράτω με τις ευκαιρίας ε, για να πω ότι υπάρχει αυτή η αναφορά από την ομάδα Βέρδε Σάλε, που είναι αυτή η πλατφόρμα που σας έλεγα και εδώ νομίζω ότι είναι... Και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ε, ναι, ναι, στους, στους συντονιστές θα πρέπει να το κάνετε και όχι στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Ελάτε σε επαφή με τον συντονιστή σας έτσι ώστε να προωθήσει ξανά το θέμα. Η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε εδώ ε, δύο αναφορές μεταξύ των ε, πολλών αναφορών που οδήγησαν σε αυτήν την ε, έκθεση αφορούν την Καλαβρία. Τέσσερα χρόνια πριν, η πρώτη φορά δηλαδή, ταυτόχρονα με την πρώτη φορά που μίλησα για το θέμα αυτό, η Ιταλία ε, κατεδικάζεται από την, ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της ε, κακής διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. 58 εκατομμύρια ευρώ με τη μία, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά, πολλοί χώροι που δεν είναι κανονικοί χώροι υγειονομικής είναι στην ουσία χώροι ελεύθερης αναπόθεσης, χωματερές απλές. Ε, ακόμα και όσον αφορά ε, τα ε, νερά της αποχέτευσης, ούτε αυτά μπόρεσαν, τα υγρά δηλαδή απόβλητα, ούτε αυτά μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν σωστά και βάσει της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όσον αφορά λοιπόν και την μόλυνση των υδάτων και του υπεδάφους και όσον αφορά το περιβάλλον, οι επιπτώσεις είναι σοβαρές. Ας μην αναφερθούμε δε επιπτώσεις όσον αφορά ε, την υγεία. Ε, επίσης, ε, πολλές επικρίσεις έχουν καταφερθεί εναντίον του πρόσφατου προγράμματος για την ανακύκλωση και για τη διαχείριση των αποβλήτων. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, δεν προωθείται η επαναχρησιμοποίηση δευτερογενώς των ισχύων και επίσης χρησιμοποιείται η αποτέφρωση για να καούν τα δευτερογενή στερεά απόβλητα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιφέρειες ε, στις ε, οποίες ε, τα ε, η περιφέρεια βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή όσον αφορά τις πράξεις της και τις αποφάσεις της. Ε, οι κοινότητες λοιπόν ε, εξανίστανται γιατί πλέον δεν έχουν εμπιστοσύνη στους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς άρχοντες. Υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις όπου εκτός από την πρώτη χωματερή υπάρχει και μία δεύτερη στην οποία θα εναποτίθενται ε, τα αποτελέσματα ας πούμε, τα αυτά που, ε, ε, η παραγωγή που προκύπτει μετά από την κομποστοποίηση ή από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν έχουμε με κανένα τρόπο το zero waste και δεν καλύπτεται με κανένα τρόπο η οδηγία πλαίσιο. Επίσης, ως εισηγήτρια για την έκθεση που αφορά ε, την ε, οδηγία ε, για την πρόληψη και όσον αφορά και την περιβαλλοντική ευθύνη, θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο μια σειράς παρεμβάσεων προληπτικών, έτσι ώστε να κινητροδοτηθούν οι κάτοικοι, οι πολίτες για να ανακυκλώνουν και επίσης να ευαισθητοποιηθούν για την αρχή και να την εφαρμόσουν ότι ο πληρώνει. Όσον αφορά τώρα την αναφορά για τα ραδιοενεργά απόβλητα, γιατί και αυτή αφορά την Καλαβρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη ε, την έκβαση των ε, ε, κοινοβουλευτικών ερευνών και μελετών για το θέμα αυτό. Η σχετική διερευνητική επιτροπή σε συνεργασία με τις αρχές της Ιταλίας και τις μυστικές υπηρεσίες έχουν καταλήξει καταλήξει ότι υπάρχει παράνομη δραστηριότητα όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο στην Ιταλία ε, έχει πλέον μπει σε αυτήν την ε, ε, διαδικασία. Επίσης ε, στην περιοχή της Αμαντέα έχουμε περίπου στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων και του οργανωμένου εγκλήματος περίπου το 90% της ανακύκλωσης. Ε, όχι αυτό δεν συμβαίνει μονάχα στην Καλαβρία αλλά και σε άλλες ε, περιοχές κυρίως της Μεσημβρίας της Ιταλίας. Επομένως χρειάζεται σωστή εφαρμογή των κειμένων που αφορούν την προστασία των υδάτων και του υπεδάφους. Ε, χρειάζεται προστασία όχι μονάχα του περιβάλλοντος αλλά οπωσδήποτε και της υγείας και φυσικά διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, ε, νομίζω πως αυτά που μας είπατε δεν είχαν σχέση με αυτή τη μελέτη. Αργότερα θα μπούμε στην ουσία των διαφορών αναφορών. Αν συνεχίσουμε έτσι, ο καθένας να παίρνει το λόγο και να ξεχνάει να το δώσει πίσω, θα ξεφύγουμε από τον έλεγχο. Κύριε Μαριά, ε, εσείς να είστε πολύ πολύ σύντομος. Ε, πράγματι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην ε, Ευρώπη είναι σίγουρο ότι αποτελεί ένα κείμενο που πρέπει να παρακολουθήσουν με προσοχή, όπως είπατε, όλες οι αρχές, ιδίω οι ελληνικές αρχές, μια και θα έχουμε τις υποθέσεις αμέσως μετά. Εγώ θέλω να προβληματιστούμε λίγο για το τι μπορεί να γίνει παραπέρα γενικώ. Διότι έρχεται μία αναφορά και καταγγέλει μία παραβίαση της κοινοτική νομοθεσίας. Πρακτικά τι συμβαίνει. Θα λάβει δράση η Κομισιόν, αλλά πολλές φορές οι κάτοικοι απαιτούν αμέσως να ληφθούν μέτρα. Αμέσως να σταματήσει η παραβίαση των όρων των περιβαλλοντικών. Διότι πολλές, ιδίως τοπικές κυβερνήσεις, δημιουργούν ε, φέτα κομπλή. Δηλαδή δημιουργούν τετελεσμένα γεγονότα. Οπότε όταν εμείς έρθουμε αργότερα, ήδη υπάρχει η χωματερή, ήδη λειτουργεί και τι θα γίνει. Θα πάει η Κομισιόν το κράτος στο δικαστήριο, θα περάσουν δύο-τρία χρόνια και μετά αν δεν συμφωνήσει το κράτος θα ξαναπάει η Κομισιόν το κράτος στο δικαστήριο και θα του επιβληθεί ένα πρόστιμο. Στην πράξη όμως επί 6-7 χρόνια θα λειτουργούν παράνομα οι χωματερές, θα παραβιάζει την νομοθεσία και κυρίως θα υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε το άμεσο αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε πολλές φορές εδώ και τώρα. Και αυτό είναι το σημείο που νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε. Πώς η Επιτροπή μας θα μπορεί να αποκτήσει αρμοδιότητες ή να κάνει τέτοιες προτάσεις, ούτω ώστε να σταματούν άμεσα οι βλαπτικές ενέργειες. Διότι αν είναι να γίνει σήμερα μια αναφορά και τελικά να σταματήσει ένα έργο μετά από 6-7 χρόνια. Αν σταματήσει, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που επιθυμούμε εμείς, που επιθυμούν οι πολίτες. Επομένως, σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να προβληματιστούμε, να δούμε και η Κομισιόν πώς βλέπει το θέμα, ούτω ώστε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα. Και στη βάση αυτή πιστεύω ότι έχουμε πετύχει σαν Επιτροπή δύο στοιχεία. Και θα τα πω αυτά γιατί μετά μπορούμε να περάσουμε στις υποθέσεις ελληνικέ. Πρώτον, ότι έχουμε ενεργοποιήσει την διαδικασία έκτακτων αναφορών. Δηλαδή όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μπορούμε να ζητήσουμε εκτάκτως άμεσα σαν κατεπήγον να συζητηθεί μία αναφορά μέσα σε δύο, τρεις, τέσσερις μήνες από τότε που κατατίθεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους τους πολίτες και για το αποτέλεσμα. Και δεύτερον, είχαμε πάρει μια πρόσφατη απόφαση που αφορούσε την Ιταλία όπου ως Επιτροπή καλέσαμε τις τοπικές αρχές και τις εθνικές αρχές να σταματήσουν άμεσα κάθε ενέργεια και δράση σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορούσε νομίζω μία λίμνη σε μια περιοχή της Ιταλίας. Και αυτό ήταν κατάκτησή μας. Αυτή λοιπόν η πρόταση η οποία από ό,τι έμαθα επηρέασε, σταμάτησε τις λειτουργίες που ήθελε να επιβάλλει εκεί ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη συνολικά και ιδίω στι επόμενε υποθέσει που θα συζητήσουμε κύριε Πρόεδρε για να προλάβουμε τη ζημία στην υγεία και στο περιβάλλον και να μην έρθουμε μετά από 7 χρόνια σε μια νέα μελέτη για να λέμε απλά ότι παραβιάστηκε το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ως συμπέρασμα της μελέτης για το πώς με δραστικά μέτρα θα παρεμβαίνουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε δίκιο, οπωσδήποτε. Κύριε Χούντι, Χοντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρήκα ενδιαφέρουσα τη μελέτη. Την άκουσα. Τυχερός είμαι. Ήρθα για τις μετέπειτα αναφορές σε ελληνικά θέματα. Όπως επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και η τοποθέτηση του εκπροσώπου της Κομισιόν. Της Κομισιόν. Αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που εν ολίγης έθεσε πρώτων ευθυνών κυρίως τα κράτη. Έχοντας το πλεονέκτημα, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, να είμαι μέλος της Επιτροπής Αναφορών το προηγούμενο διάστημα. Να είμαι ε, ευρωβουλευτής από την Ελλάδα που ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Αλλά και για τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Να είμαι για ένα διάστημα υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελλάδας όπου χειριζόμαστε και τα θέματα των, ε, της Κομισιόν επί παραβάση Έχω παρακολουθήσει λοιπόν όλη την αλυσίδα των γεγονότων και έχω ίσως μια διαφορετική γνώμη ποιες είναι οι και πού πρέπει να, τι άλλο πρέπει να κάνω. Δύο κουβέντες όμως γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η μελέτη δεν μπορούσε να πάει παραπέρα από τα στατιστικά στοιχεία που έτσι κι αλλιώς είχαμε στην Επιτροπή Αναφορών το προηγούμενο διάστημα. Που λένε ότι προβλήματα στη διαχείριση απορριμμάτων έχουμε κυρίως στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία είχαμε το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το λόγο έγινε και η σχετική επίσκεψη και γι' αυτό το λόγο υπαγορεύτηκε αυτή η μελέτη. Ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντήσει η μελέτη και είναι αντικείμενο πολιτική απαντήση, γιατί. Γιατί σε αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, έχουμε παραβιάσεις, έχουμε εμβαλωματικές λύσεις. Παλαιότερα, καμιά φορά και στη μελέτη, εξηγείται ως πολιτισμική υστέρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει περιβαλλοντική συνείδηση όσο αφορά το ζήτημα αυτό. Στη συνέχεια όμως αποκαλύφθηκε ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί μαφιόζικου και το μαφιόζικο το λέω με αφορμή την Ιταλία και τα φαινόμενα δια, μαφιόζικης διαχείρισης των κοινοτικών πόρων όσο αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των έργων δηλαδή με, με σκοπιμότητες να το πω έτσι και όχι για να βγει αυτό, κατά αυτό το έργο και δεύτερο μια αδράνεια της Κομισιόν να προλάβει το κακό. Πού υπογραμμίζω την αδράνεια της Κομισιόν για να προλάβει το κακό. Στο γεγονός ότι στις περισσότερες από τις ε, ε, μελέτες περιβαλλοντικών επιτόσεων των προβληματικών κατά τα άλλα χιτά, δεν έχει ενσωματωθεί η νεότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν έχει ενσωματωθεί. Η Κομισιόν όμως δεν θυμίζει ότι Ακόμα και όταν δεν έχει ενσωματώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία την πιο προθυμένη, πρέπει να την παίρνει υπόψη στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με συνέπεια να έχουμε αυτέ τι αχρονίε. Αυτέ είναι ορισμένε παρατηρήσει, τα υπόλοιπα τα συγκεκριμένα. Έχει, έχει ενδιαφέρον όμω αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τα γενικά, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα τα πούμε και στο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Can, can we now... Actually... Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στις αναφορές γιατί περιμένουν οι αναφέροντες εντός της αιθούσης. Βεβαίως, οι στις πρακτικές τονίστηκαν από τον κύριο Νόϊμπάγερ, αλλά και από την Επιτροπή ότι όντως αυτό γίνεται. Η Επιτροπή μπορεί να δράσει όταν υπάρχουν συστηματικά αδυναμίες ή παραβιάσεις των οδηγιών. Και πάλι σας παρακαλώ να σημειώσετε τη μελέτη με το χάρτη όπου μπορείτε να δείτε πως υπάρχουν ορισμένες χώρες που δεν επηρεάζονται καθόλου. Και τώρα μπορούμε να αντιστρέψουμε και το ερώτημα του κύριου Χουντή και να πούμε τι κάναν σωστά αυτές οι χώρες και ίσως να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα. Θα ήταν αυτός ένας έξυπνος τρόπος. Ίσως να είναι αυτή η συμβολή μας στην ε, ε, τοπική και ε, αυτοδιοίκηση. Ε, δείτε και αντιγράψτε τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είμαι βεβαία. Για την δημιουργία χωματερής στο Καρβουνάρι. Ο αναφερόμενος είναι εδώ είναι ο κ. Παπαδόπουλος και με χαρά θα σας δώσω τον λόγο για 5 λεπτά maximum. Παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτές, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών, έχουν περάσει 10 χρόνια από την ημέρα που καταθέσαμε την κοινή μας αναφορά για τους χιτά καρβουναρίου και λευκίμης. Σήμερα δεν, θα, δεν σας έφερα ούτε PowerPoint, ούτε στοιχεία, ούτε φωτογραφίες. Ούτως ή άλλως η Κομισιόν παλιότερα σε μια επιστολή είχε αμφισβητήσει τα στοιχεία μου και τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Σας υπόσχομαι ότι θα μιλήσω λιγότερο από πέντε λεπτά, θέλω όμως να με ακούσετε μέχρι το τέλος. Σε ό,τι αφορά το Χιτά Λευκήμης, όπως γνωρίζετε, το έργο ευτυχώς δεν λειτουργεί. Και κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη στεναρή αντίσταση των καντίκων που δεν, σχέση, που δεν έχει σχέση με το περίφημο νύμπι και την άγρια καταστολή που σας υπενθυμίζω και κάθε φορά που θα έρχομαι εδώ θα το υπενθυμίζω στήχησε τη ζωή σε μια μητέρα δύο παιδιών, την Μαρία Κουλούρη. Ο δεύτερος και ο κυριότερος είναι καθαρά θέμα συνείδησης. Κανένας πολιτικός, είτε είναι δήμαρχος είτε περιφερειάρχης, δεν έχει καθαρή την συνείδησή του για να ξεκινήσει τον παράλογο, παράνομο και θανατηφόρο αυτό έργο. Κανένας. Υπάρχει όμως και ένας υπόγειος σχεδιασμός, σαν αυτούς που βγαίνουν από τους βόθρους, που θέλει αυτό το καλοκαίρι να φτάσουν στο αδιέξοδο με δόλο μέσω τουριστικής περίοδου, ούτως ώστε να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα της προστασίας της δημόσιας υγείας για να ξεκινήσουν τη λειτουργία του χιτά Σε ό,τι αφορά τον χιτά Καρβουναρίου, θα ήθελα ειλικρινά να σας ζητήσω μία μεγάλη συγνώμη για όλη αυτήν την ταλαιπωρία. Τελικά παραδέχομαι δημοσίως ότι είχα λάθος. Είχα κάνει λάθος υπολογισμούς από την πρώτη μέρα, πριν 10 χρόνια, όταν είχα εξ αρχής υποτιμήσει έναν σημαντικότατο παράγοντα. Εξηγούμε αν και μετά από 10 χρόνια η τρύπα του χιτά έγινε βουνός πλέον, όπως όμως μας διαβεβαιώνουν όλα τα στοιχεία, από τον χιτά του καρβουναρίου δεν χύνονται άλλα στραγγίσματα, παρά μόνο ένα πεντακάθαρο και κρυστάλλινο υγρό παρόμοιο με το νερό των παγετώνων. Δεύτερον, η ανακύκλωση στον Δήμο Σουλίου, που ήταν ένας όρος για να λειτουργήσει οχητά, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια Επίρου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Και δεν έχουμε ούτε 10, ούτε 20% ποσοστά ανακύκλωσης, αλλά κρατηθείτε γερά στα έδρανα, φτάσαμε στο 120%. Πετύχαμε το απίστευτο, το αδιανόητο της νοητικής ανακύκλωσης. Η υπηρώτησα νοικοκυρά πλέον, μόνο που σκέφτεται το σκουπίδι, αυτό ανακυκλώνεται από μόνο του. Τώρα πώς το πετύχαμε η ταγή των Δήμων μας και της περιφέρειας με μια γυροβολιά στα πανηγύρια, δύο ευχέλια και ένα τρισάγιο έκαναν το θαύμα. Και μην νομίζετε πως σας κοροϊδεύω, γιατί μακριά από μένα μια τέτοια σκέψη. Αφού το θαύμα αυτό έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα και επικυρωθεί από το πλέον αρμόδιο όργανο, την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν. Οπότε ειλικρινά και για μια τελευταία φορά για το θέμα του Καρβουναρίου, σας ζητώ συγγνώμη που δεν πρόβλεψα, όπως η Κομισιόν, τις θαυματουργικές ικανότητες των ταγών των Δήμων και της Περιφέρειας Υπήρου. Τα ίδια ισχύουν και για το χιτά ελληνικού. Είμαι σίγουρος πως οι ίδιες ικανότητες θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε στην Ήπειρο και το θαύμα των πετρεαλικών εξορίξεων. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, now I turn to... Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα στρέφομαι στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Κουνινιώτη. Merci, Madame la Présidente. Euh, je vais vous répondre. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας απαντήσω όσον αφορά τον χιτά καρβοναρίου. Θα εστιάσω σε δύο σημεία. Το πρώτο όσον αφορά την ίδια τη λειτουργία του χιτά. Αυτή η υπόθεση, αυτή η αναφορά ξεκίνησε το 2008 λόγω της κακής λειτουργίας ε, του ΧΙΤΑ. Η Κομισιόν προέβησε δράση. Δυστυχώς χρειάστηκε να κινήσει η διαδικασία κατά παράβαση και όπως σας ενημερώσαμε στη τελευταία μας ανακοίνωση προς την Επιτροπή σας το 2015 φαινόταν ότι επί τη βάση των πολυάριθμων επιθεωρήσεων που διενέργησαν οι τοπικές αρχές η λειτουργία, μάλλον τα προβλήματα της λειτουργίας είχαν ρυθμιστεί και η λειτουργία ήταν αποδεκτή αν όχι και καλύτερη. Επί τη βάση αυτή, το 2015 κλείσαμε την ε, διαδικασία κατά παράβαση σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι χαίρομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να διαβάσω την νέα επιστολή που στείλαμε στην Επιτροπή σας στις 15 Μαρτίου με από την ε, περιφέρεια Επίρου που επιβεβαιώνει από το 2013 μέχρι το 2018 η οχητά συνεχίζει να λειτουργεί κατάλληλα. Δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα σε ελεγκτικό κλιμάκιο, άρα δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε αυτήν την ετοιμιγορία. Τώρα, τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Δεν θα επεκταθώ ιδιαίτερα εδώ, γιατί ε, υπάρχει ο στόχος ε, του 2030, να μειωθ, μέχρι το 2030 να μειωθούν ε, η χιτά και άρα και η ρήψη αποβλήτων, απορριμμάτων, αλλά μέχρι στιγμής δεν απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία να υπάρχουν χιτά. Είναι η χειρότερη επιλογή στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά δεν απαγορεύεται. Από τη στιγμή που λειτουργεί η χωματερή σωστά. Ε, και επίση στο ίδιο σημείωμα οι περιφερειακέ αρχέ λένε ότι για να βελτιωθεί η κατάσταση και ακριβώς να προχωρήσουμε προ μια καλύτερη ποιότητα, το νέο περιφερειακό σχέδιο της Περιφέρειας Υπήρου προβλέπει τη δημιουργία ε, μιας μονάδας ε, επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων και μόνο ένα κομμάτι των ήδη κατεργασμένων αποβλήτων θα πηγαίνουν στο χιτά καρβουναρίου. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο θα τροποποιηθεί, δεν θα απορροφά απορρίμματα, αλλά υπολείμματα. Άρα, λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην είναι ιδανική λύση, αλλά είναι μια λύση που οφείλουμε να δεχτούμε γιατί δεν απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία. Και, όπως οι συνάδελφοι, Έχουμε αναφέρει μέσω των διαφόρων οργάνων και διαδικασιών ότι οφείλουμε να βοηθάμε την Ελλάδα και όλα τα κράτη-μέλη, κυρίως την Ελλάδα που έχει πολλά προβλήματα στη διαχείριση απορριμμάτων, ώστε να συνεχίζεται η διαχείριση αυτών σε όλα στο ΣΧΙΤΑ και να ελπίζουμε ότι ε, η ΧΙΤΑ θα είναι σε λίγο θέμα του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα... Το λόγο μπορούν να πάρει η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας και, και με το εκπρόσωπο του κύριο Μαντζάρη. At the very back of the room, please the floor. Α, εκεί είστε πίσω πίσω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Καταρχά ε, ευχαριστώ για την ε, παρουσία. Εκ μέρους βρίσκομαι εδώ από την μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπώντας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ε, επιτρέψτε μου ε, να θέσω υπόψη της Επιτροπής ορισμένα πρόσφατα στοιχεία ε, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και συγκεκριμένα τους χώρους υγειονομικής ταφής που σχετίζονται με τις σημερινές αναφορές, όπως μας έχουν διαβεβαστεί από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ε, αν επιθυμείτε μπορώ να αναφερθώ μόνο στο συγκεκριμένο ή και σε όλες τις υποθέσεις που έχουμε συνολικά. Ε, είναι στοιχεία τεχνικής φύσης κυρίως, ε, τα οποία αν θέλετε μπορείτε να σας προβάλλω, τα έχω ήδη αποστείλει και στην γραμματεία. Ε, ως, ως προς την... We would be very grateful for, for... Θα ήμασταν ευγνώμονες για οποιοδήποτε είδος πληροφορίες μπορείτε να μας δώσετε. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο μπορούν να πάρουν οι συνάδελφοι. Η κυρία Κούνεβα πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με συγχωρείτε. Τελείωσε η... ο εκπρόσωπος της ε, Ελλάδας. Έτσι νόμισα. Ναι, Τελειώσατε. Αν επιθυμείτε να σας διαβάσω τα αναλυτικά τεχνικά στοιχεία. Γιατί και κάτι άλλο. Ε, you want to give Θέλετε να μας δώσετε παραπάνω πληροφορίες. Θέλετε να μας δώσετε ότι έχετε παραπάνω. Εγώ νόμιζα ότι κατάλαβα πως θα μας δώσετε τεχνικές πληροφορίες γραπτός. Πράγμα το οποίο θα εκτιμούσαμε. Θα σας περιγράψω τα στοιχεία που έχω ενώπιον μου. Πρόκειται για το περιεχόμενο του, σχεδίου, του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για την Ήπειρο και την Αττική. Μπορώ να σας τα διαβάσω. Επειδή έχουμε χρονικούς περιορισμούς, θα το εκτιμούσαμε να μας τα στείλετε γραπτός και μετά θα το διανύμουμε στους συναδέλφους εμείς. Thank you very much. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και ο λόγο είναι τώρα για την κυρία Κούνεβα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το προτιμούσα να μιλήσω τελευταία, να ακούσω προ τους συναδέλφου, παρακαλώ. Τώρα ο λόγο είναι η κυρία, κυρία Μάρια. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, καταρχά δεν είναι παρουσία αυτή του ελληνικού Υπουργείου αρμόδιο για τα θέματα που συζητάμε, δηλαδή ε, τα περιβαλλοντικά. Δεν είναι μορφή βεβαίω προ τον εκπρόσωπο τη ΜΕΑ, προ Θεού. Όμω, καταρχά, εδώ έχουμε τέσσερι σοβαρέ υποθέσει. Η χωματερή της χιλής, της, <laughs> της φυλής πραγματικά ε, απασχολεί όλη την πρωτεύουσα και οι υπόλοιπε υποθέσεις είναι πολύ σοβαρές όπως αυτή στο γραμματικό και θα περίμενα να είχαμε εδώ ένα εκπρόσωπο από το αρμόδιο Υπουργείο για να τοποθετηθεί τι θα γίνει επί του πρακτέου. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να λυθούν και άλλα που ίσως πάνε λίγο αργότερα. Αλλά θέλουμε μια υπεύθυνη πολιτική απάντηση για τη διαχείριση. Δεύτερον, δεν βλέπω εδώ την περιφέρεια. Υπάρχει ας πούμε η περιφέρεια, η αρμόδια. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν υπάρχουν λοιπόν σοβαρές παραλήψεις κατά την άποψή μου σε επίπεδο διοίκησης για το χειρισμό των θεμάτων. Τρίτον, έχουμε την υπόθεση ε, στη Λευκήμη. Πρόκειται για παλιά υπόθεση, έχει όλα τα προβλήματα που ανέφερα και προηγουμένως σε σχέση με το πώς γίνεται ο χειρισμός των υποθέσεων. Μην ξεχνούμε ότι υπήρξε άγρια καταστολή κατά των κατοίκων προκειμένου να μην αντισταθούν στην λειτουργία της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου χιτά στη Λευκήμη. Είχαμε, όπως αναφέρθηκε και από τον αναφέροντα, την, ε, το θάνατο της Μαρίας Κουλούρη, η οποία χτυπήθηκε κυριολεκτικά ε, δάρθηκε από τα ΜΑΤ και δυστυχώς πέθανε και από εκεί και πέρα έχουμε ένα ερώτημα τι θα γίνει το καλοκαίρι. Εγώ θα περίμενα να έρθει εδώ η αυτοδιοίκηση να μας πει τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μήπως από την πίσω πόρτα λειτουργήσει το συγκεκριμένο χιτά. Μήπως πει μαζευτήκαν πολλά σκουπίδια το καλοκαίρι στην Κέρκυρα θα έχει και πολύ τουρισμό και μακάρι να έχει πολύ τουρισμό και τελικά αρχίζει και λειτουργεί. Και νομίζω ο Περιφερειάρχης Επτανήσων έχει δείξει μία σοβαρότητα στα θέματα που χειρίζεται και γύρω από τη Φραπόρτ και θα περίμενα να έχουμε μια παρουσία. Για την άλλη υπόθεση, λέει η Κομισιόν, δεν έχω πάει επί τόπου να ελέγξω τα στοιχεία. Εμείς δηλαδή πώς θα τοποθετηθούμε ως Επιτροπή. Ισχύουν αυτά τα οποία καταγγέλει ο αναφέρον. Ισχύουν αυτά που μας λέει η Περιφέρεια Υπήρου. Δεν ήρθε καν εδώ η περιφέρεια Υπήρου για να παρουσιαστεί. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου πραγματικά κάνει μια σοβαρή δουλειά σε άλλα θέματα. Όπως και στο θέμα της ΦΕΤΑ και σε άλλα ζητήματα. Αλλά εγώ θα περίμενα εδώ να έρθει να τοποθετηθεί. Λέει η Κομισιόν, δεν έχω υπηρεσίε να πάω να ελέγξω. Και εμεί εδώ τι θα κάνουμε, τι θα ακούσουμε, ποιον θα ακούσουμε, ποιον θα πιστέψουμε. Είναι έτσι τα στοιχεία. Και μου κάνει εντύπωση γιατί η Κομισιόν δεν φρόντισε να ελέγξει πραγματικά αν είναι έτσι τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι για να είμαστε εντάξει θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές οι συγκεκριμένες. Δεν έχω εμπιστοσύνη έτσι όπως βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται και με προβληματίζει η απουσία της ελληνικής κυβέρνησης η οποία πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δεν μας λέει τίποτα. Και αφήνει σε εμά να λύσουμε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν να παραμείνουν ανοιχτές οι υποθέσεις να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ελέγξει παραπέρα τα στοιχεία στην δεύτερη υπόθεση και να επισημάνουμε στις περιφερειακές αρχές για τη Λευκή ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό πρέπει να είναι το πλαίσιο των αποφάσεων που θα πάρουμε κυρία Πρόεδρε. Thank you very much, Mrs. Mr. Marias. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαριά. Ο κύριος Χουντής. Θα είμαι σύντομος ε, το θέμα το γνωρίζω τα δύο τουλάχιστον, Λευκήμη και Καρβουνάρη. Ήταν από τα που επισκέφθηκε η Επιτροπή Αναφορών το Σεπτέμβριο του 2013. Επομένως έχω καθαρή γνώση του ζητήματος. Ισχύουν οι αιτιάσει της ε, αναφοράς και πιστεύω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή. Προσθέτω, η Λευκήμη είναι λάθος χωροθέτηση, το είδαμε, η διεισόμαση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να λειτουργήσει. Όμως κυρία Πρόεδρε, η πίεση που θα ασκηθεί λόγω καλοκαιρινής περίοδου μπορεί να οδηγήσει σε μια κατοικονομία χρήση μιας ακατάλληλης, πλήρως, πλήρως ακατάλληλης ε, χωροθέτησης ε, ε, λειτουργίας της Λευκήμης. Δεύτερο, όσο αφορά το καρβουνάρι, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία δεν ήταν επαρκής, δεν ήταν ικανοποιητική, δεν ήταν σωστή. Και το ερώτημα το δικό μου, και επομένως να μείνει ανοιχτή, με, να ζητήσουμε περισσότερες διευκρινήσεις και από την ε, ελληνική κυβέρνηση, από τον εκπρόσωπο της ΜΕΑ, τι από τον περιφερειακό σχεδιασμό που ε, επικαλέστηκε τον πείθη ότι θα είμαστε εντάξει. Δεν θέλω να προσθέσω περισσότερα σχετικά με τους περιφερειακούς σχεδιασμούς, πολύ περισσότερο για αυτά τα θέματα και αυτή την περίοδο. Γιατί γίνονται κάτω από το κράτος άλλων καταστάσεων. Επομένως, ανοιχτή, ζητώντας περισσότερα στοιχεία και από την ελληνική κυβέρνηση και από την περιφέρεια, για να μπορεί να αποφαρθεί κανείς πιο ουσιαστικά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mrs. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, ακριβώ επειδή οι προηγούμενοι συνάδελφοι αναφερθήκαν αναλυτικά πάνω στο θέμα, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπαν. Θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό το γεγονό ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, εκτό από την αναφορά έτσι όπω την έχουμε διαβάσει, και φυσικά θα πρέπει η Κομισιόν να, να, να, να φτιάξει ένα κλιμάκιο, να μπορέσει να κάνει μια επιτόπια έρευνα και να παραμείνει η υπόθεση ανοιχτή. Αυτό. Okay, Τώρα, κυρία Κούνεβα, θα είστε η τελευταία ομιλήτρια. Είσαι σύμφωνα με τους συνάδελφους που τοποθετήθηκαν πολύ καλά ε, στο θέμα αυτό και θα ήταν πολύ καλά πριν το καλοκαίρι αν καταφέρουμε να κάνουμε τη συζήτηση ξανά εδώ με όλες τις οργανώσεις και υπεύθυνοι ε, υπεύθυνες περιφερειάρχες ε, της Ελλάδας ε, με τις αναφορές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε να πάρετε για ένα λεπτό ακόμα το λόγο για να μας πείτε μετά πώς ακούσετε ποια είναι η θέση σας. Των Ευρωβουλευτών, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα είχαμε προβλέψει πριν λειτουργήσει ο ΧΙΤΑ. Και αυτό που μας έλεγε η Κομισιόν τότε είναι ας λειτουργήσει πρώτα και μετά θα δούμε. Και ειλικρινά, ενώ εμείς καταθέμε ακράταντα στοιχεία, ακόμα πήγαμε με καθηγητές πανεπιστημίων πριν ξεκινήσει καν το έργο και βγάλαμε μελέτες που δείχνουν και την επικινδυνότητα σήμερα του έργου, η Κομισιόν ποτέ δεν μας στήριξε. Φτάσαν σε σημείο να μου πούν ότι η αρχή της πρόληψης, le principe de précaution, είναι απλά ένα προήμιο της διρεκτίβας και δεν είναι μέσα στην διρεκτίβα. Αυτό θέλω να πω γιατί είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος, εγώ, όχι μόνο εγώ, όλοι οι κάτοικοι, από την στάση της Κομισιόν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τα στοιχεία που σας θέτει η περιφέρεια, ο Χιτά Καρβουναρίου έχει γίνει πλέον ένα βουνό και ανοίγουν δεύτερο κύτταρο, όταν το λεγόμενο κύτταρο ήταν να λειτουργήσει για 20 χρόνια, έχουν περάσει 10 χρόνια, έχει γίνει βουνό και δίπλα τώρα αδειοδοτούν ένα δεύτερο κύτταρο. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει πώς οι μελέτες ήταν σοβαρές. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Now, ε, ε, Τώρα, όπως ε, γνωρίζετε, έχουμε λάβει επιστολές από την περιφέρεια Υπήρου και μάλιστα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό που λένε στην επιστολή τους είναι ότι δεν τους έχουν αναφερθεί προβλήματα σχετικά με την χρήση της, του χιτά. Και σε χθεσινή επιστολή η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αναφέρεται σε αποφάσεις για την κατασκευή της χωματερής, της χωματερής Λευκήμης. Όπως γνωρίζετε, η παρούσα Επιτροπή Αναφορών, πριν αναλάβω εγώ την Προεδρία στην προηγούμενη θητεία, το 2013 πιο συγκεκριμένα, είχαν πάει σε επιτόπου επίσκεψη και στο Καρβουνάρι και στην Κέρκυρα. Τα εξέτασαν αυτά, έκαναν συστάσεις και θα ήθελα να στραφώ τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσω να εξετάσει την τρέχουσα κατάσταση υπό το φως των πιο πρόσφατων πληροφοριών που μας έχουν δοθεί. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, όπως ζήτησαν και οι συνάδελφοί μου, θα, ζητή, θα κρατήσουμε τις ε, αναφορές ανοιχτές. Η γραμματεία θα μείνει σε στενή επαφή και συνεργασία μαζί σας και θα δούμε τα όσα επιτεύχθηκαν πρόσφατα. Και βεβαίω και τι δεν έχει επιτευχθεί απολύτω. Για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Νομίζω θα χρειαστούμε τις σχετικές πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτός. Δηλαδή μια ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις. Εκπλήσωμε κάπως που κανείς δεν αναφέρεται στην ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου καθώς και στην ε, σύμβαση άρχους γιατί άνθρωποι ζουν κοντά στους χιτά αυτούς και έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν εμπλακεί με κατάλληλο τρόπο στην διαδικασία. Θα έπρεπε να έχει γίνει η δημόσια διαβούλευση, ο κόσμος, να, το κοινό δηλαδή, να, έχει, να του έχει ζητηθεί η γνώμη του και αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή Αναφορών είναι να στείλουμε επιστολές και στις αρχές, τονίζοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται εν κρυπτό. Οι πολίτες πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι και ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να γίνονται τα πράγματα. Και βέβαια, χρειάζεται να αναφερθούμε και, και θα ήθελα και εγώ μάλιστα να αναφερθούμε και να τους διαβιβάσουμε την πρόσφατη μελέτη, να τη στείλουμε δηλαδή στις περιφερειακές αρχές και να τους παρακαλέσουμε να την εξετάσουν, να τη διαβάσουν και να συμμορφωθούν με αυτήν. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, συμφωνείτε. Νομίζω ότι είναι σωστός αυτός ο τρόπος και έτσι τουλάχιστον έχουμε αναλάβει κάποια δράση και ε, με την ελπίδα ότι θα λάβουν υπόψη τους αυτές τις παρατηρήσεις μας. Ωραία λοιπόν, έχει καλώς. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη αναφορά η 1653 εξ ονόματος 360 κατοίκων της πληγής σας περιοχής σχετικά με έκθυμες παρατυπίες στην διαχείριση της χωματερής ελληνικού Ιωαννίνων πάλι στην περιοχή της Υπήρου στην Ελλάδα. Κύριε Πρέντα, νομίζω ζητήσατε το λόγο πριν να προχωρήσουμε στη συζήτηση επόμενης αναφοράς. Αργότερα λοιπόν. Α, είναι το ίδιο πρόσωπο, ναι, ο ίδιος αναφερόμενος και λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε από τον κύριο Παπαδόπουλο να είναι συντομότατος, να μας εξηγήσει ποια είναι η πιο πρόσφατη ενημέρωση που μπορεί να μας δώσει. Με καλύπτουν τα όσα είπα προηγουμένως, δεν έχω τίποτε άλλο να ε, προσθέσω. Είναι τα ίδια ακριβώς πράγματα όπως αυτά που σας εξήγησα το Καρβουνάρι. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε. Ας στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε αν έχει κάτι ιδιαίτερο να μας πει. Πρόκειται για την κυρία Κανελοπούλου. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. Ε, εδώ πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ε, Περιβάλλον και Υφόρος Ανάπτυξη κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχει ολοκληρωθεί και είναι ε, λειτουργικό κατά τη δήλωση των ελληνικών αρχών ε, μέσα από τα έγγραφα κλεισίματος όπως τα παραλάβαμε τον Μάρτιο του 2016. Ε, τις πληροφορίες που είχαμε από την περιφέρεια Υπήρου τις ε, έχουμε ήδη μοιραστεί μαζί σας, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο στον, ε, στον φάκελο. Η, η περιφέρεια Υπήρου προέβησε συγκρότηση μιας επιστημονικής επιτροπής για την ερμηνεία και την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών του έργου, δηλαδή την ερμηνεία της μόλυνσης που παρατηρήθηκε ε, στην πηγή πλησίων του ΧΙΤΑ. Ε, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Επιστημονικής αυτής, ε, η περιφέρεια προέβη ε, σε διορθωτικές εργασίες στον ΧΙΤΑ, οι οποίες όπως μας έχουν δηλωθεί έχουν ολοκληρωθεί και ο ΧΙΤΑ λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, η ποιοτική εκτέλεση των έργων, όπως και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών με βάση τις εθνικές νομοθεσίες. Η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα παρέμβασης όταν το ελάττωμα που παρατηρείται ε, συνιστά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, ο ΧΙΤΑ λειτουργεί και ολοκληρώθηκε ορθά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Προτείνω να κάνουμε ακριβώς ε, το ίδιο όπως είπαμε προηγουμένως και ας περάσουμε στην επόμενη αναφορά, την 573 του... Α, δεν συγχωρείτε, πρώτος ο κύριος Πρέντα, πριν να προχωρήσουμε σε αυτή την αναφορά. Κύριε Πρέντα, ορίστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής. Είχα προετοιμάσει το φάκελό μου και θα ήθελα να σας πω να κλείσετε αυτές τις αναφορές. Ε. Μιλάμε για αναφορές του 2018 η μία και η άλλη του 2013. Η μία δεκάχρονη και η άλλη πεντάχρονη. Ε, μιλάμε τώρα για θέματα τα οποία έχουν ξεκινήσει πριν καν έρθω εγώ στο Κοινοβούλιο. Εγώ εξελέγην το 2009. Τι να σας πω τώρα. Ε, εάν θέλω να εκφράσω την ε, θέση του ΕΛΚ, ε, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κλείσουμε αυτές τις αναφορές και άλλωστε δεν άκουσα τίποτα συγκλονιστικό ως επιχείρημα έτσι ώστε ε, να κρατήσουμε ανοιχτή αυτές ε, τις, αυτές, ανοιχτές αυτές τις αναφορές και πώς να σας το πω εάν υπάρχει ένα πρόβλημα να κλείσουμε την αναφορά δέκα χρόνια μετά σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο βέβαια χαίρομαι γιατί είναι εδώ ο αναφερόμενος ε, γιατί το 8 είχε υπογράψει ως Ιωάννης Παπαδόπουλος και το 13 ως Ζων Παπαντοπουλός. Ε, βεβαίως είναι το ίδιο άτομο, αλλά πόσο, πόσα χρόνια θα περιμένουμε μέχρι ότου ο κύριος Ιωάννης, ε, κάθετος Ζων ε, Παπαδόπουλος ε, ασχολείται με το θέμα. Θα περιμένουμε να πάρει και τη σύνταξή του και εσαΐ. E. Θα συζητούμε για το θέμα αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, έχουν περάσει 10 χρόνια. Δεν μπορεί να κρατάμε ανοιχτή την αναφορά ακόμα. Ε, εντάξει, ε, η Κομισιόν μας λέει χύψη, μετά λέει υπάρχει κάποιος που λέει όχι δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι σωστά, ε, δίνω κάποια καινούργια στοιχεία, η Κομισιόν λέει α καλά τότε αφού έχετε καινούργια στοιχεία να τα ξανακοιτάξω, να διερευνήσω πάλι την κατάσταση και το μπαλάκι πάει από εδώ και από εκεί, ε, αλλά δεν φτάνουμε πουθενά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή με την οποία με ακούσατε ο κύριος Μαριάς. Well, yeah. Θα ήθελα να πω στο φίλο μου τον ε, κύριο Πρέντα, επειδή δεν ήταν προηγουμένως κατά τη συζήτηση, ότι οι απαντήσεις που ήρθαν και από την ελληνική κυβέρνηση και από τις περιφερειακές αρχές και στις προηγούμενες αναφορές δεν ήταν πιστικές και έγινε ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Επίσης είναι δεδομένο ότι παραμένουν δυστυχώς τα προβλήματα και παραμένουν γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν λάθος. Και ουσιαστικά σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα αυτής εδώ της μελέτης την οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Με την έννοια αυτή εμείς επιθυμούμε να μείνει ανοιχτή αυτή η υπόθεση. Υπάρχει πλήρης ε, συμφωνία, όχι για να συνεχίσει να έρχεται εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά γιατί δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα τοπικά και γιατί υπάρχουν πολλοί κάτοικοι οι οποίοι διαμαρτύρονται. Αυτό είναι το θέμα. Επομένω, φαντάζομαι ότι και εσεί, σαν έτσι ένα ευρωβουλευτή με ευαισθησία σε όλα αυτά τα θέματα, θα θέλατε να συνεχίσουμε την έρευνα και να πάρουμε πιστικέ απαντήσει. Δεν ήσασταν προηγουμένω να δείτε στη συζήτηση ότι δεν πήραμε απαντήσει ούτε από το Υπουργείο, το οποίο δεν ήρθε καν εδώ. Οι εξηγήσει που δόθηκαν ήταν ελάχιστε. Η περιφέρεια, ό,τι μα είπε, δεν είναι δεδομένο, αλλά και η Κομισιόν σα είπε ότι από τα χαρτιά που πήρε από τις ελληνικές αρχές προκύπτει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως οι κάτοικοι ισχυρίζονται και διαμαρτύρονται ότι υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς που είμαστε και περισσότερο χρόνο εδώ στην Επιτροπή Αναφορών θεωρούμε ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή, να το δούμε, διότι αποδεικνύει ότι έχουν περάσει χρόνια και δυστυχώ δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ε, σε αυτή την τοποθέτηση. Ευχαριστώ. If we do not trust the Commission, we have αν, δεν εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί τη φωνάζουμε τότε να έρχεται και να μας απαντά. Αν δεν εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε έτσι επάπειρον. Θα συνεχίσουμε τα ελληνικά, διότι μας παρακολουθούν βεβαίως, ε, μας παρακολουθεί το κοινό. Ναι, και είστε και στάρ, λέει ο κ. Πρέντερ. Όχι, όχι, δεν είμαι στάρ. Ακούστε, ακούστε. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι συζητήσαμε πολύ σοβαρά θέματα που αφορούσαν και τη Ρουμανία. Ήμασταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα τρένα. Και δώσαμε μεγάλη έμφαση και συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα με ευαισθησία στους πολίτες. Διότι εδώ είμαστε για να ακούμε τους πολίτες. Δεν είπα ότι δεν εμπιστευόμαστε την Κομισιόν. Είπα ότι η Κομισιόν δεν έχει κάνει πρωτογενή έλεγχο. Πήρε τα στοιχεία από την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς αυτά που ακούσαμε από την ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν πιστικά. Επομένως, επειδή έχουμε και άλλες δύο υποθέσεις πολύ πιο σοβαρές όπως θα δείτε, καλό θα είναι να συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μας εδώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή και αυτή η υπόθεση και να το προχωρήσουμε. Και αν από εκεί και πέρα δούμε ότι πρέπει να κλείσει, ευχαρίστως θα τις κλείσουμε. σα ευχαριστώ. As the petitioner wanted. Ο αναφερόμενος ζήτησε να το συζητήσουμε. Εγώ ήθελα να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα που να κάνουμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή θα στείλουμε τις επιστολές, θα κάνουμε το ίδιο όπως και με την προηγούμενη. Αυτό πρότεινα και οι ε, συνάδελφοί μου φάνηκε να συμφωνούν. Μέχρι ότου άρχισε να κουνάει λίγο τη βάρκα ο κύριος Πρέντα. Όμως πάντως η βάρκα ακόμα επιπλέει. Εγώ πάντως βλέπω ότι έχω υποστήριξη των συναδέλφων και θεωρώ ότι η κυρία Σακοράφα μου φάνηκε ότι θέλετε το λόγο για το επόμενο θέμα. Θέλω να εξηγήσω στον κύριο συνάδελφο ότι είμαστε εδώ ναι, ναι, ναι. ακριβώς για αυτό το λόγο. Οι πολίτες ε, εμπιστεύονται εμά. Έρχονται εδώ διαμαρτυρώμενοι για προβλήματά του, τα οποία με συγχωρείτε πάρα πολύ άπτονται και τη υγεία του πια. Δεν είναι μόνο ότι είναι ιδιότροποι και θέλουν να εμφανίζονται κάθε τρει και λίγο σε αυτή την επιτροπή. Εμεί λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι εδώ και να του ακούσουμε και αν χρειαστεί να κάτσουμε και 10 και 20 χρόνια με την ίδια αναφορά. Τι να κάνουμε τώρα αν δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Αυτό. Και συμφωνώ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που θεωρείτε ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ έω ότου η Επιτροπή φέρει τα στοιχεία τα οποία θα πείσουν και εμάς που ψηφίζουμε εδώ ότι όλα πάνε καλά. I know that I have now... Η Πρόεδρος. Βλέπω ότι έχω ευρία υποστήριξη στην Επιτροπή Αναφορών, κυρία Πρέντα, ίσως την επόμενη φορά λοιπόν. Α, α, πέτεριά. Τώρα στο τέλος της συζητήσεως να μου επιτρέψετε να κάνω μια συμβαστική πρόταση και ο κ. Μαριάς έχει δίκιο και ο κ. Πρέντα έχει δίκιο χρειάζεται να εργαζόμαστε στοχευμένα. Μπορεί κανεί τότε, στην περίπτωση αυτή, να κλείσουμε μια αναφορά. Λέει και ο κ. Μαριάς ότι ε, δεν συμφωνούμε με τις πληροφορίες που μας δίνουν. Και η δεν δίκιο έχει. Η παράκλησή μου λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, πώ να πω, κάντε κάντε τα στοιχεία, πώς να το πω, να μας δείξετε, να μας δώσετε στέρεα στοιχεία, ώστε να μην υπάρχει πλέον λόγος δυσπιστίας. Εγώ θεωρώ ότι και δύο πλευρές έχουν δίκιο. Και ο Πρέντα έχει δίκιο. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουμε. Κρίστιαν, έχει δίκιο. Δεν είπα αυτό. Και η πρόεδρος νομίζω πρότεινε μια σωστή συμβαστική λύση. Ας δώσουμε εμπιστοσύνη στην Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και να βάλω και κάποια τάξη στην ε, συνεδρίαση τη ε, Επιτροπής Αναφόρων. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε και να ε, αλλάξουμε σελίδα, να πάμε στην 573 του 2011 σχετικά με σοβαρά σφάλματα και παραλήψεις στην έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτινόμενη τοποθεσία υγειονομική ταφής απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού και στην 0078 για την κατασκευή χώρου διάθεση απορριμμάτων σε τοποθεσία της Ανατολικής Αττικής. Λίγο πολύ το ίδιο θέμα, αλλά κάπως φωτισμένο από διαφορετικές σκοπιές. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους αναφερομένους, στον κύριο Παπαδηγενόπουλο και στον κύριο Γκίκα για λίγα λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, έχω καταθέσει ένα υπόμνημα 30 σελίδων και θέλω να με πιστέψετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να το συμπιέσω σε 5 λεπτά. Όμως θα το προσπαθήσω αφού αυτοί είναι οι κανόνες. Ε, πέντε ερωτήματα πρέπει να λάβουν απάντηση. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που έχει θέσει η ίδια η Επιτροπή σας είναι ικανοποιητική η τροποποίηση της περιβαλλοντικής άδειας που ζητούσε η Επιτροπή Αναφορών. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναδρομή. Το 2003 ε, πραγματοποιήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου χωρίς να ληφθούν υπόψη η τότε υφιστάμενη νομοθεσία. Η Ελλάδα δεν είχε υιοθετήσει, δεν είχε εσωτερικεύσει το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, το 2003, η μελέτη του 2003 αναφέρει και λέει ότι έχει λάβει υπόψη την τεχνολογία του 1994. Δεύτερη ημερομηνία σημαντική. Το 2009 ξεκινάει η κατασκευή του έργου, το οποίο γίνεται, όπως είπα και προηγούμενα, με τη μελέτη του 2003. Το 2009 και το 2013 έπρεπε να υπάρξει τροποποίηση όπως επιβάλλει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Κυρία Πρόεδρε, δεν υπήρξε καμία τροποποίηση διότι οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ρητά και υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα. Δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση διότι δεν έχει αλλάξει η υφιστάμενη νομοθεσία. Όμως οι, οι κύριοι βουλευτές εδώ γνωρίζουν καλύτερα από μένα ότι τη δεκαετία 2003-2013 υπήρξε μια έκρηξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μία ανόρθωση, νέες έννοιες, νέες δυνατότητες και πολύ περισσότερο την δεκαετία 2003-2013 υπήρξε μία, μεγάλο, ε, μία μεγάλη ε, ε, ε, εκτείναξη της ε, ίδιας της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Ε, τον Ιανουάριο του 2015 το κυρίως έργο, κυρία Πρόεδρε, έχει σχεδόν τελειώσει. Έχει τελειώσει. Και η μελέτη αυτή η οποία σήμερα η περιφέρεια ισχυρίζεται ότι έχει πραγματοποιήσει, μάλλον η τροποποίηση της μελέτης που, που ισχυρίζεται ότι έχει που έχει πραγματοποιήσει, έγινε το Νοέμβρη του 2015. Και τι αλλάζει η τροποποίηση επιτέλους την οποία ζητούσαμε τόσο καιρό κυρία Πρόεδρε. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Αλλάζει κάποιους δρόμους που πηγαίνουν, εισέρχονται στο χιτά, τους κάνει λίγο μεγαλύτερους και αλλάζει το χώρο του βιολογικού καθαρισμού και τον πάει 35 μέτρα αριστερά ή δεξιά, δεν θυμάμαι. Έτσι λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, έχουμε μία μελέτη που έγινε το 2003 και ε, αναφερόταν στα τεχνολογικά δεδομένα και στην ομοθεσία του 1994. Και σήμερα το 2018, 24 χρόνια μετά, έχουμε ένα έργο που έχει σχεδιαστεί το 1994. Είμαστε πίσω λοιπόν 28 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προχώρησε, ε, έχει λάβει νέα δεδομένα, υιοθετήθηκε η οδηγία IPPC και αυτή η νομοθεσία πέρασε από το έργο και δεν το είδε. Δεύτερο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε, που είναι κομβική σημασία. Το έργο αυτό έχει χτιστεί πάνω σε ρέμα ή όχι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία μνημονεύει συνεχώς η Κομισιόν, που λέει ότι δεν υπάρχουν ρέματα στην περιοχή, είναι μία απόφαση η οποία κρίνει επί της ουσίας ή επί της διαδικασίας. Αυτά είναι τα δύο βασικά ερώτημα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να σας πω για κάτι παράδοξο που αναφερόταν στις συστάσεις της ίδιας Επιτροπής σας μετά την επίσκεψη στο γραμματικό. Τι έλεγε ίδια η Επιτροπή Αναφερών. Διαβάζω επιλέξει. Να επιτρέπεται, έλεγε, στους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου να εκτελούν την εργασία τους ανεξάρτητα και έγκαιρα. Δηλαδή ζητούσε μία υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελλάδας να είναι ανεξάρτητη. Γιατί το έλεγε θα καταλάβετε παρακάτω. Ε, μετά από αυτήν την υπόθεση, οι επιθεωρητέ περιβάλλοντο, η υπηρεσία για την οποία μιλούσαν, βγάζουν την τελεσίδικη και απόφασή του, κυρία Πρόεδρε. Και τι λέει αυτή η απόφαση, ότι το έργο είναι πάνω σε ρέματα και στέλνουν την υπόθεση στον εισαγγελέα. Μετά από αυτό, κινητοποιείται ο μηχανισμό. Σε λίγου μήνε το ΣΤΕ βγάζει την απόφαση την οποία σα είπα. Έχετε λάβει, κυρία Πρόεδρε, μία επιστολή από, μία, από τι επιθεωρήτριε περιβάλλοντος, όπου καταγγέλει πολύ συγκεκριμένα ασφικτικές πιέσεις εκ μέρους της πολιτικής ηγεσία αναφέρει φωτογραφική αλλαγή της νομοθεσίας περί ρεμάτων, ώστε όλα αυτά τα θέματα να φτάσουν τακτοποιημένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ε, έχω, έχω δώσει στην Επιτροπή, στην ΠΕΤΗ, έχω δώσει ε, γνωμοδότηση ε, η οποία αναφέρεται στη φύση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ρητά λέει, και αυτός που βγάζει τη γνωμοδότηση είναι ο ίδιος δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρητά λέει ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχουν χαρακτήρα ουσιαστικό, αλλά απλώς έχουν χαρακτήρα διαδικαστικό. Τρίτο θέμα, κυρία Πρόεδρε. Ε, Οχητά γραμματικού, κατά τη δική μα αντίληψη, είναι έργο επικίνδυνο. Είναι όμω και έργο χρήσιμο. Δύο νούμερα για να σα βοηθήσουν αν αυτό το έργο είναι χρήσιμο. Υποτίθεται ότι αυτό το έργο, κυρία Πρόεδρε, έχει γίνει για να ανακουφιστεί η πολύπαθη φυλή για την οποία θα μιλήσουμε ακριβώ μετά. Τα στοιχεία έχουν ως εξή. Κάθε μέρα στην Αττική συλλέγονται 6.000 6.000 ε, τόνοι ε, απορριμμάτων. Ο χιτά γραμματικού, όπως λέει ε, η ίδια η περιφέρεια στον Πεσδά, θα πρέπει κάθε χρόνο να δέχεται 60.000. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια ανακούφιση, θα υπάρχει μόνο και μόνο για 10 μέρες. Στις υπόλοιπες 355 μέρες του χρόνου, ο χιτά φυλής θα δέχεται τα ίδια σκουπίδια. Όταν ακούνε στη φυλή ότι θα βελτιωθεί η κατάστασή τους, πραγματικά πιστεύω ότι γελάνε. Ένα τελευταίο στοιχείο, κυρία Πρόεδρε. Ο... Ζητάει, η Επιτροπή σας τα οικονομικά δεδομένα. Με μελέτες οι οποίες υπάρχουν και τις έχω παραθέσει, ο τόνος στη φυλή κοστίζει σήμερα 6.000 Παρακαλώ να κλείσετε γιατί σας έδωσα 5 λεφτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίκας. Εσείς έχετε κάτι να προσθέσετε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε ότι είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Ναι, πέντε λεπτά. Έχω και εγώ PowerPoint να σας παρουσιάσω. Προσπαθώ. Ε, θα κάνω την παρουσίασή μου στα ελληνικά. Ε, είναι τα μάτια του στραμμένα εδώ στην Επιτροπή. Ε, οι μαθητέ έχουν διαδηλώσει, οι κάτοικοι έξω από το χιτά. Συζητάμε ακόμα μια φορά για την νομιμότητα του χιτά χιτή, ο εδάγα στο γραμματικό, ενώ υπάρχει ήδη απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων που το χαρακτηρίζει παράνομο. Και ε, προσθέτω ότι το Ταμείο Συνοχή, Cohesion Funds, που το έχει, το έχει απετάξει από το προγραμματισμό του και έχει διακόψει τη χρηματοδότησή του, έργο που παραβιάζει την παραβολητική νομοθεσία. Επίσης, παραπομπή τη υπόθεση στο Όλαφ, η οποία εξετάζει την υπόθεση. Σα ζητώ λοιπόν, σαν Επιτροπή, ω Επιτροπή, να καλέσετε το Ταμείο Συνοχή, την Επιτροπή Όλαφ και να μα πει τι γίνεται με την υπόθεση του Ιχτά Γραμματικού. Γιατί το Ταμείο Συνοχή έχει πάρει πίσω τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Ε, πριν λίγου μήνε δημοσιεύτηκε μελέτη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ΙΓΜΕ, την οποία ανέθεσε η Περιφέρεια Αττικής προσποιούμενο ότι ε, συμμορφώνεται. Όμως, η μελέτη του ΙΓΜΕ που ανέθεσε η Περιφέρεια προσποιούμενο ότι συμμορφώνεται με τις εντολές της Επιτροπής Αναφορών έρχεται να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ρέματος λεκάνης απορροής 1200 στρέμματα. Το βλέπετε και στο βίντεο. Και την υδατοπερατότητα του εδάφους. Έχει γίνει σχετικό σημείωμα από τον κύριο Δημήτρη Δαμάσκο, μηχανολόγο μηχανικό, όπως και από καθηγητές για το θέμα αυτό. Ε, το τι γίνεται το βλέπετε στο βίντεο. Η κήρυξη του Νοτιού Ευρωϊκού σε ζώνη ειδική προστασία έχει τεθεί ειδική επιστολή από το Κέντρο Βιωσιμότητα. Εντάχει, είμαι στο ένα λεπτό. Ε, έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Έρευνα με πρωτοβουλία τη καθηγήτρια κυρία Αθηνά Λινού. Πανεπιστημιακοί καθηγητέ θέτουν το μείζον ζήτημα τη αρχή τη προφύλαξη για το χιτά γραμματικού. Πρώτη φορά έχω στα χέρια μου χάρτες εδώ, τα οποία θα τα καταθέσω στην γραμματεία από την περιφέρεια, που υπάρχει σε άλλους χάρτες τη της και της αδειοδοτούσας αρχής η, ο, η οριοθέτηση του ρέματο και σε άλλου το αποκρύβουν με μπλάνκο. Και ε, είμαι πολύ σύντομος, στα δύο λεπτά. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία της περιφέρειας Αττικής ως προς αυτά που επισήμως σας δηλώνει περί ελέγχου της ασφαλούς χωροθέτησης και λειτουργίας του έργου, διότι έχει ήδη εντάξει το χιτή ε, του γραμματικού στο νέο ΠΕΣΔΑ με χωρίς ε, νέες μελέτες και χωρίς να περιμένει την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών, αλλά ούτε και τα αποτελέσματα της μελέτης του ΙΓΜΕ που ήδη ε, ίδια ανέθεσε. Παράλληλα και παρά τι ανακοινώσει και τι δηλώσει τη ενώπιό σα, δηλαδή τη Περιφέρεια Αττικής, δεν έχει προχωρήσει στη διαχείριση των απορριμμάτων εφαρμόζοντα πολιτικέ πρόσληψη, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, ανάκτηση αποκεντρωμένη διαχείριση με εφαρμογή κινήτρων προ όφελο του πολίτη και ό,τι προβλέπεται από αυτήν η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και κλείνω, είμαι στα τρία λεπτά κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα μα είναι περί τι τέσσερι φορέ δαπανηρότερη ε, σύμφωνα με το κατακεφαλή ΑΕΠ από τον Ευρωπαϊκό Μέσον Όρο, όντα παράλληλα ανάμεσα στι τελευταίε από πλευρά ανακύκλωση. Σε απόλυτου αριθμού αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μα οι, πολιτι... πολίτε χάνουν από την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω παραπάνω σε αναλογικό αναλογική σχέση με τι υπόλοιπε καπιταλιστικέ ευρωπαϊκέ χώρε. Έχετε πάρει μνημονιακέ πολιτικέ κατά τη χώρα μου και μάλιστα οι περισσότερε από αυτέ χαρακτηρίζονται σκληρέ και κάποιε από αυτέ χαρακτηρίζονται από πολλού αντίρροπε με την ανάπτυξη. Ήρθε η στιγμή να πάρετε μια απόφαση που είναι για το γενικό καλό και της οικονομίας και του περιβάλλοντος, απαγορεύοντας στη χώρα μου την οποιαδήποτε διαχείριση σύμμικτων απορριμμάτων. Υπάρχει άλλωστε και η απόφαση 2012 που το αναφέρει τα αυτό. Είναι προφανές ότι γύρω από τα σύμμικτα έχουν αναπτυχθεί στευρές πολιτικές διασπάθησης ευρωπαϊκών κοντιλίων. Αφαιρώντας τους τα σύμμικτα θα προωθηθεί η ανακύκλωση με ανταποδοτικότητα προς όφελο του πολίτη. Το είπε άλλωστε και η έκθεση. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στα τέσσερα λεπτά. Νομίζω είμαι πολύ ευγενή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, would... Συνεχίζει η πρόεδρος. Διακόπτει κάποιος χωρίς μικρόφωνο. Το μόνο που θα ήθελα να πω ακόμη συνεχίζει ο αναφερόμενος. Βλέπετε εκεί από τις βροχοπτώσει Κάθε φορά που υπάρχει βροχόπτωση έχουμε την ίδια εικόνα. Τώρα, ε, το 2015 βλέπετε, ε, το 2017, ε, βλέπετε τους χάρτες της περιφέρειας Αττικής και βλέπετε τη ρήπανση στις φωτογραφίες που δείχνω. Είναι προφανής και στο σεξισμό των μαθητών που ε, ξεσηκώθηκαν για να γίνει όλη αυτό το ε, η, η αναστάτωση, για πάση περιπτώσει ο κόσμος ε, αντιδρά. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν πρέπει το σκοπίδι να μπαίνει όλο σε μια μαύρη σακούλα. Αυτή είναι η φωτογραφία από το συστημάτων μπλε κάτω ανακύκλωσης που όπως θα δείτε δεν γίνεται ανακύκλωση. Ε, σκάνδαλα με συστήματα ανακύκλωσης. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την... Ε- Διακόπτει ο κ. Μαριάς. Όχι ακόμη. Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο του Μαραθώνα να έρθει. Ναι, ναι. Με πρώτα η Κομισιόν, μετά η Περιφέρεια, μετά ο Δήμαρχος Μαραθώνος. please. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ονομαζόμαι Θεοδόσιο Σαμπανιώτη, απλώ για όσου δεν άκουσαν το όνομα, ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική. Ε, το έργο τη κατασκευή του ΧΙΤΑ, όπω ονομάζονταν τότε, της, στην Νότια ανατολικη Αττική στη θέση Μαύρου Βουνό Γραμματικού, είναι ένα έργο του Ταμείου Συνοχή τη περίοδου 2000-2006. Ε, Όπω γνωρίζετε, ήδη έχει αναφερθεί και σε περιότητε συνεδριάσει. Ε, έχουμε στείλει ένα μια επιστολή κλεισίματος στις ελληνικές αρχές, μια πρόταση κλεισίματος στις ελληνικές αρχές στις 14 Ιανουαρίου του 2015 και με την επιστολή προτάθηκε δημοσιονομική διόρθωση του 100% της χρηματοδοτικής συνδρομής του Ταμείου Συνοχής επειδή το έργο δεν ήταν ολοκληρωμένο και λειτουργικό, καθώς και για περιβαλλοντολογικούς λόγους οι ελληνικές αρχές με επιστολή τους ε, το Μάρτιο του 2015 δεν αποδέχτηκαν την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Ακολούθησε αλληλογραφία, όχι αλληλογραφία, email περισσότερο με τις ελληνικές αρχές, κατά τις οποίες κατατέθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες. Ε, κατά τις οποίες οι ελληνικές αρχές μας ενημερώνουν για την πρόοδο του έργου αναφορικά με τα κρεμούντα ζητήματα. Το έργο, κατά την άποψη τη Επιτροπή, παραμένει μη ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Έχει ετοιμαστεί και αν δεν έχει αποσταλεί ήδη, θα αποσταλεί τι επόμενε ημέρε επιστολή προδιόρθωση στι ελληνικέ αρχέ, ε, κατά την οποία ζητάμε την 100% ε, δημοσιονομική διόρθωση τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχή. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Η σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Παπαχρυσοβέργη να λάβει το λόγο. Περιφέρεια Αττικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσει πρώτος ο κύριος Δήμαρχος Γραμματικού, διότι είναι καλύτερα να μπορέσω μετά να απαντήσω σε όλα τα θέματα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό αν συμφωνείτε. Ωραία, ευχαριστώ. λοιπόν θα προσκαλέσω τον Δήμαρχο ε, Μαραθώνος κύριο Ψινάκη να λάβει το λόγο. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και εκπρόσωποι της Κομισιόν. Καταρχάς πριν αρχίσω θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που φοράω γυαλιά, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Δεν είναι από έλλειψη σεβασμού, αλλά έχω ένα προβληματάκι στο μάτι. Δεύτερον, είμαι πολύ, σαν Έλληνα, είμαι πολύ κολυκευμένο και συγκινημένο που σα άκουσα, κυρία Πρόεδρε, να μιλάτε τόσο καλά ελληνικά. Σήμερα ήρθα σε εσά γιατί είναι το ψηλότερο σημείο που μπορώ να φτάσω, μπα και σωθεί τελευταία στιγμή ο Μαραθώνα. Γιατί μετά από τη δικιά σα επιτροπή είναι ο Θεό. Αλλά τον οποίο βέβαια θα συνοντήσω σύντομα λόγω ηλικία, αλλά ο Μαραθώνα θα έχει καταστραφεί. Στην Ελλάδα Όπου και να σκάψεις, αναβλέει πολιτισμός. Ο Μαραθώνας είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Έχει αρχαία πόλη το Ραμνούντα που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της αρχαίας Ελλάδος από την Αθήνα. Αρχαίους Αιγυπτιακούς ναούς με τάφου, τάφους, αρχαιολογικό μουσείο με συγκλονιστικά ευρήματα και είναι βέβαια και όλος γνωστό σαν brand name λόγω μαραθωνίου. Ο σύγχρονος μαραθώνας που είναι ένας από τους μεγαλύτερου δήμους της έχει τεράστια πλάζ, πάρα πολλά χιλιόμετρα ε, και και, από τη, και ε, τις στην Ελλάδα και σίγουρα μεγαλύτερε στην Αττική. Έχει επισκέπτε, έχει δάση, μοναστήρια, Ολυμπιακέ και αθλητικέ εγκαταστάσει και βέβαια έχει και τον κλασικό αθλητικό μαραθώνιο που είναι το κέντρο του αθλητισμού όλου του κόσμου σε αυτό το σπορ. Βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο και αυτό έχει σημασία που σα λέω στα επόμενα ε, και δεσπόζει στην Ανατολική Αττική. Είναι 12 με 15 λεπτά από το αεροδρόμιο, το Athens International Airport και, και λιμάνι δίπλα που πάνε όλοι στα νησιά. Και αυτό σας το λέω γιατί η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας με τη, με τη βαθιά κρίση που εσείς καλύτερα ξέρετε από εμά τι περνάμε στην Ελλάδα με την κρίση είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ο τρόπος που εξαργυρώνουμε τον πολιτισμό και την ε, κληρονομιά των προγόνων μας. Ήρθα εδώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με δεχτήκατε, γιατί αυτή τη στιγμή ο μαραθώνας κινδυνεύει και είναι στο παραπέντε να σκάσει μια τοξική βόμβα που θα του καταστρέψει ολοσχερός. Η βόμβα αυτή είναι περιβαλλοντική, υγειονομική, κοινωνική και άμα σκάσει δεν θα μολύνει μόνο τον μαραθώνα, αλλά και τους όμορους δήμους και τον νότιο ευωικό κόλπο. Σας έφερα και ήρθα εδώ και σας έχω φέρει πολλά νέα στοιχεία που έχουμε μαζέψει με τους συνεργάτες μου και γι' αυτά τα νέα στοιχεία έχουν ενημερωθεί οι ελληνικέ αρχέ. Αυτά τα στοιχεία αντικρούουν αυτά που έχετε ω τώρα, τα οποία είναι, ε, λέω, ελλειπή για να μην πω ανακριβή. Έχουμε νέα στοιχεία για τα ρέματα, που εσεί γνωρίζετε καλύτερα από όλου γιατί έχετε στείλει και έχετε κάνει από, ε, που έχετε ήδη κάνει αυτοψία. Και βέβαια με τι κλιματολογικέ αλλαγέ του πλανήτη έχει επηρεαστεί βεβαίω και η Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε πλημμύρε, φωνικέ πλημμύρε, που στην πλημμύρα, σε περίπτωση που γίνει το χιτά, θα έχουμε τρομερή μόλυνση. Ε, αποδεικνύουμε με τα στοιχεία αυτά που σας φέραμε ότι το έργο δεν έχει περιβαλλοντολογική αδειοδότηση και δεν ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία που εσείς ευτυχώς έχετε θεσπίσει στην Ευρώπη. Αποδεικνύουμε την πληγή που θα δημιουργηθεί στις αγροτικές περιοχές του Μαραθώνα, γιατί είναι αγροτική η περιοχή του Μαραθώνα και τροφοδοτεί όλη την Αθήνα και την Αττική με τα προϊόντα που βγάζει. Οπότε καταλαβαίνετε τι η καταστροφή θα έχει γίνει. Και πάνω απ' όλα, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα στον Δήμο Μαραθώνα, έχουμε ένα σχέδιο διαχείριση των απορριμμάτων μα. ένα σχέδιο σύμφωνα απόλυτα με του κανόνε, νομίζω το έχετε λάβει κύριε Πρόεδρε, με του κανόνε για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντολογική Νομοθεσία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα της φυλής και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει και είναι ένα έγκλημα Ξέρουμε για τους καρκίνους που έχουν προκαλεστεί, την τοξικότητα, τις τερατογενέσεις και ξέρουμε πάρα πολύ καλά επίσης ότι δεν μπορείς να πετάς τα σκουπίδια σου στην αυλή του γείτονα. Αυτό απαγορεύεται. Το σχέδιο, το σχέδιο δράσης που έχουμε ετοιμάσει λαμβάνει υπόψη του όλα τα παραπάνω και είναι απόλυτα σύμφωνο με την ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Το δικό μας κοστίζει, το έχουμε καταθέσει με αριθμό πρωτοκόλλου, ε, on time, όταν στην αρχή της ε, θητείας μας, κοστίζει 8 εκατομμύρια ευρώ και όχι 60, που είναι το κόστος ενός τμήματος του σχεδίου της περιφέρειας. Ε, να μην συζητήσουμε για τα 33 εκατομμύρια ευρώ που ήδη έχει κοστίσει το έργο. Και όλο αυτό για να ανακουφίσει, υποτίθεται, τη φυλή για 10 μέρες το χρόνο. Δηλαδή, οι δυτικέ συνοικίε, η η δυτική Αττική έχει δηλητηριαστεί και έχουν όλα αυτά τα προβλήματα περιβάλλοντο υγεία και κάτι και είναι σε τραγική και τα παιδάκια και έχουν καρκίνους και τέτοια. Και να μολύνουμε και την άλλη τέτοια για δέκα μέρε. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι λύση. Να μολύνει τα πάντα για δέκα μέρε. Αν, αν μπορούσε να γίνει κάτι, να πει ότι. Οπότε σα καλώ να δώστε σε μένα και σε όλου του κατοίκου, όχι μόνο του Μαραθώνα, αλλά και όλων των όμορων Δήμων και των επισκεφτών, που είναι πάνω από 400.000, την ευκαιρία να ζήσουμε στον παράδεισο που σας έχω περιγράψει και πολλοί από εσά τον έχουν δει. Σας προσκαλώ να έρθετε στο Μαραθώνα, να επισκεφτείτε τους χώρους που, που δεν μπορείτε, γιατί αν μολυνθείτε δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, ούτε να κάνετε μπάνιο, ούτε να δείτε, θα έρθετε να δείτε τα μουσεία, ούτε να τρέξετε στο, σε καθαρό αέρα στο κλασικό μαραθώνιο ή όπου αλλού θέλετε. Σας παρακαλώ, πραγματικά σας παρακαλώ να απαιτήσετε να εφαρμοστούν οι κανόνες και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φροντίζουν για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Και αν γίνει αυτό, το σίγουρο είναι ότι το έργο θα σταματήσει. Αν ακούσουν τις κανόνες που εσείς θέσατε και είναι η Ευρώπη in order σε τάξη, θα σταματήσει αυτό το έργο. Δεν θα γίνει ποτέ το έργο. Θα σα αποκαλώ βέβαια σωτήρες τη Ανατολική Αττική και του Εβοϊκού Κόλπου μόνο αν απαιτήσετε να τηρηθούν αυτοί οι κανόνε. Και κλείνω για να μην σα κουράσω και προσπαθώ να το πάω γρήγορα. Κλείνω. Το 490 π.Χ. έγινε η μάχη του Μαραθώνα, η γνωστή μάχη του Μαραθώνα σε όλο τον κόσμο, που λίγοι Έλληνε εμπόδισαν την εισβολή των χιλιάδων Περσών στην Ευρώπη. Έτσι σώσανε το δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, γιατί στην αντίθετη περίπτωση τώρα εδώ μέσα θα είμαστε άλλοι. Ήταν μια μάχη σαν αυτή του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Το, το 2018 τώρα επικαλούμεθα να σώσουμε τον μαραθώνα από αυτή την τραγική καταστροφή που τον περιμένει. Είναι μια άνηση μάχη πάλι που οι συνεργάτες μου και εγώ δίνουμε και εγώ κάνω και λίγο το Δαβίδ, μόνο σε αυτή την, την περίπτωση ο Δαβίδ είναι λίγο ηλικιωμένος το όπλο μου είστε μόνο εσείς. Και οι κανόνες που κρατάνε την Ευρώπη σε αυτό το ψηλό επίπεδο και είναι οι μόνοι που αν τηρηθούν το έργο δεν θα γίνει και ο μαραθώνας δεν θα γίνει σκουπιδότοπος. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και που με ακούσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε με, με τις συναδέλφους. Ε, πρώτα, κυρία Σακοράφα. Exactly now, Α, με η περιφέρεια Αττικής. Ο κύριος Παπαχρυσοβέργης. Ορίστε παρακαλώ κύριε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, κυρίες και κύριοι. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, πρέπει να μου επιτρέψετε να τονίσω κάποια ζητήματα που αναφέρθηκαν συγγνώμη, για να ε, για να αντιληφθείτε καλύτερα την ουσία του ζητήματος και να θέσουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του ε, διαστάσεις, μιας και προτιμήσαμε να έρθουμε εδώ σήμερα από το να σας στείλουμε μια επιστολή, παρόλο που σας στείλαμε και ε, πολλά στοιχεία τις τελευταίες ημέρες. Καταρχάς πρέπει να σας ενημερώσω ότι η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής άλλαξε ριζικά την πολιτική για διαχείριση των απορριμμάτων στη βάση όσων προανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση και όλα με τη μελέτη την οποία ε, αναμένουμε με μεγάλη ε, χαρά να την ε, αναγνώσουμε. Συγκεκριμένα, από τις 23 Δεκεμβρίου του 2016 η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ένα νέο πλάνο διαχείρισης απορριμμάτων, το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής, που στηρίζεται ακριβώς στις βασικές αρχές κατευθύνσεις και στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα αναφέρουμε στην οδηγία 98 του 2008 συνάδει με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία. Το περιφερειακό σχέδιο άλλωστε αποτελεί προϊόν ευρείας διαβούλευσης, μάλιστα περιλαμβάνονται αυτούσια τα τοπικά σχέδια διαχείρισης ε, απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής. Σε αυτό δεν προβλέπεται πλέον η δημιουργία χώρων υγειονομικής σταφής απορριμμάτων στην Αττική, κυρία Πρόεδρε. Το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για την περιφέρεια Αττικής αντί το αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης των προηγούμενων δεκαετιών που ήθελε όλα τα σκουπίδια της Αττικής να θάβονται στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της φυλής, προβλέπει την αντιστοίχηση έξι μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων με τρεις χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων σε ίση και δίκαιο όσο το ε, δυνατό κατανομή σε όλη την Αττική. Βρισκόμαστε έτσι στον αντίποδα τη πολιτική τη προηγούμενη διοίκηση. Είτε πρόκειται για το χιτά φυλή, είτε πρόκειται για το χιτά γραμματικού. Συγκεκριμένα, ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή μιας πρώτης ψυχολογικής μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στο γραμματικό. Μια μονάδα επεξεργασίας που αντιστοιχεί σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής μικρής δυναμικότητας, ε, έχει μια δυναμικότητα επεξεργασίας 60.000 τόνους ε, το χρόνο. Πρόκειται για καθόλου νέο σχεδιασμό. Και αυτό γιατί ενώ στον προηγούμενο σχεδιασμό το έργο που υλοποιούνταν αφορούσε στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής και μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για την υποδοχή του 33% προσέξτε του 33% των απορριμμάτων που παράγονται σε όλη την Αττική. Ο σημερινός σχεδιασμός στη βάση της αρχής της εγκύτητας και της δίκαιης κατανομής της διαχείρισης των απορριμμάτων, ό,τι ακούσαμε ορθό σήμερα δηλαδή, προβλέπει ότι στο γραμματικό θα γίνεται διαχείριση μόλις του 3% των απορριμμάτων που παράγονται στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση που θα λειτουργήσει στο γραμματικό, εγκατάσταση ολοκληρωμένη και σύγχρονη, όχι με σχέδια το 1994, θα προσφέρεται μόνο για την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτή είναι και η υλοποίηση τη δέσμευσή μα ενώπιον σα, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, όπω πράξαμε πριν από τρία χρόνια περίπου στι 16 Απριλίου του 2015. Αποκλείσαμε λειτουργία χώρου υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο γραμματικό και το κάνουμε πράξη. Δεν πρόκειται για εξαγγελίε και θα το καταλάβετε αμέσω. Πρώτον, είπαμε, χιτά δεν θα λειτουργήσει το γραμματικό και σακούλα απορριμμάτων δεν θα θαυτεί. Δεύτερον, δεσμευτήκαμε και για το εξή. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τεκμηριωμένα με την επιστημονική συμβολή ανεξάρτητων και επίσημων εμπειρογνωμόνων εδεχόμενη κίνδυνη ρήπανση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, η Περιφέρεια Αττικής έχει δεσμευτεί να αναζητήσει τις βέλτιστες εκείνες τεχνικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την οριστική εξάλληψη των όποιων κινδύνων ελοχεύουν, προκειμένου να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υλοποιώντα τη δέσμευση αυτή, προκειμένου να έχουμε την επιστημονική διαβεβαίωση για την εγγύηση ασφάλειας και τη προστασία τη ευρύτερη περιοχή και των πολιτών εν ώψη τη λειτουργία χώρου υγειονομική ταφή υπολοιμάτων, απευθυνθήκαμε στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, γνωστό στη χώρα μα ω ΣΥΓΜΕ, έναν ανεξάρτητο φορέα της πολιτείας με θεσμικό κύρος και ζητήσαμε τη σύνταξη έκθεση αξιολόγησης. Εκπληρώνουμε έτσι τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της κοινοτικής οδηγίας της πρώτης του 2008, της λεγόμενης οδηγίας IPCC, για δραστηριότητες υψηλού δυναμικού ρήπανσης. Το κεντρικό συμπέρασμα τώρα της έκθεσης του ΙΓΜΕ είναι ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη γεωλογική διερεύνηση, προσέξτε, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν εμπόδιο στη λειτουργία του έργου. Περαιτέρω, σα γνωρίζω ότι στο πλαίσιο διερεύνηση επιπλέον θεμάτων, όπω αυτά είχα σημειωθεί στη σχετική σα πρόσκληση, κυρία Πρόεδρε, του 2015 και αφορούσε περιβαλλοντικά ζητήματα, σας γνωρίζουμε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου ανανεώθηκαν στις 4 Νοεμβρίου του 2015 με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υποβάλαμε στην αξιότιμη επιτροπή σας και τη σχετική απόφαση. Η εν λόγω αντικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου τώρα πραγματοποιήθηκε ύστερα από την προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες πράξεις παράβασης του ίδιου Υπουργείου. Και δεν υφίσταται πλέον καμία εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς είναι όχι απλά φανερό, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι το έργο αυτό δεν απειλεί ούτε τη δημόσια υγεία ούτε το περιβάλλον να σημειωθεί ότι κατά επανάληψη έχει επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο Επικρατεία τη χώρα μα αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν διαπιστώνεται καμία παράβαση τη ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή τα έργα που ε, συνεχίζονται στο γραμματικό και αναμένεται, σα ενημερώνω, να ολοκληρωθούν στι 31 Αυγούστου 2018 αφορούν ακριβώ τη συμμόρφωση στου νέου περιβαλλοντικού ε, όρου όπως για παράδειγμα γίνεται αποκατάσταση της δαστικής βλάστησης και αναδάσωση 105 στρεμάτων. Κοινοποιήσαμε στην αξιότιμη επιτροπή σας, ε, κυρία Πρόεδρε, σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ της χώρας μας για την υλοποίηση του έργου και που εξηγεί γιατί δεν πρέπει να απολεστούν κοινωτικοί πόροι από τις καθυστερήσεις που εμφάνισε η κατασκευή του στο παρελθόν και για ποιου χώρου το έργο αυτό θα αναβαθμιστεί και θα ενταχθεί στον περιφερειακό μα σχεδιασμό. Επίση, αξιοποιώντα τα πρώτα 150 εκατομμύρια που διατέθηκαν στην περιφέρεια Αττική μέσω του ΕΣΠΑ για έργα απορριμμάτων, θα συμπληρώσουμε το γραμματικό στι απαιτούμενε μονάδε επεξεργασία και κομποστοποίηση που απαιτούνται για να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Μονάδε για την πλήρη αξιοποίηση του χώρου, λοιπόν, για την τοπική και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Κοιτάξτε, οι πολίτε έχουν δίκιο να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τη χωροθέτηση μια εγκατάσταση διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή του και να μην πιστεύουν στι προθέσει των αρμόδιων αργών. Το παρελθόν αυτό του έδειξε. Αυτή είναι για μα η μεγάλη πρόσκληση. Να του πείσουμε για το αντίθετο. Ωστόσο, οι κρατικοί φορεί, οι Δήμοι, η, περι... η Περιφέρεια, εμπροκειμένου ο Δήμο παραθώνα που είναι εδώ σήμερα, πρέπει να σηκώσουν το βάρο τη ευθύνη του για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μα και στην περιφερειακή Ε, συγκεκριμένα. Η Περιφέρεια Αττικής το έχει πράξει ήδη όπως καταλαβαίνετε και θα συνεχίσει να το πράττει. Ήρθε η ώρα και του Δήμου Μαραθώνα να στηρίξει τον περιφερειακό σχεδιασμό, όπω ακούσαμε. Σήμερα ευκαιρία που έχουμε και τον Δήμαρχο μαζί μα, που στι τελευταίε συναντήσει, όπω το περιφερειακό μα, για κάποιου λόγου προσωπικού φαντάζομαι δεν τον είδαμε, να ακούσει κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι από τον Ιούνιο του 2015 που ο Δήμο Μαραθώνα μα υπέβαλε τοπικό σχέδιο διαχείριση, κάπου έχει ξεχαστεί κάπου έχει ξεχαστεί και θα μιλήσω με στοιχεία όπως το πράττουμε και συνηθίζουμε άλλωστε συνεχώ στην περιφέρεια. Το 2015 ο Δήμο Μαραθώνα, κυρία Πρόεδρε, έστειλε στο χώρο υγειονομική ταφής της φυλής της Δυτική Αττικής ανεπεξέργαστα ροού σκουπίδια 22.000 τόνους απορριμμάτων το 2015. Το 2016, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να θεωρούμε ότι δεν μα ελέγχει κανένα, ότι έχουν μια συνεργατική σχέση ω τοπική, φορή τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά το 2016, ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, απλά να πω αυτό που πρέπει να πω. Ολοκληρώνω. Έστειλε πάλι 22.000 τόνου απορρίμματα στο χώρο υγειονομική ταφή φυλή. Το 2017 να σα απαντήσω πόσα έστειλε. Θα το μαντέψετε. Η απορία μου είναι πει, Τα κλαδέματα, για παράδειγμα, Χριστιανέ μου, τι τα κάνετε τα κλαδέματά σα. Ένα Δήμο παραθαλάσσιο, με δασικό χαρακτήρα, με αγροτικό χαρακτήρα, τι κάνουν τα σκουπίδια. Υποβάλα μια πρόταση στο ΜΕΠΕΡΑ και ολοκληρώνω και την υποβάλα την πρώτη τελευταία μέρα της εκνοής του προγράμματος για ένα πρόγραμμα που αξίζει να το στείλω και δεν συνάδει με το σχεδιασμό, τον περιφερειακό σχεδιασμό της χώρας μας. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα. Θέλω να πω μόνο ότι η λύση της φυλής δεν είναι λύση για κανέναν και δεν συνιστά ένα περιβαλλοντικά, οικονομικά και οικονομικά και περιβαλλοντικά δίκαιο σχέδιο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ό,τι χρειαστείτε επιπλέον στοιχείο είναι στη διάθεσή σα Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ Πρέπει να κλείσει αυτή η υπόθεση κάπου. Αλλά τώρα πρέπει να προχωρούμε. Ε, κυρία Σακοράφα. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι τώρα ήμουν πάρα πολύ ήρεμη και άκουγα ολου του συναδέλφου. Θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της περιφέρειας. Θα πήγαινε να μείνει στη φυλή ή σε μια περιοχή δίπλα στη φυλή. Ή ακόμη και εκεί που συζητάμε για τα σκουπίδια στο Καματερό, αν θα μπορούσε να είναι εκεί πέρα. Αν θα πάει να μείνει εκεί. Για όνομα του Θεού. Ο τρόπος που μιλήσατε είναι απαράδεκτος. Και ελπίζω ο κύριος Δήμαρχος ποτέ να μην συμφωνήσει για αυτό, που γίνεται, αυτό το έγκλημα που γίνεται εκεί. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ στα τεχνικά σημεία, κυρία Πρόεδρε, γιατί έχουμε όλοι μα άπειρα χαρτιά που έχουμε διαβάσει, νομίζω και σε εσά έχουν έρθει κτλ. Εγώ θα συνοψίσω επιτρέποντά μου στο θέατρο του παραλόγου που ζούμε πραγματικά αυτή τη στιγμή και επιτρέψτε με αυτή την έκφραση, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη μπίζνα που λέγεται σκουπίδια στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και παντού. Προσέξτε, οι πολίτε απευθύνονται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή τι κάνει, κάνει τη δουλειά που πρέπει. Δηλαδή τι κάνει, στέλνει αυτοψία και παρακολουθεί από κοντά τα συμβαίνοντα. Διαπιστώνει παρατυπίες. Και αυτές τις παρατυπίες τις κάνει συστάσεις προς, το, προς τις αρμόδιες αρχές. Οι αρμόδιες αρχές ανταποκρίνονται σε αυτές τις συστάσεις. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Τι λένε. Τις υλοποιούν, λέει, τις, παραβιάσει παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων, τις, υλοποιούν με χαράξη απλών δρόμων. Και τίποτα άλλο. Και αυτό το θεωρούν μετατροπή των, των, των όρων. Αν είναι δυνατόν. Εμπέζουν δηλαδή και την Επιτροπή μα και του πολίτε, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα και είναι υποχρεωμένοι να ξαναρχίσουν τη διαδικασία από την αρχή, να είναι χρονοβόρο, όπω είπε προηγουμένω και ο κύριο συνάδελφο εδώ, μέχρι να, να, να μπει το ζήτημα για συζήτηση στην Επιτροπή μα κτλ. Το χειρότερο όμω είναι ότι αμφισβητούν αυτό που οι άνθρωποι ζουν τόσα χρόνια εκεί, που έχει να κάνει με ρέματα, κυρία Πρόεδρε. 200 χρόνια ρέματα υπάρχουν εκεί πέρα, τα οποία οι κύριοι το αμφισβητούν. Και πήγανε και στα δικαστήρια οι πολίτε. Και αποκρύπτει με το έγγραφο που στέλνει η περιφέρεια εδώ, το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν έκρινε την ουσία, έκρινε τη διαδικασία, δεν έκρινε δηλαδή αν υπάρχουν ρέματα, έκρινε τη διαδικασία. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα, ο Δημοσφυλής κυρία Πρόεδρε, τεράστιο ζήτημα. Ο μεγαλύτερος σκουπιδότοπος στην Ελλάδα με ζωή 53 ολόκληρα χρόνια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εκεί. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως να πάει να μείνει ο κύριος εκπρόσωπος δίπλα. Ο Δήμος αναθέτει μελέτες, κυρία Πρόεδρε, και εδώ θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω τα χαρτιά και θα σας τα καταθέσω κιόλας. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε μελέτες για αναλυτική καταγραφή ποιοτική και ποσοτικής σύστασης αποβλήτων και για καταγραφή ρηπαντικών στο χιτά φυλής. Μια μελέτη η οποία δεν έφτασε ποτέ στα χέρια κανενός. Πληρώθηκε από τους πολίτες, από το Δημοτικό... Την έχετε? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει εκεί μέσα τι λέει. Είναι μια βόμβα που έχει σκάσει, δεν περιμένει να σκάσει. Ήδη έχει σκάσει, προσέξτε. Βαρέα μέταλλα, ε, υδρογονάνθρακε, αρωματικοί φενόλε, μεθάνιο, αμμόνιο, ραδιενεργά στοιχεία, ράδιο 24, ράδιο, τρίτη, θόριο, μόλιδο, τα πάντα. Και εκεί ζουν άνθρωποι. Και τολμάνε και λένε αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Λοιπόν, τι έκρυψε τις μελέτες. Και ξέρετε γιατί τις έκρυψε. τι έκρυψε γιατί πολύ απλά από τα 43 ευρώ τον τόνο που παίρνει για τα σκουπίδια, τα μισά είναι αντισταθμιστικά τέλη. Δηλαδή τα παίρνει ο ίδιος ο Δήμος. Τελειώνω κυρία Πρόεδρο. Το τρίτο παράδειγμα, και θα τελειώσω με αυτό, δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γι' αυτό και ζητάω την κατανόησή σα. Το επίσημο ελληνικό κράτο υπογράφει δεσμεύσει για μείωση μεικτών απορριμμάτων. Σύμφωνα με τι οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή όλο το ΕΣΠΑ κατευθύνεται 95% για διατήρηση των χιτά και το 5% μόνο στη διαλογή και στην ανακύκλωση, κυρία Πρόεδρε. Και έχω και αυτά τα στοιχεία να στα δώσω. Προσέξτε, η περιφέρεια στην περίπτωση του γραμματικού λέει ότι θέλει να κατασκευάσει χιτή και στην απάντηση που έστειλε στην Επιτροπή Δικαιολογή για ποιο λόγο θέλει να κάνει χιτά. Μόνο γι' αυτό το λόγο το Ταμείο Συνοχή καλά έκανε πιστεύω, γιατί αυτό κατάλαβα, αν κατάλαβα καλά, απέσυρε την υποστήριξή του. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να μείνει η ανηφορά ανοιχτή και για το γραμματικό και για τη φυλή. Θα πρέπει να ζητήσετε κατά την άποψή μου, κυρία Πρόεδρε, μετεπιτάσεως και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, μου είπατε ότι την έχετε την, την, την, Τη μελέτη την έχετε, τη μελέτη του Δήμου. Εάν δεν την έχετε, θα πρέπει να τη ζητήσετε οπωσδήποτε. Αν θέλουμε πραγματικά να υπερασπιστούμε εδώ μέσα ότι είμαστε μια επιτροπή η οποία υπερασπίζεται του πολίτε που καταφέρνουν σε αυτήν. Θέλω να ζητήσετε τον ρυθμό συμμόρφωση τη Ελλάδα στι δεσμεύσει που έχει αναλάβει στη διαχείριση των απορριμμάτων και πλήρω αιτιολογημένη απάντηση για την προκλητική κατανομή του ΕΣΠΑ. Και τελειώνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Θα σα παρακαλέσω ότι για, με το, για το ότι μόλι πριν, πριν από δύο μήνες η θαλάσσια περιοχή όπου καταλήγουν αυτά τα ρέματα φαντάσματα κηρύχθηκε Natura 2000 να επανέλθετε παρότι έχετε πάει στην περιοχή, να επανέλθετε ζητώ να μάθετε σε ποια ακριβώ σημεία συμμορφώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει των οδηγιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχει γίνει μελέτη για τι επιπτώσει στην περιοχή Natura. Επισημαίνω ότι το έργο προχωράει, τελειώνει και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί και με άμεσε και επιτακτικέ τι προτάσει μα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε το έργο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Now I see that there are now the mayor of Marathon and others wanting to take the floor. Now this... Και ο δήμαρχος του Μαραθώνος αλλά και άλλοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Θα συνεχίσω όμως με τους συναδέλφους μου πρώτα, ο κύριος Μαριάς. Ε, εγώ θα μείνω μόνο σε αυτή την αναφορά, γιατί η αναφορά για τη φυλή είναι μετά. Οπότε θα το συζητήσουμε μετά φαντάζομαι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις των πολιτών για το τι συμβαίνει στην περιοχή και για την μόλυνση η οποία υπάρχει στην περιοχή και για τα προβλήματα δημόσια υγείας που υπάρχουν ήταν τεράστιες και υπήρξε σειρά διαμαρτυριών. Πάρα πολλοί από τους πολίτες ε, απευθύνθηκαν ε, σε μένα ότι κάτι πρέπει να γίνει για το ζήτημα αυτό. Είχα την ε, χαρά να συναντήσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος τον Ιανουάριο ζήτησε να μπορέσουμε να επισπεύσουμε την συζήτηση αυτής της αναφοράς. Διότι αν την αφήναμε στις διαδικασίες γνωστές θα πήγαινε πάρα πολύ πίσω. Επομένως, με πρόταση δικιά μας, την οποία απευθύναμε στους συντονιστές, ε, έγινε εφικτή η σημερινή συζήτηση. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που αποδέχτηκαν αυτή την πρόταση, διότι από το ίδιο το βίντεο, κυρία Πρόεδρε, είδατε το τι περιβαλλοντική καταστροφή συμβαίνει. Και ρώτησα πριν λίγο για να επιβεβαιωθώ ε, σε σχέση με τον αναφέροντα, ο οποίος έφερε αυτό το βίντεο πότε γυρίστηκε και είναι σκηνές πράγματα που βλέπουμε από το 2017. Δηλαδή δεν είναι προ Χριστού, είναι τώρα. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει τώρα. Επομένως είναι σημαντικό το ότι δρούμε άμεσα για να συζητήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεύτερο επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, η ίδια, οι εκπρόσωποι, ο ίδιος ο εκπρόσωπος της περιφέρειας άφησε να εννοηθεί ότι αν υπάρξουν στο μέλλον περιβαλλοντικά προβλήματα θα το ξαναεξετάσουν. Ούτε οι ίδιοι δεν είναι σίγουροι για αυτό το οποίο γίνεται. Αναφέρθηκε και αναλύθηκε από τον Δήμαρχο αλλά και τους αναφέροντες όλο το πλαίσιο των παρανομιών σε σχέση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία. Και η νομοθεσία έχει αξία γιατί προστατεύει τη δημόσια υγεία και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν είναι γενικό και αορίστος ένας νομικισμός εδώ πέρα. Είναι να προστατεύσουμε την υγεία των κατοίκων. Να μην φτάσουμε σε καταστάσεις όπως στην φυλή, όπου εκεί έχουμε τεράστιο αριθμό καρκίνου. Οι κάτοικοι εκεί δεν μπορούν να σταθούν. Έχουν πληγεί. Και αυτό είναι το επόμενο θέμα στην επόμενη αναφορά. Επιπλέον αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ρέματα. Είδατε τι συνέβη με τα ρέματα τα οποία είχαν προβλήματα στην άλλη μεριά, στη Δυτική Αττική. Και είχαμε πρόσφατα 23 νεκρούς στην περιοχή της Μάνδρας. Η ίδια περιφέρεια χειρίζεται τα θέματα αυτά. Πρέπει να βάλει λίγο μυαλό γιατί θα έχουμε προβλήματα και στην περιοχή του γραμματικού. Επιπλέον, το έργο αυτό πρακτικά τι θα κάνει. Θα ανακουφίσει κατά 10 ημέρες τη λειτουργία της φυλής. Δεν πρόκειται να λύσει το θέμα. Αντίστοιχα όμως, ο Δήμος σας είπε ότι έχει το δικό του πρόγραμμα που είναι πολύ πιο φτηνό στη διαχείρισή του για να δει τα του του και να διαχειριστεί τα ε, απορρίμματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Το ότι σταματάει το Ταμείο Συνοχής να δίνει τα χρήματα και απεντάσει το έργο αποδεικνύεται ότι είναι καραμπινάτη η παρανομία. Επομένως πρακτικά τι κάνουμε εδώ και τώρα γιατί αυτό έχει σημασία. Η περιφέρεια σκοπεύει να συνεχίσει την ιστορία αυτή. Σκοπεύει ουσιαστικά να περάσει σε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα. Και όταν μιλάμε για μαραθώνα, γιατί ίσως πολλοί συνάδελφοι να μην, καταλάβουν να μην το ξέρουν, Λοιπόν, μιλούμε για την περιοχή του αρχαίου Μαραθώνα, μια ιστορική περιοχή όπου φυσικά είναι πλέον γνωστή σε όλο τον κόσμο λόγω του μαραθωνίου δρόμου που γίνεται. Είναι περιοχή που στηρίζει, αν θέλετε, πολιτισμικά την Ελλάδα. Είναι περιοχή που έχει σχέση με τον τουρισμό. Και από εκεί και πέρα είναι γενικώ μια περιοχή που οι κάτοικοι ανεξαρτήτως αν ζουν σε αυτή ή σε άλλη περιοχή πρέπει να προστατευτούν. Πρόταση, κυρία Πρόεδρε. Πρώτον, να παραμείνει ανοιχτή. Δεύτερον, να υπάρξει μία επιστολή προς την περιφέρεια Αττικής και προς, την, ε, προς το αρμόδιο Υπουργείο που να λέει το εξής να μην λειτουργήσει το έργο αυτό καθόλου ούτε έστω και δήθεν δοκιμαστικά που θέλει να το κάνει η περιφέρεια. Και με αυτόν τον τρόπο, γυρνώντας αυτά που είπα στην προηγούμενη ομιλία μου και παρέμβαση, θα είναι καθοριστική η παρέμβαση μας. Γιατί αν γενικώ πούμε ένα ευχολόγιο, το έργο θα γίνει, η ζημιά θα γίνει και θα έρθουμε μετά πάλι από δύο χρόνια και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Άρα λοιπόν να σταλεί η επιστολή στην περιφέρεια και στο Υπουργείο ζητώντας αυτό που ζητήσαμε στην περίπτωση της Ιταλίας. Την άμεση διακοπή ή ασδήποτε λειτουργία του έργου εδώ και τώρα. Αυτό είναι το αίτημα το σωστό και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και να ζητήσουμε και από την Κομισιόν να ελέγξει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Now... Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Πρέπει να σας θυμίσω ότι τελειώνει ο χρόνος μας. Ε, ε έχουμε πολύ καθυστερήσει. Προσπαθήστε να είστε σύντομο, γιατί περιμένουν δύο ακόμη αναφέροντες και δεν θα έχουμε διερμηνία μετά τις 6 Λοιπόν, κυρία Κούνεβα. Ναι, και εγώ προτείνω να μείνει η αναφορά ανοιχτή, να ζητήσουμε από Περιφέρεια Υπουργείο και Κομισιόν διευκρινήσεις και άλλα στοιχεία και να αποφασίζουμε τότε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνεβα, πολύ σύντομη. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομος. Υπερασπίζω το υπόμνημα που κατέθεσε ο κύριος Παπαδηγενόπουλος, ότι έτσι έχουν τα πράγματα, όπως επίσης και τις εικόνες που μας έδωσε ο κύριος Γκίκας όσο αφορά το πρόβλημα. Προσθέτω, όσο αφορά την τελική μας πρόταση, αν για τα προηγούμενα υπερασπίστηκα και εγώ την άποψη να είναι ανοιχτή πρόταση για τούτο εδώ το θέμα και για το επόμενο επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω συγκριτικό βαθμό και να σας εξήγησω γιατί, αν υπάρχει τέτοιος. Στην περίπτωση του γραμματικού η, πρόταση, η, η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή και να ζητηθεί αυτό που είπε ο κύριος Μαριάς, να σταματήσει κάθε έργο και να ζητηθεί από την περιφέρεια, θα έλεγα και από τις αρμόδιες και από την Υπουργεία, θα έλεγα με αυστηρή τέτοιο, αν βγάλαν κάποια συμπεράσματα από την πρόσφατη τραγωδία που είχαμε στην Μάντρα, που ήταν μια επιπόλαιη αντιμετώπιση του θέματος ρεμάτων στην Ελλάδα, στην Αττική και στην προκειμένη περίπτωση. Και επειδή εκεί θα επικεντρωθώ, είναι κακή χωροθέτηση. Από την αρχή. Έχω άμεση εμπειρία. Όχι μόνο γιατί επισκέφθηκα σαν Επιτροπή Αναφορών, αλλά κατηδία είμαι και μηχανικός, σε συνθήκες οριακές, καταιγίδα παραμονή Χριστουγέννων και αυτά τα φαινόμενα που μας έδωσε σε slide ο κύριος Γκίκατς τα είδε μπροστά τα μάτια. Είναι ρέμα, με συμπληρωματικό ρέμα. Αυτό δεν διορθώνεται. Γιατί και τότε που πήγα εγώ υπήρχαν κάτι μικρά, ε, μικρές οχυρωματικές ας το πούμε συνθήκες για να σταματήσουν όλα αυτά τα επιφανειακά νερά που πέφτουν και μολύνουν και θα μολύνουν τον ευωικό. Αυτό είναι αναντήρητο. Η, η απάντηση του ΙΓΜΕ απαντάει όσο αφορά τη διάβρωση των νερών. Κατά τα άλλα λέει είναι ρέμα. Το ίδιο και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Επομένως, για να μην επαναλαμβάνω όλα τα υπόλοιπα, διορθωτικά όσο αφορά την εφαρμογή περιβαλλοντικής ε, νομοθεσίας που έγιναν και δεν έγιναν, δεν θεραπεύουν το πρόβλημα. Και δεύτερο, μια ποσοτική, ποιοτική ανάλυση που μας έκανε ο ο κύριος εκπρόσωπος της περιφέρειας και μια αντιπαραβολή με τη φυλή πάλι δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο το πρόβλημα διότι είναι εγγενές, είναι αρχικό. Κακή χωροθέτηση. Αυτό ζητάω και γι' αυτό το λόγο είπα και υπερθετικό βαθμό. Ευχαριστώ. Τελείωσα. Εγώ ευχαριστώ. Listen, I see that... Η πρόεδρος. Η πρόεδρος. Βλέπω ότι ορισμένοι μου ζητείτε το λόγο. Δυστυχώς και για σας κύριε Δήμαρχε είναι αδύνατον. Έχουμε ακόμα δύο αναφορές και πρέπει να προλάβουμε. Έχουμε σημειώσει όλα όσα είπατε. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβετε. Ούτε και οι συνάδελφοί μου δεν χρειάζονται να επαναλάβουν τίποτε άλλο. Παρακαλώ, Πέτερ, κάντε μια καλή πρόταση, νέα πρόταση. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με τον κύριο Μαριά. Και νομίζω κάποια στιγμή είπε κάποιος κάτι σωστό. Ότι κατανοεί τις αντιδράσεις των πολιτών. Χρειάζεται πράγματι διαφάνεια, ασφάλεια σχεδιασμού. Το είπε και ο κ. Μαρία. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και παρακαλώ να το σημειώσετε και στο πρακτικό ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του σήμερα. And that doesn't happen often. Κάτι, που δεν συμβαίνει. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, λέει ο πρόεδρος. Μου φαίνεται είναι η πρώτη φορά. Σολεδάδ, παρακαλώ. Θέλετε κι εσείς να ενταχθείτε στην λέσχη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να πω σε σχέση με αυτή την αναφορά, με ενδιαφέρει και αυτή και η επόμενη. Βεβαίω θα πρέπει να μείνει ανοιχτή μετά, μετά από όσα ακούσαμε. Όμω ε, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί όλοι οι βουλευτέ ε, έχουμε διάφορε και πολλαπλέ δραστηριότητε και θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να κλείσει. Έχω πρέπει να είμαι στι 6 αλλού αλλά θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ζητήσω ένα διαδικαστικό και θα είμαι πολύ σύντομη. Σε σχέση με το αίτημα που έκανα σήμερα, θα σας πω ότι στην ατζέντα του Απριλίου δεν, είναι, δεν θα είναι σταθερή. Προτείναμε για το Μάρτιο, αλλά επειδή δεν ψηφίστηκε, τότε ολόκληρη η ατζέντα μπορεί να είναι έγκυρη, αλλά το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να ε, ξαναψηφιστεί στην επόμενη ατζέντα των ε, συντονιστών. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για μια αναφορά. Και θα ήθελα να μην συζητούμε τέτοιο είδου πράγματα και δεν μην κάνουμε τέτοιο είδου δηλώσει. Εδώ συζητάμε τα θέματα των πολίτων. Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι εδώ οι πολίτε, αλλά είναι σημαντικό και για του πολίτε. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ε, πλειοψηφία σαφή σε σχέση με αυτή την αναφορά και προσπαθούν ε, να την κλείσουν ώστε τελικά να γίνει αυτό ενάντια στην θέληση τη πλειοψηφία. Δεν θα μιλήσω για το περιεχόμενο λοιπόν. Θεωρώ ότι στην, Απρίλη, στην ε, ατζέντα του Απριλίου δεν έχει ψηφιστεί το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ψηφίστηκε λοιπόν σε καμία, σε καμία ε, φάση. Και δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό. Θα ήθελα λοιπόν η διαδικασία να, που ακολουθείτε να είναι σαφής. Μάλιστα, σημειώνω την άποψή σας, λέει η Πρόεδρος, και τώρα προχωρούμε με αυτήν εδώ την αναφορά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να συνοψίσουμε. Βεβαίω πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και εμεί εξ ονόματο τη Επιτροπή μα θα στείλουμε επιστολέ στην Περιφερειακή Αρχή, στο Αρμόδιο Υπουργείο και θα εκφράσουμε τι ανησυχίε μα όλε αυτέ για την έλλειψη συμμόρφωση προ το Natura 2000 ε, και για την ανάγκη εκπόνησης ε, χωριστής περιβαλλοντικής μελέτης γιατί έχω την αίσθηση αφού άκουσα και το Δήμαρχο ότι οι ανησυχίες των πολιτών δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη <clears throat> Επίσης, θα ενημερώσουμε εδώ τις Επιτροπές Περιβάλλοντος την Επιτροπή Περιβάλλοντος και συμβουλεύουμε την Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει σε σχέση με την πυροή και των πολιτών. Χρειάζεται δημόσια διαβούλευση και το υπογραμμίζουμε αυτό πως είναι καθήκον σύμφωνα με την σύμβαση του Όρχους να γίνεται διαβούλευση με τους πολίτες. Προς τους αναφέροντες θα ήθελα να πω ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς ήρθατε εδώ, εμείς καταγράψαμε τις απόψεις και τα στοιχεία που μας δώσατε θα πρέπει να στραφείτε στον Έλληνα διαμεσολαβητή αυτή τη στιγμή, ακόμα και στα δικαστήρια σε μια περαιτέρω φάση. Αλλά αυτό είναι ο δρόμο να προχωρήσετε, αφού εμείς παίξαμε το δικό μας ρόλο σε αυτή την Επιτροπή. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέω το εξή. θέλω να δω ενημερωμένε πληροφορίες όπου θα ήθελα να μας σχολιάσετε τα τελευταία έγγραφα και ιδιαίτερα την μελέτη της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την άποψή σας ε, περί αυτής. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας και επίσης θα ήθελα να δούμε ακόμα μια φορά την γύρω περιοχή που είναι Natura περιοχή Natura 2000 και κατά πόσο αυτό ως όχητα εντάσσεται σε αυτήν την προοπτική. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλετε κύριε Μαριά να συμπληρώσετε κάτι. Με όλα όσα είπατε, απλά να προσθέσω ένα σημείο και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει στην επιστολή μας στην περιφέρεια και στο Υπουργείο να επισημαίνουμε ότι πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του έργου αυτού άμεσα και να μην γίνουν άλλες ενέργειες γύρω από αυτό το έργο. Κάτι τέτοιο το είπαμε και το ζητήσαμε και στην Ιταλία και νομίζω ότι είχε αποτέλεσμα, διότι καθώς παραμένει ανοιχτή αυτή η υπόθεση θα έχει αξία υπό τον όρο ότι δεν θα προχωρήσουν. Γιατί αν προχωρήσουν εμείς θα συζητούμε και σε δύο χρόνια θα είναι χειρότερη η περιβαλλοντική καταστροφή. Το δικαιούμαστε, μπορούμε να γράψουμε αυτό και θα ήθελα να το δούμε ως Επιτροπή. Το κάναμε στην περίπτωση της Ιταλίας. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να το επιχειρήσουμε και στην περίπτωση αυτή. Mr. Marias. Ε, ναι, κύριε Μαριά, δεν λειτουργεί από ό,τι κατάλαβα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το σημείο κίνησης. Σε επόμενε μέρε, πολύ ναι. σύντομα κυρία Πρόεδρε, θα ναι. γίνει αυτό. Και οπότε, εάν χρησιμοποιηθεί ω χιτά, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα ναι. θα υπάρχει. Ναι, ναι. Τώρα πρέπει να προχωρούμε. Listen, we need now to close. Λοιπόν, πρέπει τώρα να κλείσουμε αυτό το θέμα. Θα προχωρήσουμε, όπως είπαμε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθατε από τόσο μακριά και που μας ενημερώσατε με πολύ περιστατωμένο τρόπο για το ποια είναι η κατάσταση. Σας εύχομαι Καλό, καλή επιστροφή στην υπέροχη αυτή γωνιά της Ευρώπης, το Μαραθώνα, που ελπίζουμε να παραμείνει πανέμορφη αυτή η γωνιά της Ευρώπης και να σκέφτεσαι τώρα όταν επιστρέφετε στην Ελλάδα να μην επαναλάβετε αυτά που έκανε ο Φιδιπίδης που επέστρεψε μετά από τη μακρά του πορεία και είπε «Ναι, νικήκαμε. Ναι». Αλλά ναι, να, το πείτε, αλλά μην πέσετε νεκροί. Να το πείτε τον νικήκαμε, αλλά μην πέσετε νεκροί σαν εκείνον. <laughs> Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Have a safe trip back. Καλή επάνωδο. Ελλάδα και θα, θα σας μιλήσω με αργότερα. Petition... Η 17-10 αναφορά και, 200, και μάλλον η 28-87 είναι για παρόμοιο θέμα. Δεν χρειάζεται νομίζω να επαναλάβουμε πολλά πράγματα. Θα ήθελα ο αναφερόμενος κύριος Γκίκας να είναι συντομότατος. Γνωρίζω ότι έχει και PowerPoint, αλλά προσπαθήστε να μας την δείσετε γρήγορα. Με τον τρόπο αυτό μηδενίζουμε αυτή την αναφορά όταν μιλάμε για την ε, χωματερή της φυλής. Οι κάτοικοι μου στείλαν έξι σελίδες, δεν θα διαβάσω έξι, μία και αυτή τη μία μισή από ό,τι βλέπω. Επιτροπή Αγώνα Φυλής για το άμεσο οριστικό και αμετάκλητο κλείσιμο της καρκινοχωματερής στα νολιώσια φυλή και όλων των εγκαταστάσεων που υπάρχουν μέσα και γύρω από αυτήν από το 1960. Είτε εφαρμοστεί είτε δεν εφαρμοστεί η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με την παρούσα ανοιχτή επιστολή σας ενημερώνουμε ότι μετά από την επίσκεψή σας στην καρκινοχωματερή στα Άνω Λιώσια Φυλή το Σεπτέμβριο του 2013 και το έγγραφο εργασίας σας το Μάρτιο του 2014 καθώς και την συζήτηση που διεξήχθη κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Αναφορών τη 16η Τετάρτου 2015 η κατάσταση στη Φιλή και στις γύρω περιοχές αντί να βελτιωθεί έχει χειροτερεύσει και έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Στο προαναφερόμενο έγγραφό σα αναφέρεται και απαιτείται τα εξή. Η τοποθεσία του χιτάχου ματερί στη φυλή πρέπει να υποβληθεί σε επαναξιολόγηση και ειδικέ μελέτε θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με το σκοπό να καθοριστεί η προέλευση τη μόλυνση και ο υψηλό βαθμό εμφάνιση ασθενειών στον τοπικό πληθυσμό. Οι μελέτε που έχουν διεξαχθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταδεικνύουν ότι τα υπόγεια ύδατα έχουν υποστεί βλάβη που δεν μπορεί να επανορθωθεί ή αποκα... από αποκατασταθεί. Ακόμα και αν ο χώρο υγειονομική ταφή έπαβε σήμερα να λειτουργεί. Θα χρειάζονταν περίπου 200 χρόνια για την ανάκαψη του περιβάλλοντο. Τα κρούσματα καρκίνου είναι εξαιρετικά συχνά στην περιοχή, ιδίω μεταξύ των νέων και, ε, και του προσωπικού που απασχολούνται στο χώρο υγειονομική ταφή λόγω του μολυσμένου αέρα. Το σύστημα διαχείριση αποβλήτων στη φυλή πρέπει να αντικασταθεί από συστήματα ανακύκλωση και διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή, ενώ θα πρέπει να λάβει χώρα περιβαλλοντική αποκατάσταση στην ακριβή τοποθεσία του χιτά. Ο εγκύτερο οικισμό του Χιτά βρίσκεται μόλι 500 μέτρα μακριά. Οι κάτοικοι τη περιοχή θέλουν να πάυσει η λειτουργία του χώρου υγειονομική ταφή, να καθιερωθεί ένα νέο σύστημα διαχείριση των αποβλήτων. Οι κάτοικοι τη φυλή λυπούνται από το γεγονό ότι ο χώρο του Χιτά χωματερή στη φυλή λαμβάνει τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μέχρι στιγμή δεν έχουν λάβει χώρα διαβουλεύσει με την τοπική κοινωνία. Και εδώ είναι ο κύριο Μαριά που λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση και να γίνει και η στάτη και το γραμματικό και η ΦΥΛΗ. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντο στη φυλή θα πρέπει ε, να αποσταλεί ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάου, ασθενειών και ανθρώπινη δυστυχία τουλάχιστον για τι επόμενε τρει γενιέ που θα ζουν στην περιοχή. Εκτό αν συμβεί κάτι ριζοσπαστικό για την αποκατάσταση τη περιοχή και τρέχω στην επιστολή, παραβλέπω μερικά, από τις 7 παραπάνω απαιτήσει σας για τη φυλή, καμία απολύτως δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα 21 Τρίτου 2018. Αντιθέτω, η Περιφέρεια Αττικής και ο Φορέας Διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων της Αττικής, ο ειδικό διαβαθμιτικός σύνδεσμος του νομού Αττικής, με επικεφαλή στην Περιφερειάρχη Αττικής και ταυτόχρονα πρόεδρο του ΕΣΔΕΝΑ, κυρία Ρένα Δούρου, την αντιπρόεδρο του ΕΣΔΕΝΑ, κυρία Αφροδίτη Πιζά, τον Δήμαρχο Φιλή, κύριο Χρήστο Παππού και τον πρώην Δήμαρχο Φιλή, κύριο Δημήτρη Μπουραήμι και τον πρώην Δήμαρχο Κερατέα, κύριο Σταύρου Γιατρού, μαζί με όλα τα 61 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ, έπρεψαν τα κάτωθη. Πρώτον, συνεχίζουν να χορηγούν στο Δήμο Φιλή αντισταθμιστικά χρήματα ύψου πάνω από 36 εκατομμύρια ευρώ. Β. Συνεχίζουν να γεμίζουν με σύμμυκτα σκουπίδια του υπάρχοντε λάκου Β3, Β6 στη Β φάση τη καρκινομαχατερή στα Ανολιώσια. φιλή έω και το έτο 2035. Επιδίωξαν και εξασφάλισαν την έκδοση τη αδεία λειτουργία του άχρηστου εργοστασίου μηχανική ανακύκλωση και κουμποστοποίηση. Επιδίωξαν και εξασφάλισαν την ανανέωση τη Εργολαβική Σύμβαση του ΕΣΝΑ με τον Βόμπολα για την του χρήση και λειτουργία του εργοστασίου καύσεω από τεφροτήρα των άκρου επικίνδυνων μολυσματικών και τοξικών νοσοκομιακών και ιατρικών αποβλήτων. Επιδίωξαν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, επιδίωξαν και εξασφάλισαν μέσω του ΙΠΕΚΑ την αύξηση τη ισχύω του εργοστασίου καύσεω. Και τελειώνω με την τελευταία παράγραφο. Από τα ανωτέρω καθίσταται πλέον σαφέστατο από οτιδήποτε άλλο ότι το ελληνικό κράτος μέσω της περιφέρειας Αττικής και του ειδικού διαφαμιντικού συνδέσμου του νομού Αττικής θέλει να δημιουργήσει στη φυλή το μεγαλύτερο στον κόσμο σύγχρονο ταχάο κακινοπαθών, δεδομένου ότι οι θάνατοι από καρκίνο στους κατοίκους της φυλής και των γύρω περιοχών έχουν ξεπεράσει το 90%. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μειώνουμε αυτό το, το θέμα του χιτά, όσο αφορά με το χιτά φυλής και του γραμματικού και θα παρακαλούσα να μείνουν ανοιχτά και ε, να γίνει και στάτη για σας αυτές οι αναφορές. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Now I'd like to listen to the Commission representative, Mr. Diaz de Castillo. And meanwhile, I would like to ask uh, Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Δεκπεστίγιο. Κύριε Χουντή, νομίζω θα μπορούσατε σύμφωνα με τον κανονισμό να έρθετε στο έδρανο να με αντικαταστήσετε για δύο-τρία λεπτά στο Προεδρείο. Γίνεται, γιατί είστε ο γυρεότερος, αρχαιότερος. Thank you, Chair. Um... Ο κύριο Δελκαστήγιο της Επιτροπής. Ε, μάλιστα, αυτό συνδέεται πολύ καλά με τα όσα είπα και νωρίτερα. Μελέτη για ματερέ ε, και την διαχείριση απορριμμάτων που παρουσιάστηκε νωρίτερα. Η Κομισιόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη ε, γενική κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων όχι μόνο στην περιοχή της Αττική, αλλά σε ολόκληρη την χώρα όπου δυστυχώ οι χωματερές είναι 80% των, απο, των ε, απορριμμάτων. Δουλεύουμε σκληρά για τεχνική αρρωγή, περιμένοντας να υπάρξει μια μετακίνηση προς την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα, όπως έχει συμβεί σε άλλα βορειότερα κράτη-μέλη. Και όσο πιο σύντομα γίνει αυτό, τόσο καλύτερα. Έχουμε εκτιμήσει το περιφερειακό σχέδιο διαχείριση απορριμμάτων για την Αντική που υιοθετήθηκε το 2016, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων επιπλέον ε, καταστάσεις επεξεργασίας βλήτων και επιπλέον χωματερές. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτές οι νέες δυνατότητες θα έρθουν να σώσουν και να ελαφρύνουν την κατάσταση στην περιοχή Φιλή. Θα πρέπει να πω ότι οι ελληνικές ε, αρμόδιες αρχές που δημοκρατικά έχουν ε, κληγεί να άμεσα υπεύθυνε για να απαντήσουν καταλήλως ώστε να αποφύγουν καταστάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την... Ε, το περιβάλλον και έχουν υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας. Αν αυτό το αποφύγουν, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δικαστική επανόρθωση, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο εκεί ε, που τα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί. Η Επιτροπή λοιπόν θα συνεχίσει να και είναι δεσμευμένη στην παροχή της τεχνικής αρρωγής στην οποία αναφέρθηκα και νωρίτερα. Θα συνεχίσει λοιπόν να βοηθάει και να ε, διευκολύνει την περιφέρεια της Αττικής να χειριστεί τα 161 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν για την διαχείριση των οικιακών ε, λιμάτων στην περιοχή, των αστικών λιμάτων στην περιοχή. Ευχαριστώ. Τους Κομισιόν και τώρα σύμφωνα με τα, τους κανόνες το λόγο θα πάρει η κυρία Μπιζά η οποία είναι εδώ και είναι αντιπρόεδρος του ΕΣΤΝΑ και για δύο λεπτά του ενιαίου διαχειριστικού. Ναι. Κύριε ε, Πρόεδρε, δεν, δεν είναι δύο λεπτά, δεν είναι αρκετά. Νομίζω πέντε λεπτά όπως δόθηκαν σε όλους για να πω κάποια στοιχειώδη ε, πράγματα από αυτά που έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε σας παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν... Καταστάτης Πρόεδρο, όπως είδατε, οφείλω να πω τους κανόνες θα υπάρξει, αν όχι μην έχετε καμία αμφιβολία. Απλώς να είμαστε όλοι μέσα στο χρονικό που έχει η Επιτροπή, ναι. έχουμε ναι. και τους ναι. διαρμηνείς. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η, η οχητά της φυλής πραγματικά ε, λόγω της μακρόχρονης λειτουργίας του έχει επιφέρει ανυπολόγιστες βλάβες στην περιοχή και τις ε, άλλες τις γύρω περιοχές. Ε, απάντηση λοιπόν σε αυτή την κατάσταση είναι ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός τον οποίο έχει σχεδιάσει και ήδη υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί και με την έγκρισή του ε, εκπλήρωσε τη σχετική αιρεσιμότητα όπως αναγνωρίστηκε από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Σήμερα, σε συνεργασία με τους Δήμους, προχωρούμε στην αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων που βασίζεται στις αρχές της εγκύτητας και της μικρής κλίμακας και στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Οι Δήμοι πλέον, σύμφωνα με τους στόχους του νέου περιφερειακού σχεδιασμού, καλούνται να διαχειριστούν μέσω της διαλογής στην πηγή το 52,66% των αστικών στερεών αποβλήτων. Στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό προβλέπονται έξι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων που θα διαχειρίζονται το 25,56% των απορριμμάτων και τρει χιτή, του οποίου θα καταλήγει για διάθεση το υπόλοιπο των απορριμμάτων. Όσον αφορά τώρα το χιτά φυλή, στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό προβλέπεται αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση των δυνατοτήτων στοχητά φυλής ή και αξιοποίηση θέσεων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητά τους ως χιτή με τον νόμο 364 του 2003 και στη συνέχεια αναφέρεται οριστικό κλείσιμο του χώρου υγειονομικής ταφής φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων. Η Επιτροπή σας μετά την επίσκεψή της στο Χιτάφλι το 2013 είχε ζητήσει την άμεση διεξαγωγή τοξικολογικών και επιδημιολογικών μελετών από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς στον πληθυσμό του Δήμου Φιλής. Ήδη σήμερα μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα και εκτίμηση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή της. Σκοπός της είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των εργαζόμενων στην ΟΕΔΑ και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η επιστημονική έρευνα που θα διεξαχθεί θα εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών τόσο στους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις όσο και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Στην ομάδα του έργου συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, η Εθνική, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας. Ε, ήδη η ομάδα αυτή έχει παραδώσει την πρώτη τριμηνιαία απολογιστική έκθεση παρακολούθηση και αξιολόγηση τη πορεία υλοποίηση των εργασιών. Εδώ θέλω να πω ότι ακούστηκε σήμερα για μία μελέτη που υπάρχει και εμφανίζει αυξημένου ρήπου. Θέλω να βεβαιώσω ότι ο ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια δεν γνωρίζαμε τίποτα για τη μελέτη αυτή. Όμω, όπω είπα και πριν, ε, σίγουρα η μακρόχρονη λειτουργία έχει επιβαρύνει ανυπολόγιστα το, το χώρο εκεί τι γύρω περιοχέ, Γι' αυτό ακριβώ και στο περιφερειακό σχεδιασμό προβλέπουμε κλείσιμο του χιτάφυλής. Τέλο θέλω να πω σε συντομία και τελειώνω κυρία Πρόεδρε ότι έχουμε ξεκινήσει επειδή ακριβώ υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και μέχρι το κλείσιμο τη φυλής που θα συνδυαστεί και με του νέου χώρου έχουμε ξεκινήσει διαδικασία για ανάπλαση 250 στρεμάτων του ολοκληρωμένου τμήματο τη Β' φάση, με φύτευση 2.500 δέντρων και 44.000 θάμνων. Έχουν ε, ληφθεί μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους με παρακολούθησή του από γιατρό εργασίας και με διενέργεια εξετάσεων. Thank ε, κυρία Πρόεδρε, δύο θέματα ακόμα. Γίνονται συστηματικά περιβαλλοντικοί έλεγχοι στον χώρο του Χιτά ε, για να, ακριβώς για να μπορέσει να μειωθεί και να αποτραπεί αυτό το θέμα των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γίνονται επίσης συστηματικά μετρήσεις και έλεγχη της σύνθεσης των αποβλήτων, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ εκεί. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα εγκατασταθούν τρεις φωτοβολταϊκοί σταθμοί, ε, ότι προσπαθούμε με την ε, υλοποίηση των δράσεων ανακύκλωσης, ανάκτησης και κομποστοποίησης να μειώσουμε και έχουμε μειώσει ως ένα βαθμό τα απορρίμματα που φέρνουν οι Δήμοι στην ΟΕΔΑ Προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση και δεσμευόμαστε να προσκομίσουμε στην Επιτροπή σας όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς μας. Thank you very much. Η Πρόεδρος, κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ. Κύριε Μαριά, προσπαθήστε να πείτε ακριβώς τι θέλετε να κάνουμε την ε, συγκεκριμένη ε, αναφορά. Ένα λεπτό μόνο, λέει ο κύριος ε, Μαριάς. Πρόκειται για ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα, αλλά όχι, δεν είναι σημερινό. Είναι χρόνια αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή της Αττικής και ιδιαίτερα στην χωματερή της Φυλής. Έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ε, προβλήματα, τεράστια προβλήματα υγείας, δηλητηρίαση επί της ουσίας του πληθυσμού, καρκινογενέσεις ε, και όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξει αποφασιστική παρέμβαση. Να υπενθυμίσω ότι πριν δυόμιση χρόνια συζητήσαμε αυτή την υπόθεση εδώ και από τότε είχαμε πει ότι πρέπει να γίνουν τοξικολογικές μελέτες και από ό,τι ακούω μετά από δυόμιση χρόνια μέχρι στιγμής κάποιο πρώτο αποτέλεσμα δεν έχουμε. Δεύτερον, η πίεση που ασκεί η Επιτροπή είναι προφανές ότι πιέζει την περιφέρεια να πάρει μερικά μέτρα, αλλά δυστυχώς τέτοια μέτρα δεν παίρνονται. Αναφέρομαι και εγώ στις καταγγελίες των κατοίκων και της Επιτροπής Αγώνα Φιλής και προτείνω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ότι πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ανοιχτή αυτή η υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Η ίδια η εκπρόσωπος ε, μας είπε πριν λίγο ότι θα μας ενημερώσει για νέα στοιχεία, άρα λοιπόν παραμένει ανοιχτή να ελέγξουμε κατά πόσο, κατά πόσο εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα της αναφοράς. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Kuneva, do you... Παρακαλώ. Κυρία Κούνεβα, συμφωνείτε να προχωρήσω στο συμπέρασμα γιατί έχουμε και την ισπανική αναφορά. Ε, νομίζω θα συμφωνήσετε. Να κάνουμε το εξής να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ε, καταγγελίες των αναφερομένων, να στείλουμε γράμμα στο Υπουργείο Υγείας για τις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες και να αναφέρουμε και την τοξικολογική μελέτη που έχει πολύ μεγάλη σημασία και επιστολή και στις περιφερειακές αρχές όπου θα ζητήσουμε γραπτή ενημέρωση για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής και για το πώς βλέπουν την όλη κατάσταση. Και νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε και ένα γράμμα για να είμαι πολύ ειλικρινής και να είναι πολύ ειλικρινές το γράμμα και στο Δήμαρχο της Φυλής. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Νομίζω ότι συμφωνείτε κυρία Κούνεβα, έτσι δεν είναι. Δεν σας γνωρίζω καλά άλλωστε. Πολύ καλά. Θαυμάσια λοιπόν τώρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με την επόμενη αναφορά. Και έχουμε τώρα μόνο 6 λεπτά, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε στην 232 και παρακαλούμε τον αναφερόμενο να μιλήσει για 2 λεπτά. 2 λεπτά. Νομίζω ότι μπορείτε να προλάβετε γιατί σε λίγα λεπτά διακόπτουν οι διερμηνείς. You need use the microphone. Παρακαλώ με μικρόφωνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν σας είναι άγνωστο και πρόκειται για τον λίγο σεβασμό ή τον ισχνό ή τον ανύπαρκτο σεβασμό της περιφέρειάς μας για το περιβάλλον. Ε, θέλουμε να σας υποβάλουμε μια υπόθεση ε, ακόμα για ακόμα ένα επεισόδιο μιας ε, ε, χωματερήσεις στο Αλικάντε αυτή τη φορά. Ε, έχουμε την τοποθεσία, μάλλον υπάρχει μια εγκατάσταση που δεν ε, έχει αδειοδοτηθεί μέσα σε χώρο προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, αναφερόμαστε στην ε, Κανιάδα που είναι ένα φυσικό ε, πάρκο, είναι ένας ε, δρυμός και είναι μοναδικός χώρος στον κόσμο. 92-43 είναι η ε, οδηγία και πρόκειται για έναν χώρο που θεωρείται κοινοτικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται λοιπόν για ένα οικότοπο μοναδικό, είναι ένα πολύ μικρό οικοσύστημα και είναι μοναδικό στην Ιβηρική Χερσόνησο. και προστατεύεται κανονικά από την οδηγία για τους ε, οικοτόπους. Μετά την τελευταία επιθεώρηση του 2014 είχαν ενημερωθεί τη δραστηριότητα είχαν, είχε σταματήσει. Ωστόσο, εμείς είδαμε ε, πρόσφατα ε, να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη κατάσταση και θέλουμε να τονίσουμε την ε, μόνιμη προσπάθεια της επιχείρησης που διαχειρίζεται αυτόν τον χώρο ε, για να αποκτήσει την άδεια. Έχουμε στραφεί στο ανώτατο δικαστήριο της Βαλένθια και στο ανώτατο ισπανικό δικαστήριο ώστε να, ε, κάνουν, ε, να, να πάψει η δραστηριότητα αυτής της επιχείρησης. Η δική μας λοιπόν διοίκηση ελέγχει κατά πόσο διατηρείται μετά το κλείσιμο του εργοστασίου η διατήρηση αυτής της δραστηριότητα. Έχετε παληθεύσει κατά πόσο έχει εφαρμοστεί αυτό το διάταγμα. Να θυμίσω την ευθύνη των αρχών να εγγυηθούν τη συντήρηση και την αποκατάσταση του χώρου και αυτή τη στιγμή δεν μας έχουν εξηγήσει καθόλου γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο χώρο χωρίς δραστηριότητα, πώς γίνεται να φτιάχτηκε και χωρίς άδεια, πώς γίνεται να φτιάχτε και σε έναν ειδικό χώρο ε, που είναι προστατευόμενος. Πρέπει λοιπόν να πάψει όλη αυτή η ιστορία που εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο το, το, πληθυσμό μας, την πανίδα και τη χλωρίδα και ελπίζουμε πως στο μέλλον θα έχουμε καλύτερη ισορροπία με το περιβάλλον μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή σας για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι στιγμή. Θέλουμε να οι αρχές να τιμωρήσουν οποιονδήποτε λειτουργεί ε, παρανόμως οι αρμόδιες αρχές να ελεγχθεί ότι όντως κάνουν έλεγχο για την δημόσια υγεία και να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία που ξεκίνησε από αυτήν την εταιρεία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ζητώ συγγνώμη που ήμουν τόσο γρήγορος. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη που σας βιάζουμε τόσο πολύ, όμως πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσει η έκβαση και αυτό είναι το βασικότερο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι και αυτός συντομότατος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. οι πληροφορίε που έχει στη διάθεσή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν είναι λειτουργική η χωματερή για την οποία μιλεί ο αναφερόμενο και η υπόθεση είναι ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστικών αρχών. Μη λειτουργική, επαναλαμβάνω, η χωματερή, η οποία ενδέχεται να ξανανοίξει εάν συντρέχουν οι συνθήκες όπως θα αποφασίσει το δικαστήριο, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε για την ώρα. Θεωρούμε ότι τα εθνικά δικαστικά όργανα παίζουν τον ουσιώδη ρόλο για την εξασφάλιση τη εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όπου υπάρχει η διαδικασία ενώπιον Εθνικού Δικαστηρίου έχει μέγιστη σημασία να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας με την αποφυγή επικάλυψης. Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι άλλη παρά μόνον όταν θα ολοκληρωθεί η, διαδικαστική, η δικαστική διαδικασία και θα υπάρξει μέσω της διαδικασίας αυτής ένδειξη ότι έχει παραβιαστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλά εγγεγραμμένα μέλη. Θέλω να μας πείτε μόνο τι θέλετε να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε με μια θετική νότα. Κυρία Μιράντα. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να στηρίξω αυτήν την αναφορά. Συγγνώμη, αλλά η διερμηνία εδώ πάβει γιατί σχολάμε. Γεια σας. Η Σεβαστία... Ε, Οι διερμηνείς έχουν ρητές οδηγίες από την διοίκησή τους να διακόψουν ακριβώς 18 και 30. Ζητούμε την κατανόησή σας. Χαίρετε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 και να ελέγξουμε την παραβίαση που έχει διαπιστωτεί το 14 ακόμα. Fine. Um, now let's see Mrs. Sakurafa. I suggest to remain open this. And Mr. Marcelest.